colleagues, Συνάδελφοι, αποφασίσαμε να περιμένουμε λίγο, μπας και έρθουν περισσότεροι συνάδελφοι να επιστρέψουν από το γεύμα τους, από ό,τι φαίνεται όχι. Θα ήθελα όμως να υποδεχτώ τον Επίτροπο Ντεγκούχτ, ο οποίος θα μας ενημερώσει για τις εξελίξεις στην ΑΚΤΑ, την συμφωνία για την καταπολέμηση της παραποίησης απομίμησης που έχουμε συζητήσει αρκετές φορές στο Κοινοβούλιο. Του δίνω αμέσως το λόγο και μετά θα περάσουμε σε ερώτα-απαντήσεις. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη. Σας ευχαριστώ που με προσκαλέσατε στην Κοινοβουλευτική σας Επιτροπή σήμερα. Σημείωσα το ενδιαφέρον της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών και άκουσα και τις ανησυχίες που εκφράστηκαν από αρκετά από τα μέλη αυτής της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής και γι' αυτό καλωσορίζω αυτή την ευκαιρία να έχουμε μια ανοιχτή, ειλικρινή συζήτηση μαζί σας σήμερα. Πάντα ήμουνα θερμός υπέρμαχος των πολιτικών ελευθεριών και του κράτους δικαίου και θα κατανοήσετε ότι δεν θα είμαι υπέρ μιας συμφωνίας αν υπήρχε κάποιος λόγος να υποπτεύεται κανείς ότι θα είχε αρνητικές επιπτώσεις στις πολιτικές ελευθερίες. Θα επανέλθω σε αυτό το σημείο ύστερότερα. Πρώτα, επιτρέψτε μου να πω ότι το πλαίσιο αυτών των διαπραγματεύσεων αυτό που διαπραγματευόμαστε με την ΑΚΤΑ είναι μια συμφωνία που θεωρούμε ότι είναι σημαντική να διασφαλίσει την ανταγωνιστικότητα της ΕΕ στις παγκόσμιες αγορές. Και για να παραμείνουμε μια ανταγωνιστική οικονομία θα πρέπει να βασιζόμαστε στην καινοτομία, την δημιουργικότητα και την αποκλειστικότητα. Και αυτό είναι ένα από τα κυριότερα προτερήματά μα εναντί των ανταγωνιστών μα στην διεθνή αγορά. Χρειαζόμαστε ένα μέσο, ένα εργαλείο, ώστε αυτό το ανταγωνιστικό προτέρημα πλεονέκτημα να διασφαλίζεται στις ε, εξαγωγικές αγορές παγκόσμια. Και αυτά είναι θέματα τα οποία απασχολούν ε, τους ε, πολίτες, θέματα θέσεων απασχόλησης για να είμαστε δημιουργικοί και ανταγωνιστικοί. Η πραγματικότητα είναι ότι οι πολίτες ΕΕ θα υποφεληθούν από την άκτα. Δεν είναι κάτι το, που έχει κάποια αρνητική επίπτωση όπως κάποιοι το παρουσίασαν. Θέλουμε να υπάρχει ένα διεθνές πρότυπο για τα πνευματικά δικαιώματα και τα, να συμμορφώνονται με αυτές τις διατάξεις με τέτοιο τρόπο όλο, ώστε να μπορούν αναδυόμενες οικονομίες να, να μελλοντικά από αυτό, ώστε να διασφαλίσουμε ότι θα προστατεύεται η καινοτομία επαρκώς σε εκείνες τις αγορές που έχουν ρόλο και είναι σημαντικές. Αυτό είναι τέλος τέλος ο ίστατος στόχος. Και είμαι βέβαιος ότι από αυτού όλοι συμφωνούμε. Όλοι θα έχετε δει το σχέδιο κειμένου της ΑΚΤΑ που δημοσιοποιήθηκε τον προηγούμενο Απρίλιο και ελπίζω ότι σας έδωσε την ευκαιρία να διασφαλίσετε, να επαληθεύσετε ότι οι κύριες αρχές που εμπνέουν την Επιτροπή σε αυτές τις διαπραγματεύσεις και που ήδη στην Ολομέλεια ανέφερα έχουν ακολουθηθεί αυστηρά. Λοιπόν, να αναφέρω. Πρώτον, ο στόχος της αυτά είναι να αντιμετωπίσει σε ευρεία κλίμακα τις παραβιάσεις και παραβάσεις των πνευματικών δικαιωμάτων. Δεν είναι έλεγχος όσον αφορά το περιεχόμενο στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές ή στα λάπτοπ των ταξιδιωτών. Δεν θα οδηγήσει, οδηγήσει σε προβλήματα ή ενόχληση, όχληση των ε, καταναλωτών. Σε περίπτωση που έχετε κάποιες αμφιβολίες, με χαρά να ακούσω τα επιχειρήματά σας και να δούμε πώς και με ποιο τρόπο η ε, διατύπωση θα είχε επιπτώσει στις πολιτικές ελευθερίες. Δεύτερον, η άκτα είναι μόνο για την επιβολή διατάξεων για τα πνευματικά δικαιώματα. Δεν θα έχει ε, κάποιες διατάξεις που να τροποποιεί τα πράγματα όσον αφορά τα πνευματικά δικαιώματα. Θα διασφαλίζει ρήτρε και διατάξει ώστε να επιβάλλονται αυτά τα δικαιώματα δικαστικά, διασυνοριακά και μέσω του διαδικτύου. Θα διασφαλίζει η άκτα ότι, για παράδειγμα, ένα καλλιτέχνη στο ε, βιομηχανικό σχέδιο ή στην μόδα θα μπορεί να διασφαλίζει την ε, δική του πνευματική ιδιοκτησία έναντι προϊόντων μαϊμούδων και απομίμηση αλλού εκτό Ευρώπη. Τρίτον, η άκτα θα ευθυγραμμίζεται, πρέπει να ευθυγραμμίζεται με το κοινοτικό και εκτιμένο και με το σημερινό βαθμό και επίπεδο της τυποποίησης όσον αφορά και τις ε, επικοινωνίες και τέλος την εφαρμοστέα νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ε, προστασία της ιδιωτικής σφαίρας και των προσωπικών δεδομένων. Δεν θα είναι κάτι το οποίο θα ε, περιορίζει δικαιώματα από πλευράς των καταναλωτών αλλά σε μια κλιμακούμενη διαδικασία θα τα προστατεύει. Τέταρτον, θα διασφαλίσουμε ότι η άκτα δεν θα παρακολεί την πρόσβαση στα ε, φάρμακα. Γνωρίζω ότι είχαμε σε ένα από τα κράτη-μέλη ένα προηγούμενο όπου με βάση τον νόμο για τους καταναλωτές τα generics, generic medicines είναι εκείνα τα οποία έχουν οδηγήσει κάποια φορά σε προβλήματα. Κατανοούμε ότι αυτό είναι προς όφελος της Ινδίας και της Βραζιλίας να υπάρξει μια αμαργοποίηση μεταξύ άκτα και των διαπραγματεύσεων και διατάξεων του ΠΟΕ. Για να υπογραμμιστεί αυτό το σημείο όμως η άκτα δεν αφορά, την άκτα δεν την αφορά αυτό. Και έτσι δεν θα έχουμε έλεγχο ε, πνευματικών δικαιωμάτων ή έλεγχο των ε, διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας. Έτσι λοιπόν για τα generics δεν θα έχει αυτό εφαρμογή και πρόκειται εδώ για τα θέματα και τη δημόσια υγείας. Δράτω με τι ευκαιρίες σύντομα να αναφέρω τα αποτελέσματα του ένα του γύρου διαπραγματεύσεων για την άκτα που έγιναν στη Λουκέρνη στις 28 Ιουνίου μέχρι 1 Ιουλίου θετική πρόοδος ε, σημειώθηκε στο κείμενο που διαπραγματευτήκαμε, αλλά πολλές φορές ε, εις βάρος της φιλοδοξίας ε, της εμβέλειας της ΑΚΤΑ και η προσπάθεια να μείνουμε στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού κεκτημένου πέτυχε. Και σε σχέση με ένα κείμενο που προηγούμενα δεν υπήρχε συμφωνημένο κείμενο για το πολυμερές πλαίσιο, η νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ήταν μια πολύ θετική πηγή έμπνευσης για τις συμβιβαστικέ προτάσεις που θα πρέπει να διέπουν μια συμφωνία σαν την Άκτα. Όμως σε σημαντικούς τομείς όπως την επιβολή του νόμου στα σύνορα, γίνεται σαφές ότι η συνένεση μεταξύ των ε, μπλεκομένων στην άκτα θα επιτευχθεί μόνο με τη βάση ενός ελάχιστου παρονομαστή. Μια και υπάρχουν πολυσχηδείς πρακτικές και διαφορές ε, στις πρακτικές αυτές μεταξύ των εταίρων. Ένας άλλος τομέας ε, όπου ήταν απογοητευτικές οι συζητήσεις όσον αφορά τα συμφέροντα της ΕΕ αφορά τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας που θα καλύπτονται από συμφωνία. Εδώ έχουμε πολυσχηδή βάση όσον αφορά τους δικαιούχους. Ένας ε, γεωργός ή μια εταιρεία κλωστοφαντουργικών και αυτοί μπορούν να είναι θύματα προϊόντων μαϊμούδων και αυτοί πρέπει να προστατεύονται από τους κανόνες επιβολής. Το πρόβλημα είναι ότι οι διάφοροι μας εμένουν και επιμένουν ότι μόνο τα εμπορικά σήματα και τα ε, διπλώματα ευρεσιτεχνίας ε, πρέπει να προστατεύονται και θα πρέπει να ασκηθεί πίεση αυτά να είναι σεβαστά πάντα. Ο δεύτερος γύρος ε, κατά τα τέλη Ιουλίου στη Ουάσιγκτον και ενώ προσεγγίζουμε την τελευταία αυτή φάση θα χρειαστούν και άλλοι περαιτέρω γύροι για να ολοκληρωθούν πλήρως οι διαπραγματεύσεις. Για τη διαφάνεια. Η ΕΕ έπεισε τους εταίρους της το κείμενο αυτό <clears throat> να δημοσιευθεί, να δημοσιοποιηθεί. Ήταν ισχυρό αίτημα του Κοινοβουλίου και έτσι με ικανοποίηση διαπιστώνουμε ότι δημοσιοποιήθηκε το κείμενο τον Απρίλιο. Υπήρξε και αντίρρηση ε, κάποιου σε σχέση με την δημοσιοποίηση του κειμένου όσον αφορά την πρόοδο της Λουκέρνης. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή <clears throat> εκφράζει την θλίψη της ε, για αυτή την ε, μονομερή ένσταση. Και έτσι λοιπόν δεν θα πρέπει να ξαναγυρίσουμε σε υποψίες σε σχέση με το έργο στη Λουκέρνη η πρόοδος έγινε με βάση το διαθέσιμο κείμενο και επειδή έπρεπε να επιτευχθούν διάφοροι συμβιβασμοί με εναλλακτικέ λύσεις επιτραπέζης δεν προσθέθηκαν νέες διατάξεις. Τούτων λεχθέντων με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με αυτό το κείμενο θα συνεχίσετε να ενημερώνεστε επί των αλλαγών από πλευρά μα. σε σχέση με, την, με το μηχανισμό που έχει δρομολογηθεί και σε σχέση με, τη, με ευαίσθητα διαπραγματευτικά κείμενα θα είναι στη διάθεσή σας το κείμενο. Το τονίζω ότι είναι μόνο για τη δική σας χρήση και δεν θα πρέπει να κυκλοφορήσει εκτός Ευρωκοινοβουλίου. Αυτή είναι η προϋπόθεση με την οποία μπορώ να διαθέσω το κείμενο σε εσά. Ενθαρρύνομαι από τις ε, δραστηριότητες ε, του Κοινοβουλίου. Είχαμε και ένα briefing, μια ενημέρωση για τη Λουκέρνη και αυτό είναι ένα παράδειγμα του διαλόγου που αναζητώ και επιζητώ εγώ να έχω μαζί σας. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας, Πρόεδρε. Thank you very much, Commissioner. Ευχαριστούμε κύριε Επίτροπε. Μέχρι στιγμής έχουν ζητήσει ένας δύο το λόγο. Κύριε Λαμπρινίδη, παρακαλώ. Ευχαριστώ και ευχαριστώ κύριε Επίτροπε για την παρουσία σας σήμερα εδώ και για την ενημέρωση που μας προσφέρατε. Όπως διαπιστώσαμε τους τελευταίους μήνες προσπαθώντας να αποκαλύψουμε πληροφορίες για την άκτα ψάχνοντας από εδώ και από εκεί ειδικά από τον Απρίλιο και μετά, διαπιστώσαμε ότι το πρόβλημα είναι στις λεπτομέρειες. Γενικές δηλώσεις λοιπόν ότι θα διατηρηθεί το ευρωπαϊκό κεκτημένο και τα λοιπά, καταλήγουν σε κάποιες μικρές υποσημειώσεις που μπορεί και να διαγραφούν στο μέλλον όπως έγινε με το Χαντόπι. Αν λοιπόν δεν έχουμε τελικό κείμενο μπροστά μας όπου βλέπουμε τελικά τι εγκρίθηκε, μιλάμε επί θεωρητικής βάσης. Εν πάση περιπτώσει, για τα πράγματα όσο έχουν σήμερα. Μιλάτε για τα σύνορα και την προστασία της διανοητικής ιδιοκτησία στα σύνορα. Κατά τη γνώμη σας, αποκλείεται σε κάθε περίπτωση να έχουν δικαίωμα οι συνοριακές αρχές ε, να εξετάζουν τα λάπτοπ ε, ή τα τηλέφωνα των ε, ταξιδιωτών ή επιτρέπεται αυτή η πρακτική στα πλαίσια της άκτα. Πρώτη ερώτηση. Δεύτερη ερώτηση. Το γεγονός ότι η άκτα δεν ε, αναγκάζει τις χώρες να εγκρίνουν νομοθεσία τύπου χαντόπι, δηλαδή τύπου τριών χτυπημάτων είναι το ένα θέμα. Το άλλο είναι αν θα αναγκάσουν τις εταιρείε να λάβουν μέτρα για να προστατεύσουν εαυτούς σε περίπτωση που προκύψουν θέματα αστικής ευθύνης. Γιατί στο παρελθόν είχε προταθεί από την άκτα ότι νόμοι τύπου Χαντόπι θα ήταν η μοναδική λύση για να μην μείνουν ξεκρέμαστες ιδιωτικές εταιρείες σε θέματα ευθύνης. Άρα, αν η νομοθεσία τύπου Χαντόπι δεν απαγορεύεται ρητός. Εγώ ως εταιρεία, ενδεχομένως μικρή εταιρεία, μπορεί να αναγκαστώ να διαγράφω πράγματα από τις ιστοσελίδες μου για να τη φοβάμαι διώξεις. Ενδεχομένως επίσης να βρεθώ αναγκασμένος να παρακολουθώ τους τρόπους που κατεβάζουν αρχεία οι χρήστες για να διασφαλίσω ότι δεν συμβαίνει κάτι στραβό. Άρα ενδεχομένως είτε σας υποχρεώνει είτε όχι να χρησιμοποιήσετε νομοθεσία τύπου αντόπι ή άκτα ίσως τελικά να σας ενθαρρύνει, να σας επιτρέπει να το κάνετε αυτό. Και θα θέλαμε να διασφαλίσουμε ότι δεν θα υπάρξει καμία τέτοια είδους αναφορά στην άκτα. Υπάρχουν και πολλά άλλα που θα μπορούσαμε να πούμε, αλλά δεν έχει αποφασιστεί κάτι ακόμη και θα ήθελα πολύ να διαβάσω το κείμενο, δεν ξέρω όμως πότε θα γίνει αυτό. Και ακόμη και αν τώρα το βράδυ το παρουσιάζατε, πάλι μάλλον η συζήτηση θα έπρεπε να γίνει τον Σεπτέμβριο, αργά σχετικά. Σε κάθε περίπτωση Υπάρχουν πολλά ακόμη να συζητήσουμε. Θα ακούσουμε μια σειρά από ερωτήσεις πρώτα και μετά απαντήσεις. Η κυρία Κέλλερ, θα συμφωνήσω με τα όσα υπόθηκαν και θα τονίσω ότι το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου δεν ζήτησε πρόσβαση στα έγγραφα μόνο για τους ευρωβουλευτές αλλά και για το γενικό κοινό που αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει. Οπότε θα θέλαμε να μάθουμε ποιο από τα μέρη είναι κατά αυτής της πρόσβασης και γιατί. Και στον τελευταίο γύρο θα εξακολουθήσει αυτό το μέρος να αντιτίθεται στην δημόσια πρόσβαση των τελευταίων εκδοχών του κειμένου. Θα παραμείνουμε δηλαδή μόνο με το κείμενο του Απριλίου, γιατί όπως υπόθηκε είναι δύσκολο να εκτιμήσουμε ποιες θα είναι οι συνέπειες των διαφόρων κεφαλαίων της Συμφωνίας της Άκτα. Και επίσης θα ήταν σημαντικό για μας να βρούμε εξωτερική υποστήριξη, αλλά δεν μπορούμε να το κάνουμε επειδή δεν υπάρχει πρόσβαση στο κοινό. Και επίσης θέλουμε να δούμε μελέτες επιπτώσεων για τις συνέπειες ε, στα φάρμακα και στην ε, μεταφορά τεχνολογίας. Γιατί κάθε φορά που μιλάμε για το κλίμα, για την πράσινη τεχνολογία και τα λοιπά, Πάντα μιλάμε για μεταφορά τεχνογνωσίας. Ποιες θα είναι οι συνέπειες εκεί. Και λέει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι δεν θα υπάρξουν συνέπειες για τα γενώσιμα φάρμακα. Πού είναι όμως οι αποδείξεις. Δεν υπάρχουν αποδείξεις μέχρι στιγμής. Είναι λοιπόν σημαντικές οι διατάξεις της άκτα που αφορούν ε, τις ε, τα εντάλματα, τα injections και άλλα τέτοια θέματα γιατί εμείς βλέπουμε ότι θα υπάρξουν περιορισμοί στα γενώσιμα φάρμακα. Μας ενδιαφέρουν όλα αυτά, αλλά αν δεν δημοσιεύετε τα κείμενα, μπορείτε να επαναλάβετε, να επαναλαμβάνετε όσες φορές θέλετε ότι δεν υπάρχουν συνέπειες, αλλά δεν θεωρούμε ότι αυτό μας διασφαλίζει. Χρειαζόμαστε λοιπόν μελέτες αντικτύπου, χρειαζόμαστε δημόσια πρόσβαση στα έγγραφα και θέλουμε να μάθουμε ποιοι είναι κατά αυτής της πρόσβασης. Και επίσης θέλουμε να ενημερώσουμε για το πώς οι ρήτρε διασφάλισης για την προστασία της ιδιωτικής ζωής, για τα γεννόσιμα φάρμακα κτλ θα υπάρχουν γιατί αυτή τη στιγμή δεν βλέπουμε τέτοιες ρήτρες διασφάλισης. Προβλέπεται να προσθεθούν και ανεπώς. Ναι, Αυτά και αναμένουμε με ανυπομονησία το συντομότερο δυνατόν το κείμενο. Ευχαριστώ ο κύριος Έντσου. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Κυρίως θα ήθελα να πω ότι ευχαριστώ και σκέπτεται να δημιουργήσει ένα νομικό πλαίσιο κυρώσεων η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αν δεν γίνονται σεβαστά τα πνευματικά δικαιώματα. Λαμβάνονται υπόψη οι κοινωνικο-οικονομικές επιπτώσεις αυτών των ζητημάτων. Είναι κάτι το απαράδεκτο θα έλεγα να έχουμε ισότιμη αντιμετώπιση πολύ σοβαρών παραβιάσεων και παραβάσεων όπως ε, την πειρατική δράση που έχει επιπτώσεις και στην υγεία και στην φυσική σωματική ακεραιότητα των ατόμων σε σχέση με πειρατικές ε, πράξεις εμπορίου κοσμητικών προϊόντων ε, ή άλλων. Και επίσης έχουμε και σε σχέση με το ηλεκτρονικό εμπόριο, το διαδίκτυο, ε, προϊόντα πειρατεία. Θα ήθελα να μου πείτε σε σχέση με το διαδίκτυο, σε σχέση με τις δράσεις και επιπτώσεις που έχουν στους πελάτες τους. Πρόκειται να υπάρξει μια εποπτεία και μια διήθηση, ένα φιλτράρισμα των πληροφοριών αυτών, διότι έχω υπόψη μου καταστάσεις στις οποίες το δικαίωμα δίκαιο και δικαίωμα της πνευματικής ιδιοκτησίας και των παράγωγων θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη. Ο κύριος Άλβαρο, παρακαλώ. Νόμιζα ότι είχατε ζητήσει τον λόγο. Α, δεν τον είχατε ζητήσει. Εντάξει. Τότε επανερχόμαστε στον Επίτροπο για να απαντήσει. Uh, Πρώτα απ' όλα όσον αφορά τους συνοριακούς ελέγχους, να το διασφαλίσω αυτό αν επιτρέπετε. Είναι και μια γενική απάντηση, γενικότερη απάντηση και προς την κυρία Κέλλερ. Τα ειχέγγυα στην συνθήκη φυσικά ζούμε σε ένα κράτος δικαίου αν κάτι δεν επιτρέπεται από τον νόμο, απαγορεύεται ρητά και κατηγορηματικά. Η γενική ρήτρα που ισχύει σε όλα είναι αυτή και για τους συνοριακούς ελέγχους. Μάλιστα, σε αυτή την πτυχή μπορώ να διασφαλίσω ότι δεν θα υπάρχουν έλεγχοι των λάπτοπ και των ηλεκτρονικών υπολογιστών και τα λοιπά των ταξιδιωτών στα σύνορα. Για παράδειγμα, το 2003 ε, νέα διάταξη τελωνιακή και έχουμε την διάταξη de minimis που εξαιρεί τους ε, ταξιδιώτες από ελέγχους όσον αφορά άγαθα όταν δεν είναι σε μεγάλη κλίμακα η διακίνηση και όταν έχουμε διακίνηση ναρκωτικών ή όπλων ε, όταν δεν υπάρχει για παράδειγμα νομική βάση σε σχέση όπως για παράδειγμα για τα λάπτοπ ή για τους υπολογιστές. Δεν υπάρχει κάποια πρόθεση να αλλάξει αυτό. Θα πρέπει να λάβετε υπόψη κύριε Λαμπρινίδη ότι αυτό είναι όχι μέρος της άκτα ουσιαστικά. Είναι μέρος και τμήμα του ευρωπαϊκού νομικού πλαισίου αν μπορεί να το κάνει κανείς αυτό ή όχι, της νομοθεσίας ε, του πρωτογενούς ε, δικαίου. Η άκτα είναι δευτερογενές δίκαιο. Αυτές ε, τις διατάξεις δεν μπορεί να τις βρει κανείς στην άκτα, αλλά θα πρέπει να αναφερθεί κανείς είτε στο ευρωπαϊκό δίκαιο είτε στο εθνικό δίκαιο. Ο λόγος για τον οποίο δεν το βρίσκεται αυτό στο κείμενο της άκτα είναι αυτός. Επειδή η άκτα αφορά διαδικασίες, διαργασίες για την επιβολή του νόμου. Δεν είναι για το τι μπορεί να επιβάλλει κανείς, αλλά για το πώς μπορεί να το επιβάλλει κανείς αυτό ως νόμο όσον αφορά το ε, δίκαιο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και το παράδειγμα το οποίο μόλις ε, έδωσα σε αυτή την κατεύθυνση έτεινε. Τώρα, αν αυτό θα ενθαρρύνει ή αποθαρρύνει ουσιαστικά τους ε, εμπλεκόμενους στο διαδίκτυο και τους παρόχους, πώς να το πω, ευαίσθητο περιεχόμενο να το διαθέτουν στους ε, ε, όσους χρησιμοποιούν το διαδίκτυο διότι θα υπάρξει η ε, προσέγγιση αυτή μέσω της χρήσης αυτής που δεν απαγορεύεται από την άκτα. Το θέμα είναι, η απάντηση είναι πάλι ίδια. Δεν υπάρχουν κράτη-μέλη που να έχουν μια τέτοια προσέγγιση η Γαλλία για παράδειγμα η οποία ακολουθεί με την δεν θα αλλάξει η άκτα λόγω αυτού είναι τα κράτη-μέλη που θα αποφασίζουν τι θα γίνεται για μια συγκεκριμένη χρονική στιγμή και η Ευρωπαϊκή Ένωση να κρίνει διότι η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση θα μπορούσε να υιοθετήσει νομοθεσία σε σχέση με αυτό αν μπορεί να έχει μια ε, πολιτική των τριών πληγμάτων ή όχι. Three strikes approach. Και έτσι σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση αν θα μπορούσε, αν ήθελε να υιοθετήσει νομοθετικό, νομοθετικές διατάξεις από αυτού, καθώς τώρα δεν υπάρχει σε ευρωπαϊκό επίπεδο, υπάρχει σε διεθνές επίπεδο. Στη Γαλλία όμως υπάρχει. Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι η άκτα θα είναι το εργαλείο για την επιβολή του νόμου. Όμως η χώρα μου δεν το έχει. Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι δεν μπορεί να επιβάλλεται στο Βέλγιο. Όμως ε, η εμπράγματη βάση του δικαίου είναι αυτή. Θα πρέπει να υπάρχει για να γίνει τέτοια χρήση. Αλλιώς δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Κυρία Κέλλερ τώρα, σε εσά στρέφομαι. Ποιος είναι ο αντιστεκόμενος, ο διαφωνών. Νομίζω είναι λίγο δύσκολο να σας το αποκαλύψω αυτό όμως. Αν δείτε το τι συνέβη στο παρελθόν μάλλον εύκολα θα βρίσκατε την απάντηση σε αυτό το ερώτημα που διατυπώσατε εσείς ίδια. Σίγουρα δεν είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά για κοιτάξτε τι έγινε στο παρελθόν και θα πάρετε σχεδόν αυτόματα θα σας δοθεί η απάντηση. Τούτου λεχθέντος, υπό αυτού τους όρους και προϋποθέσεις δεν μπορούμε να διαθέσουμε το κείμενο στους πολίτες ε, να το δημοσιοποιήσουμε σε όλους. Έχει όμως ε, δημοσιευθεί, είναι διαθέσιμο για ε, εσάς και μπορείτε να το δείτε και να το ελέγξετε και σε σχέση με την ερώτηση για τα ε, generics, τα φάρμακα, τα συσκευάσματα, απάντηση όχι, δεν θα έχει επιπτώσεις σε σχέση με αυτά. Και κατά τα άλλα, υπήρξαν προβλήματα στα σύνορα με τέτοιου είδους συσκευάσματα, επειδή οι τελωνιακές αρχές ήθελαν να επιβάλλουν την, ε, τα πνευματικά δικαιώματα επί υλικών προϊόντων, για παράδειγμα θέματα ε, διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας. Και ήταν κάθετη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και είπε ότι αυτό μπορεί να γίνει μόνο για να ελέγχεται αν υπάρχει απομίμηση, προϊόν απομίμηση μαϊμού γιατί σε σχέση με τα ιατρικά δεν είναι μόνο ότι δεν επιτρέπεται αλλά είναι και κακή πρακτική και έχει σοβαρές αρνητικές επιπτώσεις και ένα άλλο είναι τα προϊόντα μαϊμούδες φαρμακευτικά προϊόντα και σκευάσματα που πολλούνται στο διαδίκτυο διατίθενται εκεί και πολλές φορές εμπεριέχουν και επικίνδυνες ουσίες οι προϊόντα αυτά τα φάρμακα αλλά αυτό δεν θα έχει επιπτώσει, ως είπα, στα generics. Και το καταστήσαμε σαφές επίσης και στις Ινδικές αρχές της Ινδίας, ότι θα διασφαλίσουμε ότι δεν θα υπάρξει άλλη τέτοια περίπτωση. Και γι' αυτό δεν κατανοώ γιατί όλοι ξαφνικά ζητούσαν να γίνουν διαβουλεύσεις, διότι ήταν απόλυτα σαφές προς τις Ινδικές αρχές ότι ήταν σαφές ότι σε σχέση με την ε, Συμφωνία Ελευθέρου Εμπορίου που διαπραγματευόμαστε με αυτούς, ότι αυτό θα ρυθμίζεται και δεν θα έχει επιπτώσεις σε αυτά τα ιατρικά σκευάσματα. Τώρα, φάρμακα. Προστατεύονται και αυτά με διπλώματα ευρεσιτεχνίας, έτσι τα οποία όμως δεν καλύπτονται σε σχέση με τα σύνορα, σε σύνοριακούς ελέγχους. Αυτό βρίσκεται εκτός επιβολής άκτα, λοιπόν. Αν κάναμε μελέτες επιπτώσεων, ρωτήσατε. Δεν νομίζω ότι οι μελέτες επιπτώσεων θα ήταν υποφελεί με οποιοδήποτε τρόπο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν θα ξεπεράσει τα όρια του κοινοτικού κεκτημένου. Βασιστήκαμε στις μελέτες που είχαν γίνει σε σχέση με την οδηγία του 2004 για την επιβολή των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, για την πρόταση του 2005 για την ε, επιβολή της ε, IPR που δεν έχει ακόμα εγκριθεί και επίσης και τα συμπεράσματα της μελέτης του ΟΣΑ για τις οικονομικές επιπτώσεις των προϊόντων πειρατείας του 2008 και αυτή η μελέτη αξιολογεί τις επιπτώσεις στην οικονομία των προϊόντων απομίμησης σε 250 δις δολάρια υψηλότερο δηλαδή από το ΑΕΠ δεκάδων χωρών και εμπεριέχει επίσης και μια εξαντλητική ανάλυση όσον αφορά την πειρατεία ε, ψηφιακού περιεχομένου. Αλλά θα χρειαζόμαστε πάλι συγκεκριμένες εξειδικευμένες μελέτες επιπτώσεων. Επίσης κατανόησα ότι του είδου ή ε, τις μελέτες επιπτώσεων που θα θέλετε να έχετε δεν είναι αυτές αλλά άλλες. Αυτές είναι για την οικονομική επίπτωση. Εσείς θα προτιμούσατε να είχατε μια μελέτη επιπτώσεων για τις υλικές επιπτώσεις και συνέπειε. Και αν αυτό δεν αντιμετωπίζει το ουσιώδες πρόβλημα μια και δεν είναι επί ή του εμπραγμάτου δικαίου αλλά επί των διεργασιών και διαδικασιών άκτα. Μπορεί να έχει κανείς μια μελέτη επιπτώσεων, οικονομικών επιπτώσεων ή και άλλων αλλά αυτό δεν αλλάζει τίποτα στο περιεχόμενο της άκτα. Μόνο μπορεί να καταστήσει σαφές σε κάποιους ότι είναι σημαντικό να υπάρξει μια τέτοια σύμφωνία επειδή τα οικονομικά συμφέροντα είναι τεράστια σημασία. Ειλικρινά πρέπει να πω ότι δεν κατάλαβα κύριε από τη Ρουμανία την ερώτησή σας. Ίσως φταίω εγώ γι' αυτό. Εν πάση περιπτώσει δεν κατανόησα το νόημα της ερώτησής σας. Περί τίνο επρόκειτο. Και προτού επανέλθω σε αυτό τώρα, θα ήθελα να πω κάτι. Ανέφερα στην εισαγωγή μου πιο πριν ότι ακόμα έχουμε πολλές αρκετές διαφωνίες για την άκτα μεταξύ των ε, εμπλεκομένων στις διαβουλεύσεις ε, και μία από τις μεγαλύτερες διαφωνίες είναι ότι οι περισσότεροι από τους διαπραγματευόμενους μόνο θα ήθελαν να υπάρχει η προστασία του copyright και των trademarks και δεν είναι πρόθυμοι να κάνουν το ίδιο και για σχέδια, designs ή για γεωγραφικές επισημάνσεις ή ενδείξεις. Τώρα, αυτό είναι η κόκκινη διαχωριστική γραμμή θα έλεγα. Αν δεν καταφέρουμε να πετύχουμε τα σχέδια, designs και οι γεωγραφικές ενδείξεις να συμπεριληφθούν, διαρωτώ ποιο θα ήταν το μεγάλο όφελος αυτής της συμφωνίας στο τέλος τέλος. Ας σας δώσω ένα παράδειγμα. Πρόσφατα διαπραγματευθήκαμε μια συμφωνία ελευθέρου εμπορίου με τα κράτη της Κεντρικής Αμερικής Θέλαμε οι γεωγραφικές αυτές αναφορές για προϊόντα να προστατεύονται. Καταλήξαμε στο συμπέρασμα ή το ανακαλύψαμε κιόλας ότι οι Αμερικανοί στη Συμφωνία Ελευθέρου Εμπορίου που έχουν συνάψει με τα κράτη της Κεντρικής Αμερικής προστάτευαν αρκετά trademarks. Όμως το περιεχόμενο αυτών των trademarks ήταν ακριβώς το ίδιο με αυτό το οποίο εμεί αποκαλούμε γεωγραφικές, ε, ε, γεωγραφικούς χαρακτηρισμούς. Φυσικά τα trademarks ήδη προστατευόντουσαν. Εμείς δεν μπορούσαμε να προστατέψουμε το ίδιο περιεχόμενο είτε με γεωγραφικές ενδείξεις είτε με trademarks. Χρησιμοποιούμε για τον ίδιο, αν χρησιμοποιούν, ε, για τον ίδιο στόχο τότε να το κάναμε. Αλλά αρχίζει μια, ας το πω έτσι, προσέγγιση να αποκαλύπτει αυτή την ε, υποκρισία, ε, υποκριτική προσέγγιση. Είναι η κόκκινη διαχωριστική γραμμή επιτέλους αυτή. Τώρα θα διαβουλευτούμε από πλευρά τη Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τα κράτη-μέλη και θα καταστήσουμε σαφές ε, και στις αρχές των ΗΠΑ ότι δεν μπορούμε να το δεχτούμε αυτό, να το καταπιούμε έτσι ίσως μπορούμε να έχουμε κάποιες συζητήσεις για το εύρος και, το, την έκταση του τι θα καλύπτεται και ποιες χώρες θα είναι εκείνες που όχι μόνο θα έχουν δικαίωμα αλλά και θα είναι και υποχρεωμένες να το επιβάλλουν αν σε σχέση με ένα τέτοιο σύστημα που δεν θα υπάρχει γεωγραφικών επισημάνσεως, πώς θα μπορεί να γίνει, θα είναι δύσκολο. Αλλά αν το κάνουμε από το, από το παραθυράκι, όπως για τα trademarks, θα έλεγα ότι είναι εκτός της ευστάθειας και ισορροπίας που απαιτείται να, να υιοθετήσουμε. Και τώρα είναι ένα θέμα αυτό. Επίσης για την ερώτηση αν θα ήταν δυνατό να επανέλθουμε σε σχέση με αυτό πριν από την έναρξη, την επανέναρξη των κοινοβουλευτικών εργασιών που θα αρχίσουν στις αρχές Σεπτεμβρίου. Λοιπόν, να τοποθετηθώ σε εξής και να πω ότι αν κάτι ήταν να συμβεί, συμβεί κάτι μέσα στις διακοπές επειδή ένας νέος γύρος διαπραγματεύσεων θα γίνει κατά τέλη Ιουλίου θα σας ενημερώσουμε εμείς δεν θα κατεβάσουμε τα ρολά και θα κλείσουμε το μαγαζί κατά τη διάρκεια των διακοπών αλλά κατά την έναρξη του νέου κοινοβουλευτικού ε, έτους η κατάσταση δεν νομίζω θα είναι τόσο ε, ριζοσπαστικά διαφορετική. Δεν νομίζω ότι θα έχουμε καταφέρει να έχουμε επιλύσει όλα τα άλλα προβλήματα. Εκτός αν υπάρξει αυτό το οποίο σας είπα. Αν υπάρξει ένα split σε σχέση με τους ε, διαπραγματευόμενους. Ιδιαίτερα όσον αφορά <clears throat> του τι θα έπρεπε να είναι για το τι θα έπρεπε να καλύπτουν τα πνευματικά δικαιώματα και πώς θα ρυθμιστούν αυτά μέσω της ΣΑΤΚΑ Ίσως εσείς κύριε Άντσου μπορείτε να εξηγήσετε κάπως περισσότερο αυτά τα οποία θέλατε να πείτε γιατί δεν κατανόησα απόλυτα την παρέμβασή σας. Ο κύριος Λαμπρινίδης θέλει να επανέλθει και ο κύριος Όλτραχτ έχει επίσης ζητήσει το λόγο. Παρόλο που είστε λίγοι, θα ήθελα να συζητήσω να είστε σύντομοι. Κύριε Έντσου, μπορείτε να εξηγήσετε τι εννοούσατε πριν. Ναι. Σε αυτόν τον κατάλογο των νομικών μέτρων τα άτομα τα οποία θα παραβιάζουν τους κανόνες της πνευματικής ιδιοκτησίας θα τιμωρούνται. και βάζεται στο ίδιο επίπεδο τα, την κατασκευή φαρμάκων μαϊμούδων με τον έφηβο ο οποίος φορτίζει παράνομα ένα τραγουδάκι από το ίντερνετ. Δηλαδή είναι δύο διαφορετικών δύο διαφορετικές μορφές ε, απομίμησης. Άλλο είναι το να φορτώνει κανείς στον υπολογιστή του ένα τραγουδάκι και άλλο είναι να παρασκευάζει φάρμακα μαϊμούδες. Όσον αφορά το κατέβασμα από το ίντερνετ, ήμουν σαφής νομίζω ότι πρέπει να μιλάμε για ευρείας κλίμακα κατάσταση. Τώρα, όσον αφορά τις απομιμήσεις φαρμάκων, πρέπει να γνωρίζετε ότι ακόμη και πολύ μικρές ποσότητες μπορεί να είναι επικίνδυνες. Τίθεται θέμα δημόσιας υγείας και έχουν ε, το καθήκον, ναι, το δικαίωμα οι αρχές να εξετάζουν αυτές τις περιπτώσεις, να ελέγχουν αν εισάγονται επικίνδυνα προϊόντα. Θα έλεγα ότι είναι καλό το γεγονός ότι ακόμη ότι ελέγχονται ακόμη και μικρές ποσότητες, όχι για το αν προστατεύονται ή όχι από δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, αλλά για το αν περιέχουν επικίνδυνες ουσίες. Δεν έχει να κάνει εδώ με την ευρεία κλίμακα, τη μεγάλη ποσότητα, αλλά με τον κίνδυνο. Κάποιος που αγοράζει φάρμακα από το ίντερνετ, μπορεί να έχει πολύ σημαντικό πρόβλημα. Ειδικά εφόσον υπάρχουν και βλαβερές τέτοιες ουσίες. Δεν ξέρουμε πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε την νομοθεσία εδώ, αλλά δεν πρόκειται για θέμα διαδικαστικό. Είναι θέμα ουσίας. Δεν πρέπει να επιτρέπουμε την εισαγωγή στην ευρωπαϊκή αγορά και στις χώρες μας επικίνδυνων ουσιών. Πολύ σύντομα κύριε Λαμπρινίδη. Κύριε Επίτροπε, δεν θέλω να μιλάω για βαρετές λεπτομέρειες που γνωρίζετε ήδη. Ε, γιατί είναι τόσο ευαίσθητο το θέμα, ειδικά όσον αφορά την προστασία της διανοητικής ιδιοκτησίας είναι ευαίσθητο γιατί υπήρξε τρομερή ποσότητα λόμπιν από τους γνωστούς υπόπτους εταιρείες κινηματογραφικές, μουσικές κτλ. με το επιχείρημα και χωρίς να θέλω να γίνω ηρωνικός, γιατί κανένας εδώ δεν θεωρεί ότι οι ιδιοκτήτες πνευματικής ιδιοκτησίας δεν πρέπει να λαμβάνουν αυτά που δικαιούνται. Όμως, τον 20ο αιώνα υπήρξε ένα καθεστώς για την προστασία διανοητικής ιδιοκτησίας. Και πολλοί ανησυχούν ότι αντί να προσπαθούν να βρουν νέους τρόπους ώστε να διασφαλίζεται η κατάλληλη αποζημίωση των δημιουργών και η χρήση του ίντερνετ χρησιμοποιείται η άκτα για να διατηρήσει κάποιες υπάρχουσες πρακτικές. Ερώτηση. Τι συμβιβασμό έχετε βρει όσον αφορά της ε, εμπορικής κλίμακας ε, λήψη από το ίντερνετ στην ε, Συμφωνία Άκτα. Συμπεριλαμβάνεται στη Συμφωνία άκτα στη νέα εκδοχή της και η δυνατότητα δίωξης σε άλλες περιπτώσεις ή υπάρχει πρόβλεψη μόνο για την εμπορική χρήση σε ευρεία κλίμακα. Και κάτι άλλο. Υπήρχε μία πρόταση να υποχρεώνονται οι πάροχοι ίντερνετ να δίνουν στις, ε, στους ιδιοκτήτες πνευματικής ιδιοκτησίας τα στοιχεία, τα ονοματεπώνυμα των χρηστών που κατεβάζουν περιεχόμενο. Γιατί γίνεται αυτή η συζήτηση και από ποιους να είναι υποχρεωμένοι οι πάροχοι ίντερνετ να ενημερώνουν άλλες ιδιωτικές εταιρείες για τις δραστηριότητες της δικές μου ή του οποιοδήποτε. Αυτά είναι πολύ ανησυχητικά θέματα και θέλουμε να γνωρίζουμε πού βρίσκονται διαπραγματεύσεις σήμερα, στο τελευταίο κείμενο. Γιάννα Άλμπρεχτ, τελευταίος ε, ομιλητής. Σας ευχαριστώ. Έχω τρία σημεία που θα ήθελα να αναφέρω. Πρώτα απ' όλα, Νομίζω ότι πρέπει να το αναφέρουμε κάθετα και κατηγορηματικά. Το ψήφισμά μας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έλεγε ότι θέλουμε η άκτα να είναι να περιορίζεται στον πυρήνα των συμφερόντων. Δηλαδή μέτρα κατά των προϊόντων απομίμησης, κατά των προϊόντων μαϊμούδων. Δηλαδή αυτό σημαίνει για μένα ότι η παραβίαση πνευματικού δικαίου και της πνευματικής ιδιοκτησίας δεν βρίσκεται σε αυτό το πυρήνα αρμοδιοτήτων ή στόχων που θέλουμε να ρυθμίζονται και να αντιμετωπιστούν. Η αντιμετώπιση προϊόντων απομίμησης είναι προϊόντα μαϊμούδες προϊόντα, ας το πω έτσι, ε, μαϊμούδες όσον αφορά ε, εμπορικά σήματα και δεν είναι η ε, πνευματική ιδιοκτησία. Πρέπει να γνωρίζουμε λοιπόν τι λέει το Κοινοβούλιο και να το σεβόμαστε σε ένα ευρύτερο πλαίσιο όσον αφορά το πλαίσιο αυτού του ψηφίσματος που εγκρίθηκε από εμά. Είναι απόλυτα σαφές για μας ότι αν η άκτα ξεπεράσει το κοινοτικό κεκτημένο δεν θα τύχει πλειοψηφία και έγκριση από το Ευρωκοινοβούλιο. Και αυτό είναι σαφέ μήνυμα του δικού μα ψηφίσματα και πρέπει να το ξέρετε αυτό εκ προημίου, από πιο πριν. Και αυτό σημαίνει ότι επίση όταν κάνετε λόγο για, για παράδειγμα για το μηχανισμό των τριών βημάτων ή πληγμάτων, three strikes mechanism, πρέπει να δείτε τις σοβαρές, σοβαρούς περιορισμούς. Δεν είναι δυνατόν τα κράτη-μέλη να υπονομεύουν σταθερά και ισχυρά εχέγγυα και διασφαλίσεις που έχουν αποφασιστεί στο ευρωπαϊκό επίπεδο. Ακόμα και στις διαπραγματεύσεις. Δεν μπορείτε να αναφέρετε στα κράτη-μέλη αυτό εκείνα να αποφασίζουν κατοδοκούν το δοκούν γιατί υπάρχει κοινοτικό δίκαιο και πρέπει να είναι σεβαστό. Να είναι σεβαστό και σε σχέση και με διεθνείς συμφωνίες που μπορεί βέβαια κανείς να τις διαπραγματευτεί αλλά πρέπει να ευθυγραμμίζονται απόλυτα με αυτέ τι αποφάσει ε, και αρχέ. Γιατί διαφορετικά θα υπάρχει ασυμβατότητα. Και η Ευρωβουλή το ανέφερε ότι κάτι τέτοιο δεν είναι κάτι το οποίο θα δεχόμαστε εμεί αν συνέβαινε. Και στο τέλος τέλος ουσιαστικά πρόκειται για τα θεμελιώδη δικαιώματα και για το κράτος δικαίου τη ένωμη τάξη. Είναι πολύ ευαίσθητο το θέμα. Όταν κάνουμε λόγο για μέτρα για τι ευθύνε ISP, και ποινικέ κυρώσει που θα έπρεπε να εξετάζονται σε ένα τέτοιο πλαίσιο διαπραγματεύσεων. Διότι αυτό είναι ένα τομέα όπου το Κοινοβούλιο πρέπει να εμπλέκεται όταν έρχεται ένα τέτοιο θέμα νέων μέτρων, νέων ρυθμίσεων και διατάξεων. Καλύτερα θα ήταν να το κάναμε ευθύ εξ αρχή από μηδενικού σημείου, αντί να προσπαθήσετε να παρακάμψετε αυτή τη δυνατότητα εμπλοκή του Κοινοβουλίου. Και στο τέλος τέλος είναι σημαντικό επίσης πραγματικά εμείς όχι μόνο να έχουμε μέτρα για την επιβολή του νόμου διεθνώς συμπεφωνημένα αλλά και διασφαλίσεις και ρήτρες ασφάλειες και εξαιρέσεις που θα συμφωνούμε και για την τεχνογνωσία και τη μεταφορά της ε, για πράγματα επί των οποίων έχουμε άλλη πολιτική όπως για την πολιτική ανάπτυξη για παράδειγμα και θέλουμε αυτά να είναι σεβαστά. Είναι σημαντικά για το Κοινοβούλιο αυτά τα θέματα. Ευχαριστώ. Okay, Ευχαριστώ. Κύριε Επίτροπε. Ευχαριστώ. Καταρχάς, για τον κύριο Λαμπρινίδη, η εμπορική κλίμακα δεν είναι κάτι που ορίζεται στην Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Αυτό σημαίνει ότι ο ορισμός της εμπορικής κλίμακας από κάθε κράτος μέλος θα ισχύσει ως κανόνας, είτε πρόκειται για νόμο ή δικαστήριο. Βλέπω ορισμό στο άρθρο 2, σημείο 1 1-4. Εκεί υπάρχει ορισμός για το τι είναι η εμπορική κλίμακα. Αν κάποια διεθνής ε, συμφωνία συμπεριέχει ορισμό, τότε θα υπερισχύει της εθνικής νομοθεσίας. Ναι, λέει ο Επίτροπος, αν συμπεριληφθεί στη Συμφωνία Άκτα. Τώρα, όσον αφορά τους παρόχους ίντερνετ, ευθυγραμμίζεται πλήρως με την οδηγία για το ηλεκτρονικό εμπόριο και δεν θα δημιουργηθούν νέες υποχρεώσεις. Στον κύριο Άμπρεχτ. η ύπαρξη αστυνόμευσης είναι απαραίτητη γιατί τα οικονομικά συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης προβλέπουν την προστασία της ιδιωτικής ε, ιδιοκτησίας. Για παράδειγμα, προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων, προστασία του copyright ε, στους τομείς ε, της τέχνης και της ψυχαγωγίας. Τώρα, όσον αφορά τη διαφάνεια και το πού βρίσκονται οι διαπραγματεύσεις, στην παράγραφο 9, στο έγγραφο του Μαρτίου, υπάρχει συγκεκριμένη αναφορά στην παραποίηση δεν είναι σαφές αλλά μπορεί να θεωρηθεί ότι συμπεριλαμβάνονται και οι παραποίησεις εδώ ενώ στην παράγραφο 10 αναφέρονται και τα copyright αλλά όχι η, διανοητικές, η διανοητική ιδιοκτησία. Το ψήφισμα λοιπόν αυτό του Μαρτίου ζητά εφαρμογή της ευρωπαϊκής νομοθεσίας και διαπραγμάτευση στα πλαίσια της ε, ευρωπαϊκής νομοθεσίας που είναι αυτό ακριβώς που κάνουμε. Δεν θα ελέγχει άκτα τις ποινικέ κυρώσεις στις περιπτώσεις ε, παραβιάσεων ειδικά στην περίπτωση γεννόσιμων φαρμάκων. Αυτό ευθυγραμμίζεται με την ε, συμφωνία TRIPS ε, που ζητάει διαπραγματεύσεις για όλες τις παραβιάσεις ε, διανοητικής ιδιοκτησίας αλλά στο συνδυασμό εγκληματικών και τελωνιακών παραβιάσεων είναι διαφορετικές οι διατάξεις που ισχύουν. Επίσης, οι ρήτρε διασφάλισης του TRIPS θα ισχύουν και για την άκτα. Σας ευχαριστούμε πολύ κύριε Επίτροπε. Νομίζω ότι τελείωσε και ο χρόνος μας και ο χρόνος σας και οι ερωτήσεις. Σας ευχαριστούμε πολύ που ήρθατε σήμερα. Θα δώσω την Προεδρία στον κανονικό Πρόεδρο που έφτασε εν τω μεταξύ στη συνεδρίαση για να συνεχίσουμε. Bon, bon. Καλησπέρα αγαπητοί συνάδελφοι. Καθίστε παρακαλώ. Θα συνεχίσουμε. Με συγχωρείτε που δεν μπόρεσα να παραβρεθώ στο πρώτο τμήμα της συνεδρίασης της ΛΥΜΠΕ γιατί είχα παγιδευτεί λόγω αναπόφευκτων υποχρεώσεων στην Ισπανία. Ευχαριστώ όμως την αξιότιμη συνάδελφο την Σόφιν Ντεφέλτ που προέδρευσε στην Επιτροπή νωρίτερα. Θα συνεχίσουμε τώρα από εκεί που είχαμε σταματήσει με το επόμενο σημείο στην ημερήσια διάταξη που είναι μια παρουσίαση της μελέτης για τη σχέση μεταξύ οργανωμένου εγκλήματος και διαφθοράς. Η παρουσίαση αυτή θα γίνει από το Κέντρο για τη Μελέτη της Δημοκρατίας. Η μελέτη έχει δημοσιευτεί σε δύο τόμους και αφορά ένα θέμα πολύ ενδιαφέρον για όλους τους συναδέλφους στην Επιτροπή ΛΥΜΠΕ αλλά και όλους τους άλλους που ενδιαφέρονται για την ελευθερία και την καταπολέμηση όλων των μορφών οργανωμένου εγκλήματος, ειδικά όταν συνδέεται με την διαφθορά εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο κύριος Στέφανο θα λάβει το λόγο για την παρουσίαση. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, αξιότιμοι ευρωβουλευτές. Χαίρομαι που βρίσκομαι σήμερα εδώ. Έχουμε κάνει κάποιες μικρές αλλαγές ε, στην παρουσίαση από αυτό που βλέπετε στους φακέλους σας γιατί προσπαθήσαμε να τη συντομεύσουμε για να έχουμε περισσότερες περισσότερο χρόνο στη διάθεσή μας. Θα προσπαθήσω να είμαι σύντομος ε, και να τελειώσω την παρουσίαση σε μισή ώρα. Ξεκινάω εγώ και μετά θα ακολουθήσουν ο ε, κύριοι Στογιάνοφ και Φίλιπ Γκολφ στο τέλος θα έχουμε και κάποιες υποδείξεις προς το Κοινοβούλιο, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το πώς θα μπορούσαν να δράσουν. Ξεκινάω με μία σύντομη παρουσίαση του Κέντρου για τη μελέτη της δημοκρατίας. Μετά θα περάσω σε κάποια βασικά θέματα όσον αφορά τη μεθοδολογία που χρησιμοποιήσαμε. Μετά θα κάνουμε την ε, βασική ανάλυση της σχέσης ε, οργανωμένου εγκλήματος και διαφθοράς και τέλος θα έχουμε τα συμπεράσματα και τις επιδείξεις, ε, υποδείξεις με συγχωρείτε. Το κέντρο δημιουργήθηκε το 1990 και τα τελευταία 20 χρόνια είχαμε τρεις βασικές δραστηριότητες. Έρευνα, ευαισθητοποίηση του κοινού Ελπίζουμε ότι συνεισφέραμε στη δημιουργία μιας δημοκρατικής κοινοοικονομικής κοινωνικής και δημοκρατικής μάλλον οικονομίας στη Βουλγαρία και στην Ευρώπη. Και τέλος ασχοληθήκαμε με θέματα που έχουν ευρωπαϊκό αντίκτυπο. Το κέντρο τα τελευταία χρόνια έχει ασχοληθεί με διάφορα θέματα. Επίσης έχουμε και κάποιες θεσμικές ε, συμφωνίες. Για παράδειγμα είμαστε το focal point, το κέντρο επαφής στη Βουλγαρία για το θεμελιώδη δικαιώματα. Επίσης έχουμε ασχοληθεί με το, συμμετέχουμε στο δίκτυο ανάπτυξης και είμαστε μία οργάνωση που βασίζεται σε έργα. Δηλαδή η χρηματοδότησή μας ε, προέρχεται από τα τιμολόγια, τα έσοδα που έχουμε από διάφορα έργα. Τα τελευταία χρόνια ο προϋπολογισμός μας ήταν περίπου ένα εκατομμύριο κατά έτος. Έχουμε συνεργαστεί με το Κέντρο για την Δικαιοσύνη, Ασφάλεια και Εσωτερικές Υποθέσεις για μελέτες. Επίσης με τη ΓΑΜΑ ΔΕΛΤΑ έρευνας στα πλαίσια του 7ου προγράμματος πλαισίου για τη συνεργασία σε δικαστικά θέματα. Τώρα, λίγα πράγματα για το ευρωπαϊκό πλαίσιο της έρευνάς μας και τη σημασία του. Νομίζω ότι όλοι στην Ευρώπη γνωρίζουμε πλέον ότι υπάρχουν ακόμη περισσότερες διασυνδέσεις εξαιτίας της κρίσης. Υπάρχουν πολλά προβλήματα που παραμένουν στον τομέα της ε, δικαιοσύνης και εσωτερικών υποθέσεων και η διαφθορά και το οργανωμένο έγκλημα έχουν πολλές διασυνδέσεις και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Οι ευκαιρίες που έχουμε με την νέα συνθήκη της Λισαβόνας καθώς και οι εθνικές πολιτικές ατζέντε όλες μας οδηγούν στο να δείξουμε ότι χρειαζόμαστε πολύ περισσότερη ευρωπαϊκή ενασχόληση. Και δίνω τώρα το λόγο στον κύριο Στογιάνοφ για να σας μιλήσει για το πλαίσιο της έρευνας και τη μεθοδολογία της. Σας ευχαριστώ. Ο κύριος στόχος αυτής της ε, μελέτης και ιδιαίτερα η διασύνδεση μεταξύ αυτών είναι να δώσουμε τα στοιχεία και το πλαίσιο για μελλοντικές αναλύσεις, έρευνα και κοινοτική δράση για τα κράτη-μέλη και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ο εξαιρετικός έκτακτος χαρακτήρας αυτού του εγχειρήματο βρίσκεται στο γεγονός ότι δεν υπάρχει μια κοινή κατανόηση και προσέγγιση ξεκινώντας από τους ορισμούς και φτάνοντας στο να έχει κανείς αντικειμενικά στοιχεία για τη δραστηριότητα, τη δράση του οργανωμένου εγκλήματος στα κράτη-μέλη. Για αυτούς τους λόγους, οι κυριότεροι στόχοι αυτής της μελέτης θα μπορούσαν να ήταν εν συνόψη τα εξή τρία σημεία. Να δούμε τους παράγοντες ε, της διαφθοράς ε, και του οργανωμένου εγκλήματος και ιδιαίτερα η διασύνδεση μεταξύ διαφθοράς και οργανωμένου εγκλήματος ποιες επιπτώσεις έχουν. Αυτό είναι ένα γνωστό θέμα. Το πρόβλημα είναι να χαρτογραφήσουμε και να έχουμε μια σφαιρική εποπτεία πώς αυτή η διασύνδεση εκφράζεται στα διαφορετικά κράτη-μέλη συγκεκριμένα. Δεύτερον, να εντοπίσουμε και ταυτοποιήσουμε τις βέλτιστες πρακτικές στην αντιμετώπιση της διαφθοράς και του οργανωμένου εγκλήματο στα κράτη-μέλη. Και τρίτο, να καταλήξουμε σε συμπεράσματα και ε, στοιχεία για μια, ένα μελλοντικό πλαίσιο ανάλυσης ε, και καταπολέμησης του οργανωμένου εγκλήματος που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί σε όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως πλαίσιο. Τώρα, η προσέγγιση και τα πρώτα εμπόδια τα οποία αντιμετώπισε η μελέτη μας ήταν ουσιαστικά να υπάρξει μια επισκόπηση ορισμών και να ξεκινήσουμε σε σχέση με αυτά τα στοιχεία για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος της διαφθοράς. Αυτό το οποίο είναι σχετικά καινούριο νέο στοιχείο σε αυτή τη μελέτη είναι το ότι η διαφθορά ιδιαίτερα σε σχέση με το οργανωμένο έγκλημα στο οργανωμένο έγκλημα έχουμε συμπεριλάβει επίσης ευρείας κλίμακας εγκλήματα συγκεκριμένες παράνομες αρμοδιότητες όσον αφορά και αγορές επίσης και σε σχέση με τις δραστηριότητες ποιος συνδέεται με αυτές και ποιος συνδέεται με συγκεκριμένες αγορές. Κάτι άλλο καινούριο στοιχείο στον ορισμό είναι είναι λέω ότι συγγνώμη λέει ο μιλητής και διακόπτη ο ιδιωτικός τομέας καλύφθηκε. Είναι ένα θέμα όμως κάπως αντιφατικό αυτό, διότι η διαφθορά στον ιδιωτικό τομέα αναφέρεται ως απάτη ο συνήθως και αφήνεται εκτός πλαισίου, εκτός ανάλυσης διαφθοράς και οργανωμένου εγκλήματος, διότι η διαφθορά θεωρείται κυρίως ότι είναι διαφθορά κρατικών υπαλλήλων ή κρατικών αξιωμάτων προς ίδιο προσωπικό όφελος. Λοιπόν, το συγκεκριμένο, ένα άλλο συγκεκριμένο τμήμα, το οποίο συνδέεται με την ε, μελέτη, είναι η μέτρηση του οργανωμένου εγκλήματος. Είναι ένα αρκετά καθόδες ε, και δύσκολο θέμα αυτό και προσπαθήσαμε να αναφερθούμε σε δείκτες, αντικειμενικούς δείκτες. Και τι εννοώ αντικειμενικούς δείκτες για το οργανωμένο έγκλημα. συλλέξαμε στοιχεία με δείκτες με αναφορά σε δραστηριότητες και τον όγκο αγορών. Για παράδειγμα, για την παράνομη αγορά ναρκών. Είναι ένας δείκτης του επίπεδου στο οποίο το οργανωμένο έγκλημα δρά σε μια συγκεκριμένη χώρα, ακολουθώντας την υπόθεση εργασίας ότι αν και όταν είναι αρκετά μεγάλος ο όγκος αγοράς, πιθανότητα υπάρχουν κάποιες δυνάμεις που εκμεταλλεύονται και χειραγωγούν, κάποιες ομάδες ή άτομα που δρούν παράνομα σε αυτές τις χώρες προς ίδιον όφελος. Όσον αφορά τώρα τη μεθοδολογία, μεθοδολογικά για αυτή τη μελέτη, τι κάναμε. Η μεθοδολογία συμπεριλαμβάνει διαφορετικές, διάφορες μεθόδους Πρώτα, ως ήθιστε, έχουμε μια επισκόπηση της βιβλιογραφίας, μια αστοποστάθμιση, αξιολόγηση στοιχείων που είναι στη διάθεσή μας για ε, το οργανωμένο έγκλημα και διαφθορά. Μελέτες που έχουν συνταχθεί σε διαφορετικές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεύτερο, Το δεύτερο κυριότερο τμήμα της ερευνητικής μεθοδολογίας ε, συμπεριλαμβάνει μια στατιστική ανάλυση περίπου 105 δικτών που μετρούν διαφορετικές πτυχές της διαφθοράς και του οργανωμένου εγκλήματος, διαφορετικές συνιστώσεις ως παραμέτρους. Η αξία αυτής της ανάλυσης είναι ότι με βάση αυτή είμαστε σε θέση να διαρευνήσουμε δύο μείζωνα θέματα. Πρώτο, το αν υπάρχουν στατιστικά σημαντικοί δεσμοί και διασυνδέσεις μεταξύ διαφθοράς και οργανωμένου εγκλήματος. Είναι μια αμφίδρομη, ας το πω έτσι, ένας αμφίδρομος συσχετισμός και εξάρτηση. Αν αυτό θα μπορούσε να συσχετιστεί με κάποια συγκεκριμένα χαρακτηριστικά και ιδιομορφίες ή ιδιότητες ε, των κρατών μελών κάποιες χώρες μπορούν να κατηγοριοποιηθούν, να ομαδοποιηθούν κατά κάποιο τρόπο, ώστε να μειώσουμε τις ε, παραλλαγές ε, και τις διακοιμάσεις όσον αφορά την πολυπλοκότητα του φαινομένου και να χρησιμοποιηθούν όλα αυτά υστερότερα σε μεταγενέστερη φάση για να υιοθετηθεί μια εξειδικευμένη αντιμετώπιση εξειδικευμένων κατηγοριών σε διαφορετικές χώρες εν μέρη καταφέραμε, εν μέρη λέω, μερικώς να υλοποιήσουμε αυτούς τους στόχους μας. Και έτσι έχουμε ομαδοποιήσεις 7 χωρών, ανά χώρες. Και με βάση αυτό η τέταρτη προσέγγιση μεθοδολογικά είναι η case studies, η περίπτωση η ανάλυση περιπτώσεων σε σχέση με την ανάλυση διασυνδέσεων διαφθοράς και οργανωμένου εγκλήματος σε συγκεκριμένες χώρες. Και αυτό μας παρέσχε, μας έδωσε μια σχετικά πλούσια, σύνθετη εικόνα για τους τρόπους με τους οποίους το οργανωμένο έγκλημα στοχοθετεί, στοχοποιεί θεσμικά όργανα και θεσμούς σε διάφορες χώρες και χρησιμοποιεί μεθόδους διαφθοράς ώστε να διαφθαρούν αυτοί οι θεσμοί και, τα, και οι κρατικές υπηρεσίες για να πετύχουν το στόχο τους οι εγκληματίες. Τώρα όλα αυτά για τη διασύνδεση μεταξύ ανάλυσης καταδείχθηκε ότι η διασύνδεση μεταξύ οργανωμένου εγκλήματος και διαφθοράς είναι κάτι το πολύ σύνθετο και περίπλοκο ζήτημα και θα μπορούσε να συνοψιστεί σε τρεις κατηγορίες και παραμέτρους. Επεξηγώντας τώρα πώς η διασύνδεση αυτή εκφράζεται σε μια συγκεκριμένη χώρα και το επίπεδο με το οποίο αυτή η διασύνδεση, αυτός ο συσχετισμός λειτουργεί. Μεταξύ όλων αυτών το πιο σημαντικό είναι οι ιστορικοί παράγοντες πρώτα και κύρια με το οποίο εννοούμε τις εξειδικευμένες ε, ιστορικές ε, διεργασίες που υπέστησαν διάφορα κράτη-μέλη. Μία από αυτές είναι η μεταβατική περίοδος ε, δημοκρατικοποίησης από ολοκληρωτικά καθεστώτα προς την δημοκρατία σε κέντρο-ανατολικό ευρωπαϊκές χώρες που δημιούργησε μεγάλη δραστηριότητα στο φαιό τομέα, στον γκρίζο και μαύρο τομέα με τη μεταφορά της κυριότητας της ιδιοκτησίας επιχειρήσεων σε πολλές από αυτές τις χώρες. Μια άλλη κατάσταση είναι οι εθνικιστικές κινήσεις και κινήματα σε διάφορες χώρες ως κινήματα στη Βόρεια Ιρλανδία, Κορσική, την χώρα των Βάσκων και τα λοιπά. Και μια δεύτερη ομάδα ή κατηγορία παραμέτρων σε σχέση με όλα αυτά είναι αυτό που, που δείχνει ότι χώρες με μεγαλύτερες διαφορές εισοδήματος, κατανομής του εισοδήματος και μεγαλύτερες και εντονότερες διαφορές όσον αφορά τις διαχωριστικές γραμμές που υφίστανται όσον αφορά και την πολιτική ζωή και τη διακυβέρνηση. Εδώ υπάρχει μια συγκεκριμένη τάση να χρησιμοποιείται η διαφθορά και μέθοδοι ε, του οργανωμένου εγκλήματος σε διαφορετικές δραστηριότητες όσον αφορά τις αγορές. Και τώρα κάτι τελευταίο. Αυτά τα πολιτιστικά χαρακτηριστικά στοιχεία χαρακτηρίζουν συγκεκριμένες χώρες στην κατηγοριοποίηση αυτή. Μπορεί σε μεγαλύτερο βάθος να καλυφθεί η πτυχή αυτή της ιδέας του τι εννοούμε με αυτή τη διασύνδεση αν αναφερθείτε στην έκθεση και την μελετήσετε στο αντίστοιχο τμήμα. Το πρώτο εγχείρημα, το πρώτο ζήτημα το οποίο προσπαθήσαμε να αντιμετωπίσουμε στην ανάλυση των στοιχείων είναι η χαρτογράφηση της διαφθοράς, η διασύνδεση μεταξύ διαφθοράς και οργανωμένου εγκλήματος. Τι βρήκαμε. Αυτό που βρήκαμε μελετώντας και συλλέγοντας πληροφορίες για τους δείκτες αυτούς είναι ότι κατά το μάλλον ή τον γνωστό βέβαια από προηγούμενες μελέτες αλλά επιβεβαιώθηκε, επαληθεύθηκε για άλλη μια φορά και πάλι και αυτό είναι ότι υπάρχουν δύο μορφές, δύο τύποι γενικής διασύνδεσης που υφίστανται. Ο πρώτο, το πρώτο είναι το επίπεδο οικονομικής ανάπτυξης, όπως μετράται από τα επίπεδα του ΑΕΠ ανακεφαλήν. Και οι δύο άλλες εναλλακτικές δυνατότητες είναι επίπεδο διαφθοράς και επίπεδο ελέγχου της διαφθοράς όσο ανώτερη είναι η ανάπτυξη τόσο μικρότερη είναι η διαφθορά και πιο εύκολος ο έλεγχος της διαφθοράς. Αυτή είναι η γενική διασύνδεση σε σχέση με το ΑΕΠ και τα θέματα διαφθοράς. Αποδείχθηκε ότι σε σχέση με το μεγαλύτερο βαθμό στατιστικών στοιχείων όσον αφορά τις δραστηριότητες οργανωμένου εγκλήματος και διαφθοράς αφενός είναι η κατηγοριοποίηση των χωρών όσον αφορά την αποτελεσματικότητα των θεσμικών κυβερνητικών οργάνων. Όσο πιο αποτελεσματικά είναι αυτά τα όργανα ή θεσμοί, τόσο είναι χαμηλότερα τα επίπεδα διαφθοράς. Και όσο πιο αποδυναμωμένες είναι αυτές οι ε, δομές, το αντίστροφο. Η δεύτερη διασύνδεση είναι αν ε, η διαφθορά στατιστικά συνδέεται με το οργανωμένο έγκλημα και για το συσχετισμό με άλλα λόγια σε σχέση με τους δείκτες που μετρούν αυτές τις δύο ε, είναι 0,7 η διακύμανση. Τι σημαίνει αυτό. Υπάρχει μια αρκετά ισχυρή σχέση μεταξύ των δύο αυτών παραμέτρων. Το οργανωμένο έγκλημα χρησιμοποιεί τη διαφθορά ως μέσο, ως εργαλείο. Από την άλλη πλευρά, σε ένα περιβάλλον διαφθοράς διευκολύνεται η χρήση του οργανωμένου εγκλήματος και των μεθόδων του. Και το ένα και το άλλο θέτει όρους και προϋποθέσεις με θετικό και αρνητικό τρόπο έναντι του άλλου. Ωστόσο από την άλλη όμως πλευρά ο αριθμός των χωρών, ο αριθμός των διασυνδέσεων, ο αριθμός των συνιστοσών είναι υπερβολικά μεγάλος για μια τέτοια μελέτη και για αποτελέσματα τα οποία θα μπορούσαν να είναι ευδιάκριτα. Γι' αυτό ε, ο επόμενος στόχος μας ως πρόκληση είναι η κατηγοριοποίηση χωρών και η κατάδειξη συγκεκριμένων χαρακτηριστικών στοιχείων ε, όσον αφορά τις χώρες επιλέγοντας μία χώρα ανακατηγορία κάνοντας μία, συντάσσοντας μία μελέτη περίπτωση για αυτήν την χώρα τώρα σε σχέση με την ε, ανάλυση αυτή αυτό το οποίο είδαμε είναι δημιουργήθηκε ένα σύνολο 7 κατηγοριών. Στο αριστερό, στην αριστερή πλευρά αυτών των στοιχείων εδώ μπορείτε να δείτε την πρώτη κατηγοριοποίηση που συμπεριλαμβάνει τις σκανδιναβικές χώρες και που χαρακτηρίζεται με χαρακτηριστικό στοιχείο με υψηλό επίπεδο ελέγχου της διαφθοράς, χαμηλά επίπεδα διαφθοράς, χαμηλά επίπεδα οργανωμένου εγκλήματος σε αυτές τις χώρες. Στην κάτω δεξιά πλευρά αυτών θα δείτε χαμηλά επίπεδα χαμηλό επίπεδο ελέγχου διαφθοράς, υψηλά επίπεδα διαφθοράς και υψηλά επίπεδα οργανωμένου εγκλήματος. Και στο ενδιάμεσο, στο μεσοδιάστημα εκεί υπάρχουν οι άλλες κατηγορίες όπου είχαμε δύο συγκεκριμένες περιπτώσεις. Η μία ήταν η περίπτωση της Γαλλίας. Η δεύτερη ήταν η περίπτωση της Ιταλίας που δεν μπορούσε να ομαδοποιηθεί, να κατηγοριοποιηθεί με άλλες χώρες λόγω των ειδικών χαρακτηριστικών αυτής της χώρας και της άλλης. Και οι δύο χώρες έχουν υψηλά επίπεδα ΑΕΠ. Όμως στη Γαλλία υπάρχει καλύτερος έλεγχος της διαφθοράς, καλύτερη αντιμετώπιση. Σε αντίθεση στην Ιταλία υπάρχει χαμηλότερο επίπεδο ελέγχου της διαφθοράς και υψηλά επίπεδα οργανωμένου εγκλήματος. Τώρα, με βάση με βάση αυτές τις κατηγοριοποιήσεις, τι γίνεται. Μια χώρα, ουσιαστικά είχαμε έξι μελέτες για έξι χώρες. Μία χώρα ανά κάθε κατηγορία και μία συγκεκριμένη μελέτη που έγινε ειδικά για να δειχθεί η επίπτωση, το βάθος της συγκεκριμένης κατάστασης όσον αφορά αυτή την συγκεκριμένη κατηγοριοποίηση για τη διασύνδεση οργανωμένου εγκλήματος και διαφθοράς φυσικά. Και θα ήθελα εδώ να δώσω τον λόγο στον συνάδελφο. Παρακαλώ, έχετε τον λόγο. Uh, Ευχαριστώ. Πριν συνεχίσω για να ολοκληρώσω τα όσα παρουσίασε ο Άλεξ, να πω ότι αυτές οι ομάδες κρατών, κλάστερς που αναπτύξαμε, χρειάζονται μία προειδοποίηση. Θεωρούμε ότι τα δεδομένα όπου βασιστήκαμε είναι σχετικά αναξιόπιστα οι διάφοροι δείκτες ε, της ε, διεθνούς διαφάνειας ε, και διαφόρων μελετών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής συνήθως παρακολουθούν την άποψη του κοινού και τις εμπειρίες του κοινού όσον αφορά την διαφθορά. Δεν υπάρχουν αξιόπιστοι δείκτες που να αντικατοπτρίζουν σωστά τα υψηλά επίπεδα σχέσης ε, διαφθοράς στο οργανωμένο έγκλημα αλλά και δείκτες ε, για θέματα όπως ε, η ισχύ του οργανωμένου εγκλήματος και το μέγεθος της διαφθοράς. Άρα δημιουργήσαμε μεν αυτά τα κλάστερα, αυτές τις ομάδες, αλλά στη συνέχεια προσπαθήσαμε να βρούμε επεξηγήσεις και όχι να κάνουμε μια απλή ιεράρχηση των χωρών. Στην έκθεση βλέπετε ότι προσφέρουμε τρεις προσεγγίσεις ανάλυσης του πότε και πώς χρησιμοποιεί το οργανωμένο έγκλημα τη διαφθορά. Καθαρά, καταρχάς εξετάζουμε το ποια όργανα είναι αυτά που γίνονται στόχοι και για ποιους λόγους και πότε. Δεύτερη προσέγγιση, παίρνουμε μία παράνομη αγορά και την εξετάζουμε. Για παράδειγμα, διανομή ναρκωτικών, διακίνηση ναρκωτικών πότε χρειάζεται η διαφορθώρα εκεί και πόσο χρησιμοποιείται σε διάφορες χώρες. Τώρα, περνάω σε μια σύντομη περιγραφή του πώς στοχεύονται συγκεκριμένα θεσμικά όργανα. Διαπιστώσαμε ότι η δικαστική οι υπηρεσίες, η αστυνομία και τα τελωνία είναι οι πιο στοχοποιημένοι θεσμοί. Βεβαίως ανάλογα με την εγκληματική δραστηριότητα και άλλοι οργανισμοί μπορούν να γίνουν στόχοι. Για παράδειγμα, αν μιλάμε για παράνομα πολιτιστικά προϊόντα, οι εργαζόμενοι σε μουσεία αν μιλάμε για παράνομη υλοτόμηση, μπορεί να μιλάμε για τους υποαλλήλους των δασικών υπηρεσιών. Αλλά στην μελέτη μας επικεντρωθήκαμε στους πιο συχνά στοχοποιημένους θεσμούς και οργανισμούς. Και εκεί εξετάσαμε τα θέματα που θεωρήσαμε πιο σημαντικά. Ξεκινάμε με την αστυνομία. για να επιστρέψω λίγο. Το σημαντικό είναι να διαπιστώνουμε πώς διασυνδέονται οι διάφορες διαφθορές. Όταν μιλάμε για πολιτική διαφθορά, ένας διαφθαρμένος πολιτικός μπορεί να έχει επιρροή και σε άλλους θεσμούς, άλλα θεσμικά όργανα. Δεν μπορούν δηλαδή να γίνουν διαχωρισμοί σε μια χώρα μπορεί να υπάρχει για παράδειγμα επίσης αστυνομική διαφθορά αλλά οι αστυνομικοί να προσπαθούν να επηρεάσουν τους δικαστές και τα λοιπά. Και ενδεχομένως κάπου να εμπλέκεται και κάποιος διεφθαρμένος πολιτικός που προσπαθεί να ασκήσει επιρροή. Υπάρχουν λοιπόν πολύ διαφορετικοί παράγοντες. Τώρα, πώς χρησιμοποιεί το οργανωμένο έγκλημα τη διαφθορά για να στοχοποιήσει θεσμικά όργανα. Ένα παράδειγμα. Οι κοινωνικές πολιτιστικές ε, επαφές σε μία χώρα μπορεί να διευκολύνουν σημαντικά την πρόσβαση στην αστυνομία μιας χώρα. αν υπάρχει γενικά πιο άτυπη συμπεριφορά. Σε ορισμένες χώρες όμως όπου υπάρχουν πιο τυπικές ε, σχέσεις στην αστυνομία αποθαρρύνονται οι άτυπες κοινωνικές σχέσεις και είναι πιο δύσκολο να υπάρξει διαφθορά είχαμε την εντύπωση ότι στις πρώτες περιπτώσεις η διαφθορά μπορεί να είναι πολύ μεγαλύτερη. Βεβαίως μπορεί να λειτουργήσει και ως μηχανισμός ε, πρόληψης. Σε χώρες ε, όμως που δεν υπάρχουν τέτοιες μονάδες στην αστυνομία ή τα τελωνία, επιφανειακά δεν βλέπουμε τόσο μεγάλη διαφθορά, αλλά η αλήθεια είναι ότι δεν ξέρουμε τι συμβαίνει στην πράξη. Η αστυνομία είναι γενικά ο πρώτος στόχος του οργανωμένου εγκλήματος. Παντού ουσιαστικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση είδαμε στοχοποίηση της αστυνομίας ακόμη και σε χώρες όπου δεν θεωρείται σημαντικό πρόβλημα η διαφθορά. Είναι και το θέμα το οποίο συζητείται το περισσότερο. Είχαμε πολλές συνεντεύξεις στο Ηνωμένο Βασίλειο όπου μια σοβαρή υπηρεσία για το οργανωμένο έγκλημα που αναλύει τα στοιχεία για τη διαφθορά μας είπαν ότι έχουν αποφασίσει να μην δημοσιοποιούν τα στοιχεία τους, να μην δημοσιοποιούν τις αιτήσιες εκθέσεις τους για να μην μειωθεί η εμπιστοσύνη του κοινού στην αστυνομία. Επίσης, να πω ότι παρόλο που πρόκειται για ένα κοινό θέμα στις χώρες μας. Το επίπεδο στο οποίο υπάρχει επιρροή του οργανωμένου εγκλήματος στην αστυνομία διαφέρει. Σε ορισμένες χώρες ε, ολόκληρα τμήματα της αστυνομίας είναι διαφθαρμένα, ολόκληρες ε, μονάδες. Ενώ σε άλλες ε, χώρες έχουμε συγκεκριμένες υποθέσεις με μεμονωμένους αξιωματούχους συχνά κοντά στη συνταξιοδότηση που γίνονται στόχοι. Βεβαίω, ανάλογα με τη χώρα διαφέρει πολύ και η πίεση προς τις αστυνομικές αρχές. Σε χώρες όπου η πορνεία ή τα ναρκωτικά είναι παράνομα, μπορεί να είναι πολύ αυξημένη η πίεση προς τους ε, αστυνομικούς τους χαμηλόβδαθμους. Ενώ σε χώρες όπου είναι νόμιμη η πορνεία μπορεί να είναι μικρότερη η διαφθορά σε αυτό το επίπεδο. Επίσης ένα άλλο θέμα είναι ότι διαπιστώσαμε ότι σε πολλές χώρες τα τοπικά εγκληματικά δίκτυα έχουν διασυνδέσεις και με μετανάστες εγκληματίες, δίκτυα μεταναστών. Αυτό το διαπιστώσαμε και στην Βόρεια Ιρλανδία αλλά και στην Γαλλία, στη Μασαλία όπου είδαμε τους μουσούς να λειτουργούν ως ενδιάμεση για την ε, διαφθορά των τοπικών αστυνομικών. Κάτι άλλο που πρέπει να συζητήσουμε είναι η πολιτική διαφθορά. Σίγουρα η πολιτική δεν είναι τόσο συχνά διεφθαρμένοι όσο οι αστυνομικοί, όμως οι συνέπειες της πολιτικής διαφθοράς μπορεί να είναι πολύ μεγάλες. Γιατί μπορούν για παράδειγμα να ασκήσουν επιρροή στις δικαστικές υπηρεσίες στα τελωνία και αλλού. Με βάση την ανάλυση μας προκύπτει σαφής διάκριση μεταξύ των τοπικών πολιτικών και της τοπικής διαφθοράς όπου Πρόκειται για φαινόμενο που εμφανίζεται σχεδόν παντού στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ οι περιπτώσεις υψηλής διαφθοράς βουλευτών, υψηλών κυβερνητικών αξιωματούχων, εκεί οι περιπτώσεις ήταν πολύ περιορισμένες και σχεδόν απούσες. Επίσης είχαμε μεγάλη δυσκολία να βρούμε πληροφορίες για αυτά τα θέματα. Κάτι που διαπιστώσαμε και είναι ενδιαφέρον είναι ότι παντού στην Ευρωπαϊκή Ένωση όταν αλλάζει η κυβέρνηση, η νέα κυβέρνηση εξετάζει πολύ την πολιτική διαφθορά του προηγούμενου καθεστώτος και όσο πιο συχνά υπάρχουν κυβερνητικές αλλαγές τόσο πιο συχνές είναι και αυτές οι έρευνες και υπάρχουν και μάλιστα κάποιες συγκεκριμένες χρονικοί περίοδοι που είναι ιδιαίτερα συνδεδεμένοι με αυξημένη διαφθορά. Και αυτό φαίνεται και στις δημοσκοπήσεις, άρα όταν βλέπουμε αυξημένη ανησυχία του κοινού για τη διαφθορά μπορεί αυτό να οφείλεται στην αυξημένη δραστηριότητα μιας νέας κυβέρνησης κατά της προηγούμενης. Όσον αφορά τώρα τη διαφθορά στον ιδιωτικό τομέα, πολύ σύντομα. Όταν μιλάμε για τις ε, ιδιωτικές εταιρείες τις οποίες στοχεύει το οργανωμένο έγκλημα, δεν μιλάμε για δωροδοκίες αξιωματούχων. Αυτό στο οποίο επικεντρωθήκαμε ήταν εγκληματικές ομάδες ή επιχειρήσεις που σχετίζονται με παράνομες δραστηριότητες και οι οποίες ε, στοχεύουν σε... στην αστυνομία ή άλλους φορείς. Αν δείτε εδώ την εικόνα βλέπετε ότι για παράδειγμα όταν έχουμε το λαθρεμπόριο τσιγάρων μπορεί να χρησιμοποιηθούν τα εργοστάσια τσιγάρων για να μεθοδεύσουν τη διακίνηση των παράνομων τσιγάρων ή κάτι αντίστοιχο μπορεί να γίνει και με τους εργαζόμενους στα μουσεία Πολύ ευάλωτες εδώ μπορεί να είναι οι μεταφορικές εταιρείες και το προσωπικό τους. Επίσης οι εταιρείες ασφάλειας και το προσωπικό ασφαλείας. Και επίσης διαπιστώσαμε και περιπτώσεις όπου για παράδειγμα οι ιδιοκτήτες σούπερ μάρκετ δωροδοκούνται για να διακινούν λαθρέα τσιγάρα. Κάτι που βλέπουμε με τη διαφθορά στον ιδιωτικό τομέα είναι ότι παρόλο που υπάρχει απόφαση του Συμβουλίου για την διαφθορά στον ιδιωτικό τομέα, εξακολουθεί να μην έχει εφαρμοστεί σε αρκετές χώρες. Σε πολλές χώρες η διαφθορά στον ιδιωτικό τομέα είτε δεν θεωρείται έγκλημα, δεν είναι ποινικοποιημένοι, είτε δεν υπάρχουν υπεύθυνοι για αυτήν, δεν υπάρχουν διατάξεις για αυτή. Σε πολλές χώρες δεν γνωρίζαμε καν σε ποιον να απευθυνθούμε. Υπάρχουν μόνο κάποιες ελάχιστες έρευνες σχετικά. Θα πηδήξω τα υπόλοιπα και θα δώσω το λόγο στο συνάδελφο για να περάσει στις τελικές συστάσεις της έρευνας. Ευχαριστώ. Και με τρία λεπτά για την... να ολοκληρώσουμε. Έχουμε δύο ομάδες συστάσεων που όπως ζητήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζητήθηκε να αναπτυχθούν υπό το φως του προγράμματος της Στοκχόλμης και της υλοποίησης του προγράμματος της Χάγης και της υλοποίηση της συνθήκης της Λισαβόνας. Δύο ομάδες συστάσεων. Η πρώτη, η πιο φιλόδοξη, αλλά και εναλλακτική λύση με μεγαλύτερη πρόσθετη αξία που παρουσιάζω. Να υπάρξει ένας μηχανισμός που θα εκπονηθεί για την επιτήρηση, την εποπτεία της διαφθοράς, για να αναβαθμιστεί ή να, βελτιωθεί, να βελτιωθούν οι μηχανισμοί που χρησιμοποιούνται στο επίπεδο ΩΣΑ, Συμβουλίου της Ευρώπης, Europol, όκτα ε, στοιχείων των Ηνωμένων Εθνών και της ε, ε Σύμβασης ε, κατά της θεωρούμε ότι θα μπορούσαν να είναι πρόσθετης αξίας αυτά τα μέτρα ώστε να υπάρξει μια μονάδα συλλογής στοιχείων και πληροφοριών όπως για τα, ε, τον οργανισμό των, για τα, ε, τα πολιτικά δικαιώματα ή το παρατηρητήριο κατά της, ε, του ρατσισμού και της ξενοφοβίας που θα επιτρέπει μια ανεξάρτητη εικόνα και επισκόπηση τοπικά αναχώρα των σημείων αυτών διότι η διασύνδεση μεταξύ διαφθοράς και οργανωμένου εγκλήματος συνδέεται άρρηκτα με την τοπική κατάσταση, επιτόπου, την επιτόπου κατάσταση, αλλά και να μπορούμε να μοιραζόμαστε αυτές τις, αυτά σε ευρωπαϊκό επίπεδο χρειάζεται, πιστεύουμε, ένα, ένας μηχανισμός benchmarking indicators, βελτιστοποιημένων δικτών σε ένα μηχανισμό για αυτές τις ενδείξεις. Και θεωρούμε ότι όχι μόνο θα πρέπει να συλλέγουμε στοιχεία από τις ομάδες καταπολέμησης διαφθοράς, από τις αστυνομικές ε, δυνάμεις, ε, για παράδειγμα, αλλά και αντίστροφα να έχουμε ε, σε σχέση με τους παραβάτες και τον ιδιωτικό τομέα συλλογή πληροφοριών. Έτσι λοιπόν ένας τέτοιος μηχανισμός θα μπορούσε να είναι μια ανεξάρτητη νέα υπηρεσία που θα λογοδοτεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αλλά πρέπει να υπάρξει μια πολύ πιο στεναρή, πιο σοβαρή μελέτη για τις επιπτώσεις και τον χαρακτήρα αυτού του θεσμού. Ένα δεύτερο, μη όχι τόσο φιλόδοξο επίπεδο είναι να χρησιμοποιηθεί το άρθρο της Συνθήκης Λισαβόνας που ζητεί την εκπόνηση ελάχιστων κανονισμών ή κανόνων και με βάση αυτούς να οικοδομήσουμε ένα οικοδόμημα. Θα μπορούσε να είναι μια καλή βάση για την, τον κοινό ορισμό από τα κράτη-μέλη αυτών των στοιχείων από πλευρά αστυνομικών δυνάμεων ή τελωνίων. Αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε εναρμονισμένα στατιστικά στοιχεία για το πώς θα μπορούσαν να δημιουργηθούν προγράμματα κατά της διαφθοράς από πλευρά Ευρώπη. Ένωση ε, κατά τη εκπαίδευση, Ένα από τα πράγματα που διαπιστώσαμε ότι απουσιάζει και λείπει είναι τα προγράμματα επιμόρφωσης και κατάρτισης ε, για τη διαφθορά και το οργανωμένο έγκλημα είναι θεωρητικού χαρακτήρα, γενικόλογου χαρακτήρα. Πολύ λίγα πρακτικά πράγματα ή περιπτώσεις ε, πρακτικές καθημερινής καταπολέμησης εξετάζονται και αυτό θα μπορούσε να εμπλουτιστεί. Σας ευχαριστώ. Thank you for that σε ευχαριστούμε και έχουμε ακόμα στενό χρονικό πλαίσιο όσον αφορά ερωτήσεις. Θα το εκτιμούσα αν είσαστε σύντομοι στα σχόλια ή παρατηρήσεις σας για να μπορέσουμε έγκαιρα να ολοκληρώσουμε. Ο κύριος Ντε Γιόγκ πρώτος. Έχετε τον λόγο παρακαλώ. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ επίσης θερμά τους ερευνητές για το έργο που επετέλεσαν. Θα ήθελα όμως κάποιες ε, κριτικές ε, παρατηρήσεις να κάνω. Οι ίδιοι οι ερευνητές ε, δεν μπορούν οι ίδιοι να πούν πολλά, αλλά θα πρέπει να το σημειώσουμε αυτό όμως παρόλα αυτά. Η μεθοδολογική προσέγγιση αυτής της ανάλυσης θεωρώ ότι είναι αμφισβητήσιμη. Αν δούμε εδώ ένα γράφημα ή μια απεικόνηση όπου τα κράτη-μέλη τα οποία επελέγησαν κατηγοριοποιημένα αναφέρονται για το μέτρο, το ύψος της διαφθοράς και των ελέγχων, δημιουργεί αυτό καταρχήν την εντύπωση, ίσως με μια πρώτη ματιά, ότι αυτό θα μπορούσε να ήταν αξιόπιστο. Αλλά αυτό δεν επιχειρηματολογείται σοβαρά, δεν μπορεί κάτι τέτοιο να γίνει σοβαρά δεκτό. Ε, υπάρχουν κάποια στοιχεία, κάποιοι δείκτες στα οποία βασίζονται αυτά, αλλά δεν είναι όμως αξιόπιστο αντικειμενικό υλικό. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή αξιόπιστο αντικειμενικό υλικό για τη μέτρηση της διαφθοράς. Δεν υπάρχει αντικειμενικό μέσο ή εργαλείο για τη μέτρηση του οργανωμένου εγκλήματος και ούτε υπό το πρίσμα της αποτελεσματικότητας των ελέγχων, ελέγχων για την καταπολέμηση της διαφθοράς. Ο αριθμός των καταδικών δεν λέει πολλά πράγματα. Αυτό μπορεί να σημαίνει σε μια χώρα υπάρχει εξαιρετικός έλεγχος της διαφθοράς, ε, τότε ο αριθμός ε, των περιπτώσεων α, καταδικών το, της διαφθοράς δεν είναι κάτι το αξιόπιστο για το βαθμό της διαφθοράς. Αυτό μπορεί να σημαίνει ότι τα πράγματα βαίνουν καλώς. Ενώ σε ένα άλλο κράτος μπορεί να υπάρχουν λίγες καταδίκες, αλλά αυτό δεν μπορεί να σημαίνει υποχρεωτικά ότι ε, οι έλεγχοι δεν λειτουργούν. Λοιπόν, αυτά πρέπει να τα λάβουμε υπόψη. Θέλω να πω δύο λόγια για τη μελέτη, για την έρευνα. Είναι ενδιαφέρον να δούμε τη διασύνδεση διαφθοράς και οργανωμένων αντικείμενο εγκλήματος. Πιστεύω όμως από την άλλη πλευρά ότι εμείς στο τέλος τέλος δεν θα πρέπει να διαφοροποιούμαστε μεταξύ μεγάλων και μικρών περιπτώσεων διαφθοράς. Αν κάποιος για παράδειγμα πρέπει να πληρώνει ένα ποσό, να λαδώνει για να έχει πρόσβαση στην εκπαίδευση, στην παιδεία ή στην υγεία, ε, τότε αυτό είναι κάτι διαφορετικό από ότι αν συμβαίνει αυτό σε, ένα, σε μια τεράστια κλίμακα διαφθοράς. Εδώ πρόκειται όμως για κάθε μορφή διαφθοράς και όμως για κάποιες, και όχι για κάποιες λίγες, ε, για κάποιους λίγους τύπους διαφθοράς. Τώρα, σε σχέση με τις επιλογές, πιστεύω ότι το, ο κατεπήγων χαρακτήρας, διότι και στη δική μας Κοινοβουλευτική Επιτροπή και στο Ευρωκοινοβούλιο πρέπει να δούμε και να ε, παρακολουθήσουμε το τι γίνεται για την καταπολέμηση της διαφθοράς και του οργανωμένου εγκλήματος. Αυτό όμω δεν επαρκεί. Εκπονεί μια ανακοίνωση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πάνε όμως ε, πολύ αργά οι ρυθμοί και τα πράγματα από πλευρά της. Πρέπει να ασκηθεί μεγαλύτερη πίεση να επιταχυνθούν οι ρυθμοί. Τώρα τι μπορεί να γίνει. Θα έλεγα πραγματικά θα πρέπει να το καταφέρουμε και αυτό ισχύει για την Ευρωπαϊκή Ένωση και για τα κράτη-μέλη και που ε, για την καταπολέμηση της ε, διαφθοράς έχουν ε, υπογράψει και τη σύμβαση, τη συνθήκη ουσιαστικά, ένα καλό σύστημα εποπτείας χρειάζεται. Και για νέες πρωτοβουλίες που πρέπει να αναλυφθούν. Υπάρχουν παραδείγματα σε παγκόσμια κλίμακα, στη Λατινική Αμερική. Υπάρχουν καλύτερα μέσα μέτρησης ώστε να μπορεί κανείς να μετρά αυτά τα θέματα πιο αποτελεσματικά. Δεν δημιουργείται, δεν ερωτάτε για την εντύπωση που δημιουργεί διαφθορά, δηλαδή ε, perception, πώς, ποια είναι η απήχηση, αλλά τι πλήρωσε κανείς ε, παραπάνω και υπερβολικά στις αρχές για λαδώματα. Και υπάρχουν ίσως και πιο δημιουργικές δυνατότητες να μετρηθεί η διαφθορά και το επίπεδό της μέσα στο πλαίσιο των μηχανισμών εποπτείας. Για τη δημιουργία μιας τέτοιας υπηρεσίας να μην ξεχνάμε ότι και οι υπηρεσίες και οι οργανισμοί μπορούν να ε, διαφθαρούν και να είναι διεφθαρμένοι ή διεφθαρμένα. Και γι' αυτό πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι και εδώ και στην Επιτροπή και στην αντιπροσωπεία της Επιτροπής και σε άλλες χώρες μπορεί να υπάρχει κάποιο ποσοστό διαφθοράς. Πρέπει και οι ίδιοι να αυτοεπιτηρούμεθα. Κατά άλλα είναι καλό ότι δίνουμε προσοχή σε αυτό το θέμα. Έχουμε πολλά όμως να κάνουμε και ελπίζω θα έχουμε μια θετική συνέχεια στη συζήτηση όσον αφορά την εποπτεία που είμαστε υποχρεωμένοι να διασφαλίσουμε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε λίγο διαφορετική η άποψή μου. Θεωρώ ότι τα ευρήματα αυτής της έρευνας, το περιεχόμενο της παρουσίασης ε, και της έκθεσης είναι ιδιαίτερα υποσχόμενα. Για διάφορους λόγους. Καταρχάς, δεν μιλάμε για κάτι που είναι εύκολο να μετρηθεί, να παρακολουθηθεί. Πρόκειται για το πιο πολύπλοκο και κρυφό κομμάτι της ζωής μιας κοινωνίας ε, ή μιας κοινότητας. Άρα πρέπει να είμαστε γενναίοι και με ενθουσιασμό να μπούμε σε αυτό το σκιώδες κομμάτι της κοινωνίας. Βεβαίως ε, μια επικριτική στάση είναι απαραίτητη γιατί μιλάμε για ένα φαινόμενο που θα παραμείνει μαζί μας για πολύ χρόνο. Και εδώ εντάσσεται και η ερώτησή μου. Μιλώντας ε, για τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά διαφθοράς και οργανωμένου εγκλήματος ε, σε διάφορα σημεία της Ευρώπης και του κόσμου, προφανώς ε, οι συγγραφείς της έκθεσης έλαβαν υπόψη και την κοινωνική δομή σε ορισμένες κοινότητες της Ένωσης, ε, τις ε, φατρίες, τις πατριές που υπάρχουν, ε, τη δύναμη της οικογένειας αν θέλετε και αναρωτιέμαι αν τέτοιου είδους περιστάσεις μπορεί να αυξήσουν ακόμη περισσότερο τη μεταβατική περίοδο. Και επίσης αναρωτιέμαι μήπως τα επόμενα χρόνια θα πρέπει να αφιερώσουμε ακόμη περισσότερη προσπάθεια και πόρους προκειμένου να αποφύγουμε την εγκατάσταση του οργανωμένου εγκλήματος σε ορισμένες χώρες που είχαν ολοκληρωτικό καθεστώς στο παρελθόν. Σε ορισμένες περιπτώσεις η έκθεσή σας κάνει πολύ καλή δουλειά και το εκτιμώ αυτό γιατί Συχνά βλέπουμε στον τύπο απλές ιστορίες για δωροδοκία και νεποτισμό, ενώ η δική σας έκθεση νομίζω ότι ήταν πολύ πιο φιλόδοξη. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κυρία Ελετσέβα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους τρεις εμπειρογνώμονες για την σωστή και εύστοχη παρουσίαση που κάνανε. Είναι πολύ πολύπλοκα όλα αυτά τα κείμενα και τους ευχαριστώ που μας διαφώτισαν για όλα αυτά τα δύσκολα θέματα. Εγώ θέλω να συγκεντρωθώ σε τρία βασικά θέματα ένα το οποίο αφορά στη Βουλγαρία και στη Ρουμανία και ένα το οποίο αφορά στις προπτικές γενικότερα. Εσείς είπατε ότι ήδη υπάρχουν άλλοι μηχανισμοί αξιολόγησης από ότι το Ευρωμαρόμετρο ε, ή την Ευρωπόλ ή την Ευρωπαϊκή Οργάνωση για τη Συνεργασία και την Ανάπτυξη. Ρωτάω λοιπόν ποια είναι η προστιθέμενη αξία του μηχανισμού που εσείς προτείνετε έναντι των υπαρχόντων μηχανισμών. Δεύτερο, αφορά στην προστιθέμενη αξία που προτείνει ο μηχανισμός της μελέτης σας. Τι, θέλετε εσείς να συνεισφέρετε με τη μέθοδό σας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στους μηχανισμούς της ε, και αναφέρομαι εδώ στη διεύρυνση πιο συγκεκριμένα και πώς μπορείτε να βοηθήσετε τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία. Τρίτο τώρα για την Κομισιόν. Η Κομισιόν λέει εφαρμογή του προγράμματος της Στοκχόλμης και θέλει μία ανακοίνωση για την ε, καταπολέμηση της διαφθοράς στα κράτη-μέλη και προβλέπει και ένα μηχανισμό αξιολόγησης όπως επίσης και συνεργασία στα πλαίσια του Συμβουλίου της Ευρώπης με τις διάφορες χώρες. Ρωτώ λοιπόν, τι σκέφτεσαι εσείς για έναν τέτοιον μηχανισμό αξιολόγησης για την ε, διαφθορά ή την αντιδιαφθορά, δείτε εσείς ποιος είναι ο καλύτερος όρος, ο κάθε μηχανισμός είναι δύσκολος να στηθεί από τεχνικής πλευράς και για την πρόσβαση και για την πληροφόρηση. Παρακαλώ λοιπόν να μου πείτε τι λέτε εσείς σχετικά. Έχετε κάποια ιδέα για το ποια είναι η πρόκληση, ποια είναι τα εμπόδια που έχουμε να αντιμετωπίσουμε, αλλά και επίσης τα πλεονεκτήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης από αυτούς τους μηχανισμούς. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Εγώ θέλω να ευχαριστήσω τους εισηγητές ε, για τη μελέτη που μας ε, θέτει πολύ ενδιαφέρουσες εχμές. Ίσως ε, θα έπρεπε να αποφύγουμε να κάνουμε εμείς έναν έλεγχο, βαθμολογικό έλεγχο των ε, διαφόρων χωρών λέγοντας ποιοι είναι οι καλοί μαθητές ή κακοί μαθητές γιατί τα στοιχεία που έχουμε είναι ανεπαρκή. Μόνο τάσεις μπορούν να μας δείξουν Ευθύνη λοιπόν της Κομισιόν μαζί με το Συμβούλιο και με τα κράτη-μέλη να ξεκινήσουν μια πραγματική στρατηγική έτσι όπως προβλέπεται στο πρόγραμμα της Στοκχόλμης που θα ορίζει και έναν ε, ορισμό συμφωνημένο για το τι εστί διαφθορά διότι είναι δύσκολο εμείς ε, να φτιάξουμε στατιστικές άμα δεν έχουμε τους ίδιους ορισμούς ή να φτιάξουμε τους ίδιους νόμους. Για την κατασταλτική πολιτική επίσης ε, θα πρέπει να βάλουμε σε δίκτυο τα διαθέσιμα στοιχεία, τα επίσημα στοιχεία των κρατών μελών της Ευρωπόλ όλων των ενδιαφερομένων οργανισμών και να δημιουργήσουμε μία πλατφόρμα η οποία ε, ε, νομοθετική πλατφόρμα η οποία θα μπορούσε να είναι κοινή για όλα τα κράτη-μέλη. Σίγουρα αυτή η μελέτη είναι χρήσιμη, αλλά χρειαζόμαστε μία πιο θεσμική τοποθέτηση, με πιο βέβαιες βάσεις. Ο κύριος Μπουσουτήλ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Και εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω τον φιλοξενούμενο μας, τους φιλοξενούμενους μας για την παρουσίαση αυτής της μελέτης που είναι πολύ ενδιαφέρουσα. Σε πολύ καλή χρονική στιγμή υποβάλλεται. Κάποιες εβδομάδες πριν, Πρόεδρε, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε μια γραπτή διακήρυξη για την διαφθορά, για την καταπολέμηση της διαφθοράς. Και θα έλεγα αυτό είναι ένα πρώτο βήμα σε μια ολόκληρη σειρά και αλυσίδα βημάτων που αυτό το Ευρωκοινοβούλιο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να αναλάβουν, να προαγάγουν, ώστε να υπάρξει θέσπιση προτεραιοτήτων στην θέσπιση προτεραιοτήτων για την καταπολέμηση της διαφθοράς. Είναι ένα θέμα όπου δυστυχώς η Ευρωπαϊκή Ένωση λίγα φαίνεται να έκανε μέχρι σήμερα. Και όμως όλοι γνωρίζουμε ότι αυτό το ζήτημα αξίζει πραγματικά να δουλέψει κανείς για να πετύχει καρπούς. Υπό αυτό το πρίσμα θα ήθελα να ακούσω την αντίδραση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για αυτή την έκθεση και υπό το φως των δεσμεύσεων που η κυρία Επίτροπος Μάλμστρομ έχει αναλάβει για τις πρωτοβουλίες που θα ήθελε να αναλάβει σε αυτό το επίπεδο. Θα ήθελα επίσης να υπογραμμίσω ότι Σίγουρα πιστεύω ότι ένας μηχανισμός ο οποίος μας δίνει μια εικόνα και ιδέα για το ποιες χώρες είναι ενάρετες και ποιες είναι αμαρτωλές είναι σημαντικό στοιχείο να το έχουμε. Και εδώ διαφωνώ ελαφρά από αυτά τα οποία ανέφερε ο η προλαλή σας. Συμφωνώ όμως σίγουρα μαζί της ότι αν θέλουμε να έχουμε αυτόν τον πίνακα επιδόσεων αυτός πρέπει να βασίζεται όχι σε οικοτολογίες, οικασίες ή κάποιες διαισθήσεις, αλλά σε σαφή αντικειμενικά στοιχεία και αποδείξεις που καθορίστηκαν σε σχέση με την καταπολέμηση της διαφθοράς. Και αυτό σίγουρα είναι πολύ δύσκολο να θεσπιστεί όπως ακούσαμε, να μετρηθεί. Αλλά αυτή είναι η πορεία που πρέπει να ακολουθήσουμε για να φτάσουμε στο στόχο. Αν θέλουμε να επικεντρωθούμε σε αυτό το στόχο, το να κατονομάσουμε και να καταγγείλουμε και να κατηγορήσουμε είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό τμήμα αυτού του παιχνίδιου, αυτής της αλληλουχίας. Καμιά χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν θα θέλει να είναι κάτω-κάτω στις επιδόσεις όσον αφορά την καταπολέμηση της διαφθοράς. Ευχαριστώ. Mr. Crocetta, signore... Σε ευχαριστώ. Κοτσέτα. Crocetta. Io trovo sinceramente interessante il, questo Βρίσκω ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα αυτή τη μελέτη της Κομισιόν και μάλιστα θα λέγω ότι μέχρι και θαραλέα τη βρίσκω. Διότι σε αυτήν την μελέτη έχουμε πλέον το κουράγιο να δίνουμε αναλυτικά στοιχεία για τομείς που είναι μέχρι και ταμπού. Δηλαδή αστυνομία, σχέσεις με την πολιτική. Έχουμε την ε, μελέτη η οποία αναφέρει παραδείγματα ας πούμε, για την Ιταλία, για την Ισπανία ή τις ανατολικές χώρες. Έχουμε λοιπόν μία χαρτογράφηση η οποία είναι πραγματική, πραγματικά δραματική. δεν έχουμε μπροστά μας κάποια κατάσταση ήρεμη ας πούμε, που τη συζητάμε λέγοντας εντάξει πώς πήγε το, το παγκόσμιο κύπελο. Έχουμε χώρες με αρχαιότατο πολιτισμό και όπου το σύστημα διαφοράς έχει διακλαδωθεί βαθύτατα. Κύριε Μπουσουτήλ, εγώ εκτιμώ ιδιαίτερα που ζητήσατε να γίνει παρουσίαση αυτής της μελέτης. Είναι σίγουρο να πολύ θετικό να το παρουσιάζουμε, αλλά δεν μπορούμε εμείς να φανταζόμαστε ότι αυτά τα φαινόμενα είναι απόλυτα απομονωμένα και μπορεί η προσέγγιση που έχουμε εμείς ε, απέναντι σε αυτή την έκθεση πρέπει να είναι η προσέγγιση ενός εισαγγελέα ή ενός αστυνομικού ε, δηλαδή όπου εξετάζονται μεμονωμένες περιπτώσεις. Όταν εμείς διαπιστώνουμε ότι υπάρχουν ολόκληρες περιφέρειες όπου υπάρχει μία διακλαδωμένη οργάνωση και διασύνδεση μεταξύ ε, πολιτικών αρχών ε, εξουσίας και οργανωμένου εγκλήματος. Τα πράγματα λοιπόν είναι πολύ διαφορετικά. Πρέπει να μιλάμε πλέον για δίκτυα και όταν μιλάμε για την Ιταλία, μιλάμε για την περίπτωση Μπερλουσκόνη για την περίπτωση Κέρμης Στην Ιταλία όμως ξέρετε άμα κανείς πει αυτά τα πράγματα τον φωνάζουν κομμουνιστή. Ενώ εδώ από τις μελέτες τελικά φαίνεται ότι αυτά τα πράγματα δεν είναι επικίνδυνες δηλώσεις επικινδύνων κομμουνιστών που υποσκάπτουν το σύστημα αλλά ότι έχουμε πλέον μία καταφανή κατάσταση καταχρήσεων. Τι να κάνουμε λοιπόν, εμείς κάναμε μία ακτινογράφηση του συστήματος διαφθοράς. Εγώ την, ε, θεωρώ την έκθεση αυτή να υποτιμάει τη διαφθορά και το έγκλημα. Αυτή ίσως είναι η αδυναμία της, διότι οι μελέτες πρέπει να εμβαθύνονται. Αν εμείς ε, πραγματικά εμβαθύνουμε σε αυτή τη μελέτη, τότε θα δούμε τη σχέση οργανωμένου εγκλήματος, διακίνησης όπλων, σχέσεις μεταξύ μαφίας και διεθνούς τρομοκρατίας. <coughs> Θα ανακαλύψουμε το ρόλο των μυστικών υπηρεσιών ε, σε ορισμένες χώρες θα, ανακαλύψουμε το πώς δολοφονούνται οι διάφοροι ε, δημοσιογράφοι στις, ε, στις ανατολικές χώρες, μπορεί κανείς ε, να δει τι, πώς κλείνουν στόματα στην Ιταλία όσων δεν συμφωνούν με το σύστημα. Εγώ πιστεύω λοιπόν ότι αυτό το βιβλίο είναι ένα μια πολύ σοβαρή δουλειά που μπορεί να αποτελέσει τη βάση προβληματισμού. Πέρυσι είχαμε πει να φτιάξουμε μία επιτροπή για να εξετάσουμε το θέμα των μαφιών στην Ευρώπη. Μπορούμε εμείς να αρχίζουμε να φανταζόμαστε ότι το ε, μοντέλο της μαφίας είναι το μελλοντικό μοντέλο το ευρωπαϊκό μοντέλο πλέον διαφθοράς ε, γιατί αυτό το μοντέλο θα κατακλείσει την Ευρώπη του μέλλοντος στη διακλάδωση μεταξύ εξουσίας, απάτης κλπ. Και δίνω τώρα ένα παράδειγμα και κλείνω. Αν ας πούμε μια μαφιόζικη επιχείρηση θέλει να κερδίσει έναν διαγωνισμό, μια δημοπρασία στο Παλέρμο θα έχει μεγάλα προβλήματα διότι η νομοθεσία είναι πολύ προσεκτική. και αν τα καταφέρει τότε πρέπει να παρουσιάσει και την έκθεση αντιμαφίας. Εγώ ως δήμαρχος στην πόλη μου έλεγα ότι όσοι συμμετέχουν σε έναν διαγωνισμό θα πρέπει να έχουν αυτό το χαρτί του αντιμάφια, δηλαδή το πιστοποιητικό καθαρού ποινικού μητρώου για την έναν της μαφία. Το ζήταγα από πριν. Αλλά όμως η επιχείρηση αυτή η οποία δεν μπορεί να κερδίσει τη δημοπρασία στο Παλέρμο ή στη Ρώμη τότε κερδίζει μια δημοπρασία, έναν διαγωνισμό στο Βερολίνο, στη Μαδρίτη ή στο Παρίσι ή στο Λονδίνο για τον απλούστατο λόγο ότι αυτές οι χώρες δεν έχουν καμία προληπτική διάταξη σχετικά. Και εμείς αφελώς σήμερα πιστεύουμε ότι έναντι της μίας μαφίας ε, σαν την Ιταλική ας πούμε που διαχειρίζεται 250 δις ευρώ το χρόνο αυτά που χρειάζεται δηλαδή η Ελλάδα στις παράνομες δραστηριότητες μιλάμε της μαφίας ε, Ε, και πόσο μάλλον σε ευρωπαϊκό επίπεδο όταν διαχειρίζονται δύο τετράκις εκατομμύρια ευρώ το χρόνο ε, δεν μπορούμε να γνωρίσουμε λοιπόν ότι αυτή η διαχείριση δημιουργεί και διαβρώνει τον κορμό της οικονομίας. Πήραμε μια ολόκληρη ώρα με αυτή τη συζήτηση. Έχουν εξαντληθεί τα θέματα. Υπάρχουν κάποια σημαντικά ακόμα, αλλά θα ήθελα κάποια πρόσθετα σχόλια να γίνουν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλει να παρέμβει, παρακαλώ, ναι. Θέλετε. Έχετε τον λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα είμαι πολύ σύντομος, Πρόεδρε. Έχουμε ξεπεράσει τον χρόνο για αυτό το θέμα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καλωσορίζει τα, τη μελέτη και τα αποτελέσματά της. Θεωρούμε ότι είναι επικοδομητικά αυτά για τη δουλειά. Δεν μπορώ τώρα να αναφερθώ σε όλα τα σχόλια που έγιναν από τους ευρωβουλευτές. Επιτρέψτε μου όμως ένα κέριο σημείο να αναφέρω. Δεν πρέπει να ξεχαστεί αυτό ότι ουσιαστικά όλα τα στοιχεία για τη διαφθαρά που υφίστανται και είναι διαθέσιμα μέχρι σήμερα είναι όπως επίσης υπογράμμισε η έκθεση βασίζονται στην ε, εντύπωση που δημιουργείται από αυτά perception και αυτό είναι ένα πρόβλημα εδώ. Και αναφέρθηκε ότι είναι βραδύσια η ρυθμή τη εργασία τη Ευρωπαϊκή Επιτροπής. Θα θέλω όμως να σας διασφαλίσω ότι εργαζόμαστε για την καταπολέμηση της ε, διαφθοράς ε, Κάνουμε τη δουλειά μας και αξιολογούμε αυτή τη στιγμή, σε αυτή τη φάση, το πως μπορούμε να αντιμετωπίσουμε την Situation Report, την έκθεση πεπραγμένων για την αντιμετώπιση της διαφθοράς στην Ένωση, τι μπορεί να γίνει για την data collection, τη συλλογή στοιχείων, ώστε να επιτευχθεί αυτή, αυτός ο στόχος και βρισκόμαστε στη διαδικασία αξιολόγησης assessing της ε, απόφασης πλαισίου για την ε, αδιαφθορά και στον ιδιωτικό τομέα. Να δούμε με πόσο επιτυχή τρόπο υλοποιήθηκαν οι προτάσεις μέχρι σήμερα. Ευχαριστώ Πρόεδρος. Σας ευχαριστούμε. Και υπάρχει σχετικά, είναι η βεβαιότητα, με βεβαιότητα μπορούμε να πούμε ότι δεν είναι η τελευταία φορά που συζητάμε την διαφθορά και το συσχετισμό της με το οργανωμένο κλίμα, ε, έγκλημα σε αυτή την κοινοβουλευτική μας Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών. Σίγουρα και στο ανώτατο επίπεδο θα τύχει συνέχεια του θέματος και θα έχουμε επαφή με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ε, για πρόσθετα πέντε λεπτά που απομένουν έχετε τον λόγο εσείς ε, για να κάνετε κάποια σχόλια ή συμπεράσματα να διατυπώσετε σε σχέση με τις παρατηρήσεις και τις ερωτήσεις που έγιναν από τα μέλη της Επιτροπής. Σας ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Κυρίες ε, και κύριοι μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, είναι πραγματικά χαρά να βλέπει κανείς τόσες πολλές ερωτήσεις και υποστήριξη από πλευρά σας. Θα ήθελα να αναφέρω μόνο δύο πράγματα πριν δώσω τον λόγο στον συνάδελφο για τις τελικές παρατηρήσεις του. Θα ήθελα να πω ότι πραγματικά δεν είναι αξιόπιστα τα στοιχεία είπαν μέχρι σήμερα. Είχαμε όμω ε, τη μέθοδο έρευνα που διασφάλιζε ότι θα είναι πιο αξιόπιστα αυτά τα στοιχεία αν πρόκειται να ληφθεί κάποια απόφαση σε ευρωπαϊκή κλίμακα με βάση αυτά τα στοιχεία. Και έχουμε όχι εντυπώσει, ε, perceptions ή απεικονίσει, αλλά και αντικειμενικά στοιχεία, αξιόπιστα στοιχεία. Και για να πω για την πρόσθετη αξία κάτι αυτού του εγχειρήματο, ήταν μία από τι ερωτήσει που διατυπώθηκαν από την κυρία Ντέλτσεβα το καταστήσαμε σαφές όμως θα έπρεπε να πω ότι και ο τελευταίος που παρενέβη το κατέστησε σαφές ότι δεν υπάρχει εύρυθμη ε, λειτουργία τη εσωτερική αγορά στην Ευρωπαϊκή Ένωση αν δεν αντιμετωπιστούν όλα τα θέματα και τα προβλήματα με τον σωστό τρόπο. Και θα ήθελα να επισημάνω ότι έχει ήδη πείρα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στι βέλτιστέ προδιαγραφέ, benchmarking για την ε, ε, καταπολέμηση τη διαφθορά. Και υπάρχει και μηχανισμό για την καταπολέμηση τη διαφθοράς στη Βουλγαρία και Ρουμανία. Και πρέπει να επεκταθεί αυτό το πλαίσιο με ένα πιο ανοιχτό, σε ένα πιο ανοιχτό ευρύτερο πλαίσιο και έτσι να μπορέσει μπορέσει να ε, λειτουργήσει για να είναι πιο αποτελεσματικό. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Μονογραφική η απάντηση και τα υπόλοιπα μπορούν να δοθούν γραπτός ε, για τις παρατηρήσεις ε, συμφωνώ για την ανεπάρκεια των πληροφοριακών στοιχείων. Θα ήθελα να δείτε όμως αυτήν την έκθεση διαφορετικά και όχι μόνο σαν κάτι εγκυκλοπαιδικής αξίας Βλέπετε τι είναι, για παράδειγμα, η διαφθορά της αστυνομίας. Δεν μπορείτε να δείτε πώς εκφράζεται για κάθε χώρα, αλλά θα σας δώσει κάποια κατευθυντήρια γραμμή, ένα προσανατολισμό για να αρχίσει η έρευνα. Είναι αφετηρία λοιπόν αυτή η έκθεση και όχι τερματισμός, όχι η γραμμή του τέρματος. Και σας δίνει μια εικόνα καλή πόσο ε, επεκταμένη είναι η χρήση του οργανωμένου εγκλήματος στους ε, διάφορους ε, τομείς για τα σχόλια που έγιναν από τον κύριο Ρούτσεκ. Ίσως έχει τερματιστεί η μεταβατική περίοδος προς τη δημοκρατία στις κεντροανατολικές ε, ε, ευρωπαϊκές χώρες, όμως η καταπολέμηση της διαφθοράς εκκρεμεί ακόμα. Πρέπει να προχωρήσει. Για αυτό που είπατε, η θεσμική προσέγγιση. Συμφωνώ ότι αυτό είναι που χρειαζόμαστε. Αν δείτε την αστυνομική διαφθορά σε μια χώρα, και τη διαρροή πληροφοριών που θα μπορούσατε να την χαρακτηρίσετε μη ηθική, ε, μη διοντολογική συμπεριφορά σε μια άλλη χώρα αυτό θα ήταν φαινόμενο διαφθοράς. Πρέπει να υπάρξει λοιπόν μια ευθυγράμμιση όλων αυτών των ε, ρητών και διατάξεων. Δεν μπορούμε να έχουμε ισοπεδωτικά έναν ορισμό διαφθοράς που θα λειτουργεί για όλες τις περιπτώσεις. Πρέπει να δούμε τα διαφορετικά θεσμικά όργανα και να καθορίσουμε τι είναι πράξεις διαφθοράς ή διαφθορά για κάθε ένα από αυτά τα όργανα. Γιατί διαφορετικά αυτό που βλέπουμε για παράδειγμα στη Γαλλία, που βλέπουμε σε σχέση με τις καταδίκες για τη διαφθορά, ε, βλέπουμε λιγότερες, ε, πιο λίγες ε, καταδίκες, ενώ αλλού μπορεί να υπάρχουν περισσότερες. Σε σχέση με τους ορισμούς συνδέεται αυτό. Και για τον κύριο Μπουσούτη και την παρατήρηση που έκανε για τις, ε, την σαφήνεια των περιπτώσεων. Δεν μπορούμε να βασιστούμε μόνο σε αυτές τις περιπτώσεις. Χρειαζόμαστε πληροφορίες ε, μέσω των υπηρεσιών ε, δίωξης και συλλογής πληροφοριών, των, των υπηρεσιών πληροφοριών. Η έκθεση για την Ιταλία συντάχθηκε από ένα καθηγητή που ουσιαστικά είναι κομμουνιστής όπως πρέπει να πω. Δυστυχώς αυτή είναι η πραγματικότητα. Αυτά είχα να πω. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Μάλιστα, ευχαριστώ λέει ο Πρόεδρος. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε τους εισηγητές και εξ του Κέντρου Δημοκρατικών Μελετών για την μελέτη και μελέτη της Δημοκρατίας για την παρουσίασή τους. Σας ευχαριστούμε λοιπόν. Και τώρα προχωράμε στο επόμενο σημείο στην ημερήσια διάταξη. Ποιο είναι αυτό? Αυτό είναι το σημείο 13 στην ημερήσια διάταξή μας και αφορά το 13 την τροποποίηση στο ψήφισμα που αναφέρει τις τρίτες χώρες των οποίων οι υπήκοοι πρέπει να έχουν θεωρήσεις διαβατηρίων όταν ε, περνούν τα εξωτερικά σύνορα και εκείνων που απαλλάσσονται από αυτές τις θεωρήσεις διαβατηρίων. Είναι σε σχέση με την Επιτροπή μας η συζήτηση αυτή για αυτό το θέμα η συγγήτης ήταν η κυρία, η συγγήτρια η κυρία Τάνια Φαζόν και έτσι θα μπορούσαμε σε σχέση με την εξέταση των σκεπτικών για το σχέδιο έκθεσης για την απελευθέρωση θεωρήσεων διαβατηρίων για την Ελβανία και Βοσνία Ζεγοβίνη μετά από την παρουσίαση από πλευρά. Ε, Τη εισηγήτριας κυρία Φαγιών. Θα ακούσουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τη Βελγική Προεδρία. κυρία Φαγιών, έχει τον λόγο, παρακαλώ. Ε, Σα ευχαριστώ, Πρόεδρε, και ευχαριστώ όλους τους συναδέλφους ε, που είναι θαραλέοι και είναι ακόμα παρόντες στην αίθουσα αυτή την ε, ώρα αυτού του απογεύματος που έχει προχωρήσει και λίγο πριν από τις ερηνές διακοπές τόσο όψιμη. Νομίζω είναι ένα πολύ σημαντικό σημείο αυτό το οποίο συζητάμε και θα ευχόμουν περισσότεροι να ήταν παρόντες διότι πολλοί από τους πολίτες, πολίτες στη Βοσνία, Ζεγοβίνη και Αλβανία παρακολουθούν εκ του σύνεγγυς από πολύ κοντά τις ε, διαβουλεύσεις και συζητήσεις στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τη διαδικασία απελευθέρωσης του καθεστώτος ε, θεωρήσεων διαβατηρίων. Οι θεωρήσεις διαβατηρίων απομόνωσαν τους πολίτες των Δυτικών Βαλκανίων επί υπερβολικά μεγάλο χρονικό διάστημα διάστημα και πέρσι όταν καταργήθηκαν οι θεωρήσεις διαβατηρίων για την Μακεδονία λέει ομιλήτρια Σερβία και Μαυροβούνιο είδαμε ποια μεγάλη επίπτωση είχε για τους πολίτες. Είναι περισσότερο ψυχολογική η επίπτωση, θετικό αποτέλεσμα να μπορεί κανείς να έχει αποκομίσει την εντύπωση ότι ελεύθερα μπορεί να ταξιδέψει κανείς στο εξωτερικό. Και αυτό ήταν θετικό για την, ε, τα Δυτικά Βαλκάνια και για την ε, Βοσνία Ζεγοβίνη και την Αλβανία. Ήθελα να πω ότι στην αρχή αυτού του έτους, το 2010, όταν είχαμε την απελευθέρωση από θεωρήσεις διαβατηρίων για τρεις χώρες, είδαμε ίσως κάποια μικρή αρνητική επίπτωση όταν κάποιοι μετανάστες ε, ή κάποιοι υπήκοοι από αυτές τις τρεις χώρες, ιδιαίτερα από τη Μακεδονία και το Μαυροβούνιο, έφτασαν στο Βέλγιο, στην Ολλανδία και ε, αναζητούσαν εκεί άσυλο ή μια θέση μια εργασίας και θέλω να πω ότι ε, αντέδρασαν καλά οι κυβερνήσεις ε, των χωρών διότι είχαν παραπλανηθεί οι πολίτες αυτοί. Δεν γνώριζαν ότι οι χωρίς θεωρήσεις διαβατηρίου, τα χωρίς θεωρήσεις διαβατηρίου ταξίδια υπέκυντο σε κάποιους περιορισμούς. Ήταν όμως καλό για την Βοσνία Ζεγοβίνη για παράδειγμα και την Αλβανία. Έχουν επενδύσει μεγάλα κεφάλαια για να ε, ε, καταστήσει σαφές ότι ε, υπάρχουν περιορισμοί για, και για 90 ημέρες κιόλας διάρκεια ταξιδίων. Δεν δίνουμε δουλειά ή δεν χορηγείται άσυλο με μια τέτοια δυνατότητα. Υπάρχει η ελευθερία ταξιδίων προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ταξίδεψα πολύ στις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων τους τελευταίους μήνες ως εισηγήτρια και το τελευταίο διάστημα και στη Βοσνία Ζεγοβίνη και στην Αλβανία. Μου δόθηκαν διασφαλίσεις από τις αρχές, κρατικές αρχές, ότι πολλά είχαν γίνει υπό την τεχνική πλευρά και την ετοιμότητά τους. Έκαναν πολλά θετικά βήματα αυτές οι χώρε και αναγνωρίζει αυτό την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και υποστηρίζω απόλυτα εγώ την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο σχέδιο έκθεσή μου χωρίς καμιά τροπολογία να ολοκληρωθεί και να εγκριθεί το καθεστώς απελευθέρωσης από θεωρήσεις διαβατηρίων και να περάσουν από το παράτημα στον λευκό πίνακα. Και προτείνω να εγκρίνουμε όλοι και να δώσουμε σαφή δέσμευση όλοι ότι είμαστε αφοσιωμένοι στη συμφωνία που πετέχθη τον Νοέμβριο σε αυτό το κτίριο με μεγάλη υποστήριξη και με υποστήριξη του Συμβουλίου ότι θα αντιμετωπιστούν αυτές οι δύο χώρες με κατεπήγοντα χαρακτήρα για να αντιμετωπιστούν οι ανάγκες τους. Είναι τώρα το θέμα της δικής μας αξιοπιστίας και κύρους να ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία φέτος. Αυτή την εβδομάδα υπάρχουν πραγματογνώμονε στην Αλβανία αξιολογώντας την το τελικό επίπεδο επίπεδο ετοιμότητας αυτής της χώρας για να προχωρήσει αυτό το καθεστώ. Και από την Βοσνία Ζεγοβίνη και από την Αλβανία έχω διασφαλίσεις και καλέ ενδείξεις ότι πολλά έχουν γίνει και ότι μπορούν πολλά να επιτευχθούν. Υπάρχει πολιτική βούληση και δέσμευση να συνεχιστεί η υλοποίηση και οι δεσμεύσει με τους, ε, τις ε, ε, τομεακές πολιτικές όσον αφορά και τις θεωρήσεις διαβατηρίων. Θα ήθελα να υπογραμμίσω ότι λαμβάνοντας υπόψη ότι αποφασίζουμε αυτά ιδιαίτερα προς όφελος των νέων νέων, της νεολαίας. Και λαμβάνοντας υπόψη ότι πριν από 20 χρόνια οι πολίτες αυτών των χωρών μπορούσαν να ταξιδεύουν χωρίς ε, ε, θεωρήσεις διαβατηρίων. Και σήμερα υπάρχει μια ολόκληρη γενεά νέων που δεν κατάφεραν να ταξιδέψουν ποτέ εκτός της χώρας τους. Και είναι καμιά φορά πολύ δύσκολο να συζητήσει κανείς για ευρωπαϊκές αξίες και αρχές μαζί τους αν δεν γνωρίζουν ε, ε, πράγματα σε σχέση με ε, τα όσα έχουν γίνει. Και θα ήθελα να τονίσω νέα γενναία, για τους νέους, είναι σημαντικό αυτό. Θα τους δίναμε μια ευκαιρία να σπουδάσουν, να κυκλοφορήσουν, να ταξιδέψουν ελεύθερα, να επισκεφθούν ε, στο εξωτερικό οικείους τους και να υπάρξει αυτή η ευκαιρία που θα τους προσφερθεί. Αυτό που θα ήθελα να πω ίσως είναι, και για να ολοκληρώσω εν κατακλείδη, ότι έχουμε την δέσμευση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ότι κατά την αρχή την έναρξη Σεπτεμβρίου όταν θα έχουμε την ε, έκθεση, την προφορική παρουσίαση για το έργο των πραγματογνωμόνων σε αυτές τις δύο χώρες αναμένω ότι θα υπάρξει μια θετική έκθεση που θα δοθεί θετική τελική έκθεση για την ετοιμότητα αυτών των δύο χωρών και είμαι πεισμένη ότι αξίζουν να τύχουν του καθεστώτος απελευθέρωσης θεωρήσεων διαβατηρίων το δυνατόν ταχύτερα. Τώρα είναι δέσμευση από δική μας πλευρά στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που πρέπει να υλοποιηθεί. Ελπίζω το Σεπτέμβριο θα προχωρήσουμε με θετική ψήφιση στην Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών και στην Ολομέλεια νωρί το φθινόπωρο, ώστε να δώσουμε το τελικό πράσινο φω, να προχωρήσει αυτή η έγκριση απαλλαγή από θεωρήσει διαβατηρίων. Ζητώ το Συμβούλιο να πορευθεί προ αυτή την κατεύθυνση και έχουμε δεσμευτεί αυτή η διαδικασία να ολοκληρωθεί με κατεπήγοντα χαρακτήρα. Απευθύνω έκκληση να εγγραφεί αυτό το θέμα στην ημερήσια διάταξη για τον Οκτώβριο και όχι για τον Νοέμβριο, όπω κάποιε φήμε ανέφεραν. Γιατί κάθε μήνα καθυστέρηση στην Ολομέλεια και καθυστέρηση για την απαλλαγή θεωρήσεων διαβατηρίων δημιουργεί πολιτικά προβλήματα σε χώρες που έχουν, ζουν σε μια πολιτική αστάθεια στην περιοχή αυτή. Το τίμημα το οποίο θα πληρώναμε αν δεν υπήρχε η απελευθέρωση θα ήταν πολύ ψηλότερο. Ολοκληρώνω. Είναι ευθύνη μας αυτό. Αποφασίζουμε για την ποιότητα ζωής και την ευημερία των πολιτών αυτών στο, στα Δυτικά Βαλκάνια. Και φυσικά η κύρια ανησυχία όλων παραμένει το Κωσυφοπέδιο και βρίσκεται πάρα πολύ ψηλά στην ημερήσια διάταξη για να βρούμε έναν τρόπο και οι πολίτε του Κωσυφοπεδίου, οι υπήκοοι του Κωσυφοπεδίου να μπορέσουν να τύχουν αυτή τη απελευθέρωση θεωρήσεων διαβατηρίων με τη Βοσνία Ζεγοβίνη και την Αλβανία που θα ακολουθήσουν τις Βοσνία Ζεγοβίνη και Αλβανία, που ελπίζω νωρί το φθινόπωρο να απαλλαγούν από αυτέ τι θεωρήσεις διαβατηρίων. Παρακαλώ, η κυρία εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έχει τον λόγο. Έχετε τον λόγο, παρακαλώ. Uh, Χαιρόμαστε ιδιαίτερα για την έκθεση της κυρίας Φαγιών. Γνωρίζετε τη θέση της Επιτροπής για τα επόμενα βήματα. Από την πλευρά μας πρέπει να οριστεί ενεργοποιηθούν οι τεχνικές αποστολές για να εντοπιστούν τα προβλήματα στα σύνορα και επίσης επαναλάβω βάνω τη δέσμευσή μας να σας ενημερώσουμε για τα αποτελέσματα προφορικά το Σεπτέμβριο. Είναι κάτι που το είχαμε προτείνει πριν από κάποιες εβδομάδες. Ευχαριστώ που ήσασταν σαφείς και σύντομοι. Ας ακούσουμε και τη Βελγική Προεδρία τώρα. Εμίλ Ρέιν. Παρακαλώ. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Αξιότιμοι Ευρωβουλευτές, ε, σήμερα το πρωί ακούσατε αρκετά από τον ε, κύριο ε, Υφυπουργό Γουατλέ από πλευράς της Βελγικής Προεδρίας η Βελγική Προεδρία θέλει να καταβάλει κάθε προσπάθεια να ανταποκριθεί στις κοινοβουλευτικές υποχρεώσεις που έχει, έχουν ανάληφθει έναντι της Βοσνίας Ζεγοβίνης και της ε, Αλβανίας ε, που η απελευθέρωση θεωρήσεων διαβατηρίων είναι ένα πρώτο σημαντικό βήμα υπέρ αυτών. Προτού γίνει αυτό είναι σημαντικό οι νομοθέτες να μπορούν να έχουν πιστεί ότι όλοι οι όροι και οι προϋποθέσεις υλοποιήθηκαν επαρκώς ε, όπως έπρεπε και γι' αυτό χαιρετίζουμε την πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής νέοι πραγματογνώμονες και αποστολές πραγματογνωμόνων να αποσταλούν που θα δραστηριοποιηθούν για να αξιολογήσουν τα πράγματα στις χώρες αυτές. Με την έκθεση των πεπραγμένων αυτών των πραγματογνωμόνων και με την έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής το φθινόπωρο, το Σεπτέμβριο, θα γνωρίζουμε επακριβέστερα σε ποιο βαθμό, σε ποιο μέτρο ανταποκρίνονται στις υποχρεώσεις τους αυτές οι δύο χώρες. Και θα αξιολογήσουμε αν και οι δύο χώρες θα απαλλαγούν από την, ε, τις θεωρήσεις διαβατηρίων. Είναι τεχνικό το πρόβλημα. Πρέπει να, έχει επαρκή, να υπάρχει επαρκής χρόνος ώστε να αξιολογηθούν ε, τα στοιχεία από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και αν διαπιστωθεί ότι ανταποκρίνονται σε αυτές τις υποχρεώσεις χώρες αυτές, τότε να είσαστε σίγουροι ότι η Προεδρία μας θα εγγράψει αυτό το θέμα στις, στην ημερήσια διάταξη του αντίστοιχου Συμβουλίου προ, η και θα ξεκινήσουν οι διαδικασίες ώστε να εγκριθεί τελικά η απελευθέρωσή τους. Έχει μελετήσει την έκθεση της κυρίας Φαγιόν η Προεδρία, η Βελγική Προεδρία και χαίρεται για αυτή τη συνεργασία και τις μελλοντικέ αυτές προοπτικές. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Σχόλια τώρα. Η κυρία Λάτφορντ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Δυστυχώς δεν άκουσα το πρώτο κομμάτι των σχολείων της κυρίας Φαγιόν, αλλά με βάση την προηγούμενη εμπειρία είμαι σίγουρη ότι συμφωνώ με όλα όσα λέει. Αυτό τουλάχιστον γινόταν στο παρελθόν και έχει κάνει πολύ καλή δουλειά για την Επιτροπή ΛΥΜΠΕ. Τουλάχιστον αυτό έκανε πέρυσι. Νομίζω ότι υπάρχουν πολύ καλά επιχειρήματα υπέρ και βεβαίως οι δύο χώρες έχουν κάνει πολύ καλή πρόοδο. Λειτουργεί η αιρεσιμότητα και πιστεύω ότι θα έχουμε μια γρήγορη θετική απόφαση. Είμαι η συγγήτρια της νομοδότησης της ΑΦΕΤ που θα είναι πολύ σύντομη και ελπίζουμε η ψηφοφορία να γίνει αν όλα πάνε καλά στις 6 Σεπτεμβρίου. Στηρίζω λοιπόν και εγώ την έκκληση της συγγήτριας να μπορέσουμε να περάσουμε αυτό το θέμα πολύ γρήγορα στην Ολομέλεια τον Οκτώβριο. Και ένα σύντομο σχόλιο σε αυτά που είπε το Συμβούλιο. Αυτό το θέμα είναι τεχνικό επειδή υπάρχουν τεχνικές προϋποθέσεις για την ε, εκπλήρωση των ε, κριτηρίων απελευθέρωσης των ε, θεωρήσεων και κανείς δεν προτείνει να μειώσουμε αυτές τις τεχνικές προϋποθέσεις. Θα ήταν όμως πολιτική απόφαση να μην εγκριθεί η άρση των θεωρήσεων. Αν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεωρεί ότι πληρούνται τα κριτήρια, αλλά το Συμβούλιο εμποδίζει, καθυστερεί τον φάκελο. Αυτό είναι πολιτική απόφαση και ατυχής απόφαση. Και επίσης είναι απόφαση αντίθετη στα ε, συμφέροντα ασφαλείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπό την ευρεία έννοια. Και να πω επίσης ότι δεν μιλάμε για τους ε, συνήθεις υπόπτους ε, του κέντρου και της αριστεράς που το πιστεύουν αυτό, έχω ακούσει και κεντροδεξιούς να λένε ότι τα ευρεία συμφέροντά μας για την ασφάλεια είναι να υπάρξει προσέγγιση με τους λαούς των Βαλκανίων και των Δυτικών Βαλκανίων. Έτσι λοιπόν μπορούμε να αντιμετωπίσουμε την ε, στενή άποψη που διευκολύνει τις εθνικές εντάσεις σε αυτές τις χώρες. Άρα μιλάμε για μια πολιτική απόφαση επί τη βάση τεχνικών κριτηρίων. Thank you. Σας ευχαριστούμε. Κύριε Μπουσούτη, παρακαλώ. Ναι, σας ευχαριστώ Πρόεδρε υπό το φω τη παρέμβαση τη Σάρα Λάτφορντ να, αποφασι... να αποσαφηνίσω ποια είναι η θέση τη κεντροδεξία. Πρώτα απ' όλα καλωσορίζω την παρέμβαση τη Τάνια Φαγιών και τον τρόπο που αντιμετώπισε αυτό το χαρτοφυλάκιο ευθύ εξ αρχή, θυμίζοντας πάντα τις πολιτικές ε, επιπτώσεις αλλά και τη σημασία των τεχνικών προϋποθέσεων και όρων. Παρεμβαίνω εξ ονόματος ε, της ε, σκιώδους εισηγήτριας Άννα Μαρία Κοράτσα Μπίλτ και εμείς οι ίδιοι θα πρέπει να δούμε τις προοπτικές της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και με την Αλβανία και τη Βοσνία Ριζεγοβίνη ως προοπτική με ανοιχτό πνεύμα και με θετική αντιμετώπιση. Στο τέλος τέλος αυτή είναι η φυσική τους κατοικία θα έλεγα και δεν χρειάζεται να προσθέσω τίποτα επ' αυτού. Τώρα, όσον αφορά για την, την απελευθέρωση από τις θεωρήσεις διαβατηρίων, φυσικά υπάρχουν κριτήρια που πρέπει να υλοποιηθούν και να ικανοποιηθούν. Χαίρομαι ότι μέχρι το Σεπτέμβριο άκουσα ότι θα έχουμε τα τελικά αποτελέσματα για την τήρηση αυτών των κριτηρίων. Και αν τα αποτελέσματα αυτά θα είναι θετικά, ε, τότε φυσικά η κυρία Φαγιών, όπως είπε στη σύστασή της, θα πρέπει να δοθεί συνέχεια και να απελευθερωθούν. Πολύ σωστά το είπατε και έχετε δίκιο ότι έχουμε ευθύνε που επομιστήκαμε και ότι η αξιοπιστία, το κύρος μας διακυβεύεται και ότι είναι βέβαιο ότι θα πρέπει να αρθούμε στο ύψο των περιστάσεων για να είμαστε σωστοί. Ευχαριστώ. Final point. Τέλος, η κυρία Ευχαριστώ και ευχαριστώ και για την υποστήριξη του συναδέλφους. Θεωρώ ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δείχνει συνεχώς σημαντική υποστήριξη στη διαδικασία απελευθέρωσης των θεωρήσεων και χαίρομαι που ακούω και το Συμβούλιο να μας λέει ότι πρόκειται για τεχνική διαδικασία αν και έχω και εγώ τις ίδιες ε, επιφυλάξεις με τους συναδέλφους θεωρώ ότι η τελική απόφαση είναι πολιτική απόφαση σας ζητώ λοιπόν να μην καθυστερήσετε καθόλου την τελική σας απόφαση αφού λάβουμε τις ε, εκθέσεις ε, των των εμπειρογνωμόνων. Και ελπίζω όταν ακούσετε τους εμπειρογνώμονες το Σεπτέμβριο θα μπορέσετε να διευθετήσετε το θέμα με την ίδια ταχύτητα που θα το κάνει και το Κοινοβούλιο, δηλαδή στο τέλος του φθινοπόρου ή στις αρχές του χειμώνα. Ολοκληρώνοντας να πω ότι είμαι σίγουρη ότι το Κοινοβούλιο θα δώσει το τελικό πράσινο φως ε, το φθινόπωρο και θα παραμείνουμε αφοσιωμένοι στη διαδικασία. Θα διασφαλίσουμε ότι οι πολίτες της Αλβανίας και της Βοσνίας Ζεγοβίνης ε, θα είναι ελεύθεροι να ταξιδεύουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και εγώ είμαι πεπισμένη ότι τους αξίζει περισσότερο από ποτέ. Ευχαριστώ. Τελειώνουμε με το χρονοδιάγραμμα. 2 Σεπτεμβρίου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα παρουσιάσει τα αποτελέσματα της αποστολής της Θερινής. 3 Σεπτεμβρίου, 6 το απόγευμα, προθεσμία για τις τροπολογίες. Έχοντας ακούσει και την άποψη της ΑΦΕΤ, μέσω της κυρίας Λάτφορντ μπορεί να έχουμε ψηφοφορία στην Λίμπε στις 17 Σεπτεμβρίου. 17 Σεπτεμβρίου η ψηφοφορία. Σημειώστε το και περνάμε στο επόμενο σημείο της ημερησίας. Περνάμε στο 15, όχι, 14 διευθύνει ο πρόεδρος στην ημερησία διάταξη, ενώ είναι το 15 στην ελληνική ημερησία διάταξη. Ναι, η κατάσταση όσον αφορά τους Ερυθρέους μετανάστες στην Λιβύη μια συζήτηση, μια συζήτηση που διεξάγεται και με εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για ένα θέμα το οποίο εθίγει θέμα το οποίο αναφέρθηκε και υπό το, την κατεπίγουσα διαδικασία από κάποιους από μας με τη διαδικασία του κατεπήγοντος εδώ στην Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών ΛΥΜΠΕ Πρώτα απ' όλα και κύρια, καλωσορίζουμε τον Γενικό Διευθυντή από την ε, ε, Γενική Διεύθυνση Home Affairs εσωτερικών υπό την αρμοδιότητα και ε, καθοδήγηση της ε, Επιτρόπου κυρίας Μάλμστρομ, τον Γενικό Διευθυντή Μασερβίση, ο οποίος ε, θα μας ενημερώσει για την κατάσταση των Ερυθρέων αυτών μεταναστών που ήθελαν να, να περάσουν στην επικράτεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όμως κρατήθηκαν στην Λιβύη. Και το θέμα αυτό πρόσφατα συζητήθηκε και οδήγησε σε μια παρέμβαση για τα ανθρώπινα δικαιώματα, όχι μόνο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά και από τις ε, υπηρεσίες και των Ηνωμένων Εθνών όπως την είπατε αρμοστία ε, των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα του ανθρώπου και το Διεθνές Γραφείο Μετανάστευσης. Μόλις ακούσαμε το επικεφαλής της τελευταίας αυτής αποστολής στην Λιβύη, ο κύριος Λόρενς Χάρτ, είναι εδώ ανάμεσά μας σήμερα. Τον καλωσορίζουμε και αυτόν σίγουρα και του δίνουμε τον λόγο, θα του δώσουμε τον λόγο στη συνέχεια. Όμως η κατάσταση φαίνεται να βελτιώνεται. Και όμως από την άλλη πλευρά το θέμα της αντιμετώπισης των μεταναστών και προσφύγων στην Λιβύη, στην επικράτεια της Λιβύης, βρίσκεται ακόμα στο τραπέζι και διαπραγματεύσεις βρίσκονται υπό εξέλιξη μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Λιβύης για μια γενικότερη συμφωνία μεταξύ ΕΕ και Λιβύης και για το θέμα της ε, επανυποδοχής ε, ε, και ήδη επαφές έχουν γίνει στην αρχή του, έναρξη του 2009 με τον Αντιπρόεδρο Μπαγό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που είχε επιληφθεί τότε του θέματος. Δίνουμε τον λόγο λοιπόν στον Γενικό Διευθυντή κύριο Μαρζερβίζη και μετά θα έχουμε μια σύντομη ανταλλαγή απόψεων ίσως ο συνάδελφός μας κύριος Παντζέρη θα ήθελε να παρουσιάσει ένα θέμα το οποίο αναφέρθηκε ως κατεπήγον. Κύριε Παντζέρη παρακαλώ έχετε τον λόγο. Θα θέλατε να το σχολιάσετε. Μα σερβίσει, παρακαλώ. Εδώ είσαστε θέλετε να λάβετε τον λόγο παρακαλώ. Okay. Then, apparently... Προφανώς ο κύριος Μαρσερβίση βρίσκεται καθοδόν, δεν είναι εδώ ανάμεσά μας. Και ίσως λοιπόν μπορούμε να δούμε κάποιο άλλο θέμα, κάποια, να ακούσουμε κάποια άλλα σχόλια επί του θέματος, ίσως από τον εκπρόσωπο του IOM, του κυρίου Χάρτ που είναι παρόν, να ακούσουμε τις παρατηρήσεις του. Θα θέλατε να μας κάνετε κάποια σχόλια και παρατηρήσεις ενώ αναμένουμε να προσέλθει ο κύριος Μαρσερβίση. Θα θέλατε εσείς να παρέμβετε. Εδώ είναι, προσέρχεται. Μάλιστα, πολύ ωραία. Κύριε Μασεβίση, παρακαλώ. Εδώ είσαστε, έτσι. Αν θέλετε να λάβετε τον, να καθίσετε και μετά σας ευχαριστούμε που ήρθατε. Καλώς ήρθατε. Καλώς ορίσατε. Ecco, di qua, di Ecco, abbiamo risolto il vuoto occasionato dalla non presenza del... lisame το κενό που είχαμε. Κύριε Μασερβίση, έχετε το λόγο. I did. Now we hear from you. Uh, uh, um, Ευχαριστώ. Θα ήθελα να υπογραμμίσω ότι ουσιαστικά ήρθα για να ακούσω τις ανησυχίες σας. Ας σας πω όμως ε, και λίγο τι κάναμε. Γιατί υπάρχει δημόσια συζήτηση αλλά δεν ε, υπάρχουν πολλές πληροφορίες από πρώτο χέρι. Καταρχάς, τι γινόταν με αυτή την ομάδα πολιτών της Ερυθρέας στη Λιβύη. Γνωρίζουμε μέσω ατύπων επαφέων από τον τύπο, από μη κυβερνητικέ οργανώσεις και άλλες επαφές Βεβαίω είμαστε σε επαφή και με τον είπα αρμοστή του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες. Τι γνωρίζουμε λοιπόν. Προς το παρόν υπάρχουν 400 που έχουν συλληφθεί, κρατούνται ως λαθρομετανάστες. Μέχρι προσφάτως 250 σκόπευαν να ταυτοποιήσουν οι Λιβιακές αρχές. Κρατούνται στο κέντρο υποδοχής στη Μιζουράτα Γνωρίζουμε επίσης ότι τότε είχαν γίνει πολλές άτυπες παρεμφάσεις, αλλά και μια ισχυρή παρέμβαση από την Ιταλική κυβέρνηση, τον Υπουργό φατίν και τον κύριο Μπαρό που μαζί με τις πρωτοβουλίες του ΟΗΕ οι Λιβιακές αρχές έκαναν τις εξής διευκρινήσεις ότι δεν σκοπεύουν να απελάσουν κανένα και σκοπεύουν να συνεργαστούν με οποιονδήποτε ενδιαφέρεται για να υπάρξουν καλές συνθήκες ε, κράτησης και για να επιστρέψουν οι πρόσφυγες ε, στο αρχικό κέντρο κράτησης στη Μιζουράτα που από ό,τι φαίνεται έχει καλύτερες συνθήκες. Μας ανησυχεί ιδιαίτερα το θέμα. Όμως Έχουμε λάβει διάφορες πληροφορίες εμέσως αλλά και άμεσα από τον Υπουργό, τον κύριο Μουσακουσούν, τον Υπουργό Εξωτερικών που είπε ότι θα μας δώσουν όλες τις απαραίτητες πληροφορίες και διασφαλίσεις για τη μεταχείριση των ατόμων αυτών καθώς και διασφάλιση ότι δεν έχουν καμία πρόθεση απέλασής τους. Ζητούν όμως από την Ευρωπαϊκή Ένωση να συνεργαστεί μαζί τους γιατί όπως μας υπενθυμίζουν συνεχώς η Λιβύη έχει 4.000 ε, χιλιόμετρα σύνορων με την υπόλοιπη Αφρική και χρειάζονται βοήθεια στη διαφύλαξή τους. Αυτό είναι κάτι που επανέλαβε και ο κύριος Μοσακός, αλλά είπε ότι θέλουν να τους μεταχειριστούν ανθρώπινα και θέλουν να συνεργαστούν με την τη ορμοστία του ΟΕ για τους πρόσφυγες. Πάντως δεν υπήρχε συμφωνία με τον ΟΕΕ και η Λιβύη δεν έχει υπογράψει τη σύμβασή της να του 51. Παρόλα αυτά θέλουν να συνεργαστούν και η Γενική διεύθυνση, ο Γενικός Διευθυντής επισκέφθηκε τη Λιβύη σε γενικές γραμμές. Εμείς έχουμε συνεργαστεί σε πολλά project με τη Λιβύη και πρόκειται να κάνουμε το ίδιο και στο μέλλον στα πλαίσια των διαφόρων κανόνων συνδρομής. Στο πλαίσιο αυτό, οι διαπραγματεύσεις για την Συμφωνία Πλαίσιο Συνεργασίας περιλαμβάνει και ένα κεφάλαιο για τις εσωτερικές υποθέσεις που ασχολείται με όλα αυτά τα θέματα. Όμως, προς το παρόν, επί του κεφαλαίου αυτού δεν έχουν υπάρξει συζητήσεις ούτε και πρόεδρος. Η συνάντηση όμως με τον Υπουργό, τον κ. Μουσακούσιλ, από ό,τι φαίνεται άνοιξε το δρόμο γιατί μας λένε ότι ενδιαφέρονται να συζητήσουν αυτό το θέμα τις επόμενες εβδομάδες. Άρα, ενώ η συμφωνία με τη Λιβύα μέχρι στιγμής περιοριζόταν στα άλλα γνωστά κεφάλαια συνεργασίας και δεν είχε γίνει τίποτα στο κεφάλαιο εσωτερικές υποθέσεις, τώρα με την πίεση που υπάρχει και εξαιτίας αυτού του περιστατικού ο κύριος Μουσακούσελ και η Λιβύη ενδιαφέρονται να συζητήσουν αυτά τα θέματα όπως υπόθηκε και στην κυρία Μάλστρομ. Αυτά λοιπόν μπορούμε να πούμε από πλευράς στοιχείων που διαθέτουμε. Βεβαίως παρακολουθούμε εκ του εγγύς το θέμα και προσπαθούμε να λάβουμε πληροφορίες σε πολιτικό επίπεδο. Γιατί εδώ μιλάμε για τις πολιτικές μας σχέσεις με τη Λιβύη, δεν μιλάμε για εφαρμογή νομοθεσίας ή συμφωνίας συγκεκριμένης. Αυτά από την πλευρά μου. Ευχαριστώ. Μάλιστα, σας ευχαριστούμε. Τώρα ήρθε ο χρόνος να ακούσουμε από τον εκπρόσωπο του IOM. Παρακαλώ η Επιτροπή Εξωτερικών, η κυρία Γκόμες, θέλει να παρέμβει. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Είμαι εδώ υπό την ιδιότητά μου ως αναπληρωματικού μέλους αυτής της Επιτροπής επιπλέον. Το μικρόφωνο σας κυρία μου, το μικρόφωνο δεν λειτουργεί, δεν είναι αναμένο. Έτσι νόμιζα. Απλά θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο για τις πληροφορίες που μόλις έδωσε. Συμπίπτουν με τις δικές μου πληροφορίες που έχω όσο, καθώς κατάφερα από τα Ηνωμένα Έθνη, από την ύπατη αρμοστία να λάβω. Δεν το ήξερα και το καλωσορίζω ότι θα υπάρχει μια συνάντηση της κυρίας, υπάρχει μια συνάντηση της κυρίας Επιτρόπου Μάλμστρομ με τον κύριο Μασακούσα, Υπουργό Εξωτερικών είναι ένα πολύ θετικό θα έλεγα στοιχείο στις εξελίξεις αυτές. Εγώ ίδια ως εισηγήτρια για τη μελλοντική συμφωνία πλαίσιο για τη Λιβύη που είναι αντικείμενο διαπραγμάτευσης ήρθα σε επαφή με την πρεσβεία της Λιβύης και η πληροφορία που είχα, οι πληροφορίες που είχα πριν από μια εβδομάδα για αυτά τα προβλήματα με τους 400 υπηκόους της Ερυθρέας και και βλέπω ότι πραγματικά δεδομένης της προσοχής που έτυχε αυτό το θέμα εδώ από την Ευρωβουλή και από τα μέσα ενημέρωσης και σε κάποια κράτη-μέλη ήταν πραγματικά, πώς να το πω, με θετικό τρόπο. Ήταν το γεγονός ότι οδήγησε αυτό στις άμεσες αυτές επαφές μεταξύ της κυρίας Μάνστραμ και του Υπουργού Εξωτερικών της Λιβύης τώρα πια. Και ότι υπάρχουν αυτές οι διασφαλίσεις που δίνονται από τη Λιβύη ότι αυτά τα άτομα δεν θα επιστραφούν στην Ερυθρέα. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Οι πληροφορίες οι οποίες πήρα πρέπει να πω ότι λένε ότι κάποια από αυτά τα άτομα είχαν πραγματικά, πώς να το πω, ήταν άτομα που είχαν επιστραφεί από κάποια κράτη-μέλη στη Λιβύη λόγω του ότι θεωρήθηκαν σαν παράνομοι μετανάστες ήταν άνθρωποι οι οποίοι ποτέ δεν είχαν εξεταστεί από την ύπατη αρμοστία των Ηνωμένων Εθνών διότι είχε ε, διωχθεί η ύπατη αρμοστία από τη Λιβύη είχε εκδιωχθεί όπως αναφέρθηκε σαν αποτέλεσμα αυτής της ειδική περίπτωσης πέρα από τις διασφαλίσεις που ανέφερε ο κύριος Μασεβίση ότι δεν θα επιστραφούν στην Ερυθρέα υπάρχει και μια άλλη θετική εξέλιξη ότι η ύπατη αρμοστία για τους πρόσφυγες τώρα συζητεί την δυνατότητα της πιθανής επιστροφής αυτών αυτών των, ε, της πιθανής επιστροφής της στη Λιβύη με το καθεστώς της είπα της αρμοστίας. Αυτό είναι πολύ χρήσιμο για τη συμφωνία που προσπαθεί να πετύχει η Ευρωπαϊκή Ένωση με τη Λιβύη αυτή τη στιγμή και που αφορούν και τα θέματα μετανάστευσης αλλά και προσφύγων και που πρέπει πολύ σοβαρά αυτά να ληφθούν υπόψη. Γιατί μια και κάνουμε λόγο για μια χώρα η οποία ποτέ δεν επικύρωσε τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για την προστασία των προσφύγων. Ούτε καν αναγνωρίζει ότι υπάρχουν πρόσφυγες καν στον κόσμο. Παρόλο το γεγονός ότι η Λιβύη είναι πραγματικά μέρος της ε, σύμβασης της ε, Ένωσης της ε, Αφρικής, των χωρών της Αφρικής για τους πρόσφυγες. Για μας λοιπόν όσον αφορά αυτή την προσέγγιση και την επίλυση αυτού του προβλήματος, αυτού του συγκεκριμένου προβλήματος, εμένω ότι δεν θα επιστραφούν στην Ερυθρέα αυτά τα άτομα, αυτό είναι κέρια σημασίας στοιχείο και ότι προφανώς θα τους δοθεί κάποιο καθεστώς ώστε να παραμείνουν και να μπορέσουν να εργάζονται στη Λιβύη. Παρ' όλα αυτά όμως πέρα από αυτά θα είναι πολύ σημαντικό να αντιμετωπιστεί το βασικό θέμα. Τι κάνει η Λιβύη και πώς συνεισφέρει για την προστασία των προσφύγων ώστε να δοθεί ευκαιρία στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο Ευρωκοινοβούλιο να εγκρίνει μια συμφωνία που θα εντάσσει στο πλαίσιο της αυτά τα θέματα. Αυτά είχα να πω Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ. Πρόεδρο σας ευχαριστώ. Και τώρα σύντομα να ακούσουμε από την IOM, εκπρόσωπο του IOM. Θα θέλατε να λάβετε εσεί τον λόγο παρακαλώ. Σα ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Καλό απόγευμα κύριε και κύριοι. Ευχαριστώ κύριε Μασεβίση για την ε, εισήγησή σας που με χαρά επιβεβαιώνω ικανοποιημένος επιβεβαιώνω στα όσα αναφέρατε ως στοιχεία. Η προαναγγελία της απελευθέρωσης των Ερυθρέων αυτών πολιτών ε, επισημοποιείται τώρα επίσημα και έχουμε και από πλευράς των οργανώσεων στη Λιβύη από το 2006 που από την ύπατη αρμοστία των ΗΕ για τους πρόσφυγες εργαζόμαστε από κοινού για την προστασία και επανεγκατάσταση των προσφύγων και των ετούντων άσυλο. Αυτές τις μέρες αυτό που κάναμε ήταν είχαμε μια άτυπη δράση σε σχέση με τις πρεσβείες ε, και όσους εμπλέκονται στη Λιβύη αλλά και τους εκπροσώπους της κυβέρνησης της Λιβύης για να αναζητηθεί μια λύση έναντι της απέλασης που επετεύχθη θα έλεγα τώρα και τώρα βρισκόμαστε και σε σταθερή μόνιμη επαφή με την κοινότητα της Ερυθρέας που αναφέρει επανεγκατάσταση αυτών των ατόμων ως τελικό του στόχο. Αυτό ως λύση το βλέπουν ως μια μεσ μεσοπρόθεσμη λύση, μια ενδιάμεση λύση και όχι μια, ως μια τελική λύση. Σε σχέση με το Υπουργείο Εργατικού Δυναμικού της ε, ε μουσουλμανικής Τζαμαχηρία, της ε, Ισλαμικής Δημοκρατίας ε, της Λιβύης δηλαδή, έχει αναλυφθεί ε, υποχρέωση ότι θα υπάρχει δυνατότητα να υπάρξει απασχόληση για αυτά τα άτομα και όσον αφορά και τους Σομαλούς στο παρελθόν, όπου απελευθερώθηκαν τότε οι Σομαλοί από τα κέντρα κράτησης και επετράπει να εργάζονται τώρα και να παραμείνουν εργαζόμενοι στη Λιβύη. Καθώς μιλάμε τώρα η κατάσταση είναι ενρευστό ακόμα και μετεξελίσσεται διαρκώς. Πριν από κάποιες ώρες ε, μας είπαν ως στοιχείο ότι υπάρχει μια εντολή που εκκρεμεί από το Υπουργείο Εσωτερικών να απελευθερωθούν όλα τα άτομα που βρίσκονται στα κέντρα κράτησης. Όχι μόνο οι πήκοοι της Ερυθρέας αλλά όλα τα άτομα σε τέτοια κέντρα κράτησης. Χιλιάδες άτομα λοιπόν που κρατούνται σε 18 τέτοια κέντρα κράτησης στην Λιβύη υποτίθεται ότι θα απελευθερωθούν. Δεν γνωρίζουμε ακόμα αν σε αυτή τη φάση οι υπήκοοι της Ερυθρέας θα επιτραπεί να εργάζονται ή θα απελευθερωθούν απλώς. Είναι ενρευστό η κατάσταση, δεν έχει οριστικοποιηθεί ακόμα. Προσπαθούμε να παρακολουθήσουμε τις εξελίξεις στο μέτρο του δυνατού. Θα δούμε τι γίνεται. Το Υπουργείο Εσωτερικών επίσης ζήτησε από την IOM άτυπα σήμερα το απόγευμα να επιτηρηθεί η απελευθέρωση των ε, υπηκών της Ερυθρέας. Θα το κάνουμε εμείς αυτό, θα αναλάβουμε αυτό το καθήκον, τη απουσία της ΥΠΑ της Αρμοστίας των Ηνωμένων Εθνών που έχει απελαθεί από τη Λιβύη, να δούμε πώς θα διαμορφωθεί αυτή η απελευθέρωση αυτών των πολιτών. Να προσθέσω δύο-τρία πράγματα για την προστασία των προσφύγων που σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία είναι 12.000 αυτοί στη Λιβύη σήμερα. Είναι ένα de facto σημαντικό στοιχείο για την προστασία αυτών των ατόμων. Πέρσι δεν έγιναν απελάσεις ε, προς την Ερυθρέα και επίσης και προς την Σομαλία που είναι οι δύο κυριότερες χώρες από τις οποίες προέρχονται αυτοί οι πρόσφυγες και οι αιτούντες άσυλο στην Λιβύη. Όπως σας προανέφερα η κατάσταση είναι η εξής Κάποιοι μεταφέρθηκαν σε ένα κέντρο στο νότο της Λιβύης και αυτό δημιούργησε κάποιες ανησυχίες. Γι' αυτό το κέντρο κράτησης στο νότο της Λιβύης είναι το σημείο αφετηρίας για τις πτήσεις επιστροφής προς τις χώρες προέλευσης. Απεφεύθει όμως αυτή η απέλαση και το καλωσορίζουμε ως καλά μαντάτα. Αυτό αφήνει, ανοιχτά κάποιες, ε, αφήνει ανοιχτές κάποιες ε, άλλες εναλλακτικές δυνατότητες, αλλά αυτά είχα να σας πω για να σας ενημερώσω πολύ σύντομα. Σας ευχαριστώ. Από τον συνάδελφο κύριο Πατσέτη να ακούσουμε παρακαλώ τώρα. Εγώ τις προηγούμενες εβδομάδες είχα ρωτήσει την Κομισιόν αν οι διμερείς συμφωνίες διευκολύνουν την ε, τις ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες ή όχι και μου απάντησε η Κομισιόν ότι πολλές φορές οι διμερείς συμφωνίες δυσχεραίνουν αντί να διευκολύνουν. Η κατάσταση λοιπόν είναι, υπάρχει, εκεί είναι. Και σίγουρα υπάρχουν χώρες οι οποίες έχουν σύνορα τα οποία είναι περάσματα και σίγουρα εφαρμόζουν με το, ε, μεταναστευτικές πολιτικές που αυτοί θεωρούν καλύτερες. Αλλά το λέω όμως εδώ και στον εκπρόσωπο της Κομισιόν ε, πραγματικά αγνοούνται οι διμερείς συμφωνίες κυρίως όσον αφορά στις ε, συμφωνίες απέλασης κλπ. Και υπάρχει και μια άλλη σημαντική πλευρά ότι τελικά δεν υπάρχει μία ολοκληρωμένη συμφωνία με όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά είναι μεμονωμένες διμερείς συμφωνίες. Η κυρία Μάλστρομ είπε πρόσφατα σε μία συνέντευξη ότι τα κράτη-μέλη συνάπτουν συμφωνίες αλλά χωρίς να έχουν τη συνένεση των Βρυξελών. Το πρόβλημα λοιπόν υφίσταται. Και το θυμίσατε εδώ ότι η Λιβύη δεν έχει υπογράψει τις διεθνείς συμβάσεις ούτε αναγνωρίζει το καθεστώς του πρόσφυγα. Έχουμε λοιπόν δύο προβλήματα να αντιμετωπίσουμε. Ένα, τι θα απογίνουν αυτοί οι 400 Ερυθρέοι. Τώρα να χρησιμοποιηθούν ε, για εργασίες ε, κοινωνικής ωφέλειας. Ε, τώρα στη Λιβύη είναι λίγο υπερβολικός αυτός ο όρος, άμα φανταστεί κανείς δηλαδή με τι συνθήκες εκπληρούν αυτές τις ε, κοινωνικές εργασίες. Ξέρετε ότι είναι νέοι όλοι αυτοί και στην Ερυθρέα ανυπότακτοι θεωρούνται μέχρι 40 χρονών. Οπότε καταλαβαίνετε τι θα γίνει όταν όλοι αυτοί επανέλθουν πίσω. Βέβαια, κάποιος μπορεί να επιλέξει να ζήσει και να μην πεθάνει, αλλά μπορεί όμως μετά αυτός να, πεθάνει, να αρχίσει να πεθαίνει σιγά σιγά παρότι έχει επιλέξει να ζήσει. Πρέπει λοιπόν να το παρακολουθήσουμε το θέμα από πολύ κοντά. Και αν τελικά θεωρούμε ότι όλοι αυτοί ε, ε, είναι δικιούχοι του καθεστώτος του πρόσφυγα, η Ιταλία πρέπει να ασκήσει τις πιέσεις της. Και απ' την άλλη ρωτώ, τι κάνει η Ευρώπη. Σίγουρα ε, γίνεται διαπραγμάτευση. Ξέρω ποιες είναι οι δυσκολίες, αλλά δεν χρειάζεται μία όθηση προς αυτήν την κατεύθυνση ούτως ώστε οι διμερείς συμφωνίες να υποκατασταθούν από μια ευρωπαϊκή συμφωνία και έναν ευρωπαϊκό έλεγχο. Πρέπει να τα σπρώξουμε όλα αυτά μέχρι βάθος. Ξέρω ότι πίσω από όλα αυτά υπάρχουν τεράστιες δυσκολίες κυρίως έναντι μιας χώρας σαν αλλά είναι απαραίτητο να προχωρήσουμε προς αυτήν την κατεύθυνση. Και πρέπει κάτι τέτοιο να γίνει το νωρίτερο δυνατό. Τώρα μπορούν να γίνουν ερωτήσεις. Παρακαλώ, σύντομα, για να μην υπερβούμε το χρονοδιάγραμμα της διερμηνίας. Γιατί έχουμε και άλλα σημεία της ημερήσιας διάταξης που πρέπει να εξετάσουμε. Κυρία Αντζεντίνη. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Είχαμε εγγράψει στην ημερήσια διάταξη προκαιρού το θέμα η απάντηση ποια είναι. Είναι η απάντηση που έδωσε ο κύριο Πατσέρη. Έχουμε τρία προβλήματα δηλαδή μπροστά μα. Η Ερυθρέα είναι η Βόρεια Κορέα τη Αφρική. Όποιο εγκαταλείπει αυτή τη χώρα δεν μπορεί να επιστρέψει σε αυτήν. Διότι τότε, πώ να το πω έτσι, ε, θα τιμωρείται και θα πληρώνει. Όλοι όσοι έχουν εγκαταλείψει την Ερυθρέα έχουν κάποιο λόγο να ετούνται άσυλο ή έχουν λόγο να μην, σοβαρό λόγο να μην επιστρέψουν στη χώρα αυτή. Ποτέ. Όταν γνωρίζει ότι κάποιο έχει εγκαταλείψει την Ερυθρέα, το καθεστώς, τότε η οικογένειά του αντιμετωπίζει προβλήματα. Ε, υφίσταται τα πάνδυνα για την παράνομη αυτή, ας το πω έτσι, μετανάστευση. Είναι πράγματα για τα οποία πρέπει να ε, επομιστούμε τις ευθύνες μας. Δεν υπάρχει καν το πώς θα, το, θέμα, η ρύθμιση, πώς θα αντιμετωπίσει η Λιβύη αυτά τα άτομα. Έχουμε δηλαδή απέναντί μας άτομα που προσπάθησαν να προσέλθουν στην Ευρώπη. Αυτοί οι άνθρωποι δεν είχαν τη δυνατότητα να θέσουν καν αίτηση ετούντες άσυλο σε εμά και συνελήφθησαν εκεί. Έχω ένα άρθρο από μια ε, Ιταλική εφημερίδα της 29ης Απριλίου. 24 ώρες είναι η ε, προθεσμία η οποία αναφέρεται σε αυτό το άρθρο. Μετά λέει από την προαναγγελία ε, σύμβασης μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Λιβύης. Και θα έπρεπε λέει και άλλοι να ακολουθήσουν σε αυτή την πορεία τέτοιων συμφωνιών με τη Λιβύη. Έπρεπε λοιπόν να συμβεί αυτό. Ε, ήταν υποχρεωτικό να συμβεί. Δηλαδή διμερείς συμφωνίες με μια χώρα σαν τη Λιβύη Λιβύη πολυμερείς συμφωνίες με μια χώρα σαν την Λιβύη που με αυτόν τον τρόπο αντιμετωπίζει ετούντες άσυλο επιτρέπεται εμείς να έχουμε μια τέτοια σχέση με μια τέτοια χώρα και να προωθούμε σε τέτοιες συμφωνίες και πώς ε, συμφωνούμε όταν αφορά τις αιτήσει ασύλου από αυτά τα άτομα και δεύτερον πώς θα μεριμνήσουμε τώρα ώστε άνθρωποι που βρίσκονται καθοδόν προς την Ευρώπη θα αφαιρούνται δεν θα έχουν το δικαίωμα να θέσουν αίτηση ασύλου επαρκούμε τα σχόλια πρόεδρε. Πρέπει να τα δούμε όλα αυτά υπό το φως που πρέπει ε, των υποχρεώσεών μας έναντι της Βόρειας Κορέας της Αφρικής που είναι η Ερυθρέα. Και υπό αυτό το πρίσμα όσοι έχουν, ε, έχουν πολιτι... Ε, ε, υποχρεώσεις στράτευσης και έχουν εγκαταλείψει τη χώρα και έτσι υφίστανται τα πάνδυνα αυτοί δεν έχουν καν τα δικαιώματά τους. Ευχαριστώ. πρόεδρο ευχαριστώ. Έχουμε ένα κατάλογο, τώρα ε, ολοκληρώθηκε, έληξε αυτός ο κατάλογος. Παρακαλώ, δύο λεπτά ο καθένα για να ολοκληρώσουμε. Κυρία Φλότρο. Ε, δύο λεπτά, κυρία Φλότρο. Bon, évidemment, euh, euh, ε, ναι, Φυσικά αυτή η νέα υπόθεση των Ερυθρέων με το δραματικό της χαρακτήρα και που αφορά σε πρόσφυγες που όπως είπε και η συνάδελφος ε, προέρχονται από μια χώρα όπου δεν συζητιέται ιδιαίτερα το θέμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ε, υπάρχει και το θέμα της ε, συμφωνίας της Λιβύης με την Ιταλία, δηλαδή με την απέλαση των μεταναστών και καταδικάστηκε ε, και από την ε, αρμοστία και από άλλους οργανισμούς ε, και από το δικαστήριο του Στρασβούργου. Ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι με τη Λιβύη δεν έχουμε κανένα περιθώριο συζήτησης ούτε για δικαιώματα ούτε για τίποτα. Και οι Ευρωπαίοι έχουν ε, πολλαπλές επαφές ε, και συνομιλητές ε, στην Λιβύη αλλά από την άλλη μεριά βλέπουμε ότι οι Λίβοι πραγματικά έχουν σκυλιάσει με αυτή την υπόθεση. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει 400 άτομα, τι θα απογίνουν αυτοί. Αλλά η ύπατη αρμοστία έχει βρει ότι είναι 9.000 άτομα τα οποία κρατούνται και τους κακομεταχειρίζονται ε, και ε, η κράτηση είναι σε κάκιστες ε, συνθήκες και η Ευρώπη δεν μπορεί να ασκήσει τον ελάχιστο έλεγχο για τους συγκεκριμένους όρους υποδοχής. Αυτό που εμείς ξέρουμε ε, για όσους επισκέφθηκαν μερικά από αυτά τα κέντρα, η κατάσταση είναι καταστροφική και βασιλεύει η απόλυτη ευθερεσία. Λοιπόν, και το βασικό ερώτημα, μα τι κάνουμε όταν συζητάμε με τη Λιβύη και τις λέμε να ελέγχει τις ροές, να κρατάει τους μετανάστες ε, στα σύνορα και να ε, κρατάει και αυτούς ε, που ψαρεύονται στη Μεσόγειο. Λοιπόν, από αυτήν τη δραματική υπόθεση, τι συμπέρασμα ανασύρει η Κομισιόν για τις τρέχουσες διαπραγματεύσεις με την Λιβύη. Ο κύριος Γιακολίνο, δύο λεπτά. Ακούσαμε μερικά νέα στοιχεία, τα οποία δεν γνωρίζαμε. για τους 244 Ερυθρέους που πέρασαν αυτή τη δραματική περιπέτεια και τις 12.000 που έτυχαν παρέμβασης σήμερα Είχαμε εδώ την Βελγική Προεδρία, τον Υπουργό για τη, τη Μετανάστευση, ο οποίος τόνισε ότι υπάρχει αναγκαιότητα να οικειοποιηθεί η Ευρώπη όλων αυτών των διημερών συμφωνιών που έχουμε. Γνωρίζει πολύ καλά ο συνάδελφος Παντζέρη σήμερα η Ιταλία μαζί με άλλες χώρες, την Μάλτα, την Ισπανία που έχουν κάνει αυτές τις διμερείς συμφωνίες. Αλλά αυτή την ε, πραγματική αλληλεγγύη όπως την ορίζει και το πρόγραμμα της ε, Στοκχόλμης και πρέπει αυτό να το συμφωνήσουμε όλοι και δεξί και αριστερή και κεντρώη ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να λειτουργήσει συμπληρωματικά με τα κράτη-μέλη και να δώσει μία όθηση σε αυτήν την υπεύθυνη στην υπεύθυνη αλληλεγγύη. Δεν είναι η Ολλανδία ο Βιν van der ο οποίος ε, θα υποστεί την μετανάστευση. Είναι οι παράλληλες χώρες που μπορεί να τις προσεγγίσει κανείς πιο εύκολα. Και ξέρετε ότι οι ε, μεταναστευτικές ε, ρότες έχουν αλλάξει. Πολλοί πλέον φεύγουν από την Τινησία σήμερα. Πρέπει λοιπόν να υπάρξει ρύθμιση των μεταναστευτικών ροών όπου οι δύο οδηγίες για τους εποχιακούς εργαζόμενους και τις επιχειρησιακές μεταθέσεις και μεταφορές πρέπει να λυθούν. Ο κύριος, Ταβάρης, δύο λεπτά παρακαλώ. Σας ευχαριστώ πρόεδρε. Φυσικά καλά μαντάτα είναι ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν θα καταλήξουν σε ισόβια ή σε εκτέλεση επιστρέφοντας στη χώρα τους και έτσι δεν θα επιστρέψουν εκεί. Όμως εδώ να δούμε, να μην διολυστήσουμε σήμερα σε μια άγνωστη κατεύθυνση. Η Human Rights Watch είπε ότι οι κρατούμενοι ε, βρίσκονται υπό καθεστώς περιορισμένο τριών μηνών και έτσι έχουν περιορισμένη διάρκεια και μετά όταν θα λήξει αυτή η περίοδος θα πρέπει να αναζητήσουν ένα έγγραφο ταξιδιωτικό ε, ηθαγένειας της Λιβύης. Για να το κάνουν αυτό πρέπει να έχουν ταξιδιωτικά έγγραφα της Ερυθρέας. Αυτά τα καλά μαντάτα εντό εισαγωγικών μας φέρνουν αντιμέτωπους με ένα ηθικής διάστασης ε, εμβέλεια στοιχείο. Συμφωνίες με τη Λιβύη ήταν λέει καλές, καλά μαντάτα για τη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών από πλευρά τη Ευρώπης. Πού καταλήγουμε. Νομίζω ότι δύο κύρια σημεία έχουμε μπροστά μας. Το ένα αφορά τους υπηκόους της Ερυθρέας συγκεκριμένα. Η ιδέα ότι θα έχουν ένα κοινωνικό, πώς θα το πω, καθεστώς κοινωνικής εργασίας στη Λιβύη, να μην μας δημιουργεί αυτά ότι οικονομικά είναι, θα είναι οικονομικοί μετανάστες, αυτό θα ήταν μία από τις πιο τρομερές ε, παράπλευρες επιπτώσεις αυτής της ε, κατάστασης. Είναι άτομα που θα είχαν δικαίωμα να θέσουν ε, αίτηση ασύλου. Αυτό με φέρνει στη δεύτερη παρατήρηση. Η γενική δηλαδή η διασφάλιση ότι δεν τηρεί τις υποχρεώσεις και τις δεσμεύσεις της υπό το διεθνές δίκαιο και ανθρωπιστικό δίκαιο η ΕΕ. Ή σεβόμαστε τα ανθρώπινα δικαιώματα ή όχι. Αν επιστραφούν αυτοί, πηγαίνουν στη Λιβύη και καταλήγουν σε αυτή την κατάσταση. Χωρίς να σεβόμαστε τα, το διεθνές δίκαιο και τις υποχρεώσεις μας, ε, πρέπει να αρθούμε στο ύψος των περιστάσεων. Υπάρχουν ευθύνε. Δεν έχουμε σχεδόν πληροφορίες. Πότε και πώς έγινε αυτό. Στη συγκεκριμένη τοποθέτηση. Ποιος επέστρεψε αυτά τα άτομα στη Λιβύη. Ποιος τους έστειλε πίσω εκεί. Ε, λοιπόν, αυτά τα ερωτήματα θα πρέπει να απαντηθούν. Θα πρέπει να διατυπωθούν στην Ιταλική κυβέρνηση Αφενό και στην Frontex αφετέρου. Πρέπει να συζητηθεί περαιτέρω και περισσότερο αυτό το είναι σημαντικό. Υπάρχουν νομικά προβλήματα. Πρέπει να πάμε στην ε, Επιτροπή αυτή και ε, να καταβάλουν τις απόψεις τους και οι της Frontex και οι της Ιταλικής κυβέρνησης. Ο επόμενος αγορητής, δύο λεπτά παρακαλώ. Η κυρία Μπορσελίνο. Για μια ακόμη φορά Θα επαναλάβω ότι ζήτησα πολλές φορές πληροφορίες για αυτή τη συμφωνία με τη Λιβύη και για αυτή τη συμφωνία κανένας δεν μας μιλάει, κανένας δεν μας απαντάει. Και μιλάμε για μια χώρα για σαν τη Λιβύη, άκουσα διάφορους εφημισμούς σήμερα. Μίλησα ας πούμε για κοινωνική ωφέλεια εργασίες, μα εγώ δεν έχω καμιά εμπιστοσύνη. Τι θα πει αυτό ας πούμε στην ε, Λιβύη θα μπορούσε να ερμηνευτεί ναι. ως καταναγκαστική εργασία. Ρύθμιση των μεταναστευτικών ροών σημαίνει ξαναστέλνω όλο αυτόν τον κόσμο στην έρημο και τους εγκαταλείπω εκεί. Μιλάμε για τη Λιβύη που δεν υπέγραψε καμία σύμβαση. Δεν έχει υπογράψει ποτέ τη σύμβαση της Γενέβης. Λοιπόν πρόκειται για έναν συνομιλητή που πρέπει να τον παίρνει κανείς με τα τσιμπιδάκια. Θέλω να πω το εξής, ότι με τη συνθήκη της Λισαβόνας ε, το Κοινοβούλιο ε, καλείται να, να, να δώσει τη συνένεσή του για τη Συμφωνία Επανεισδοχής και σύμφωνα με το άρθρο 218 της συνθήκης πρέπει να ενημερωνόμαστε άμεσα και πλήρως. Πρέπει λοιπόν να είμαστε και εμείς ε, πληροφορημένοι και ζητώ η Κομισιόν να έρχεται να μας αναφέρει εδώ για τις διαπραγματεύσεις σε τακτικά χρονικά διαστήματα και από κοινού με την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων και τις αντιπροσωπίες ε, για τις σχέσεις με το Μαγκρέπ και τη Λιβύη. Θα ήταν μια χειρονομία καλής θέλησης. Αν εμείς θέλουμε να καταλήξουμε σε ένα πραγματικό συμπέρασμα, δηλαδή ε, στο τι θέλουμε που είναι να διασφαλίσουμε τα δικαιώματα των ανθρώπων πρέπει να κάνουμε να χρησιμοποιήσουμε όλα τα μέσα που έχουμε στην διάθεσή μας και όσο το δυνατόν πιο γρήγορα. Μιλήσαμε για 400, μιλήσαμε για 240, αλλά ξέρουμε ότι ο αριθμός είναι πολύ μεγαλύτερος, δεν ξέρουμε ακριβώς πόσο, πόσοι είναι και φυσικά στα κέντρα που πήγαμε ε, μας έδειξαν αυτά τα οποία θέλανε αυτοί να δούνε να δούμε και όχι αυτό που έπρεπε να δούμε. Δύο λεπτά η κυρία Αντζελίλη. Φυσικά η ανησυχία υπάρχει και εγώ την συμμερίζομαι μαζί με τους συναδέλφους ανησυχία για τα ανθρώπινα δικαιώματα και την μεταχείριση. Αλλά σήμερα όμως ακούσαμε και θετικά νέα. Ας πούμε ε, την διάθεση της Λιβύης να ξαναδεχθεί την παρουσία της ΥΠΑ της αρμοστίας για τους πρόσφυγες. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Μία ερώτηση όμως που θέλω να την κάνω στον κύριο Παντζέρη. Διότι ο κύριος Παντζέρη, αν κατάλαβα καλά, είπε στην αρχή ότι η Κομισιόν ε, πολλές φορές είπε ότι οι διμερείς συμφωνίες παρακολύουν την άσκηση ευρωπαϊκών πολιτικών. Και εδώ εγώ διαπιστώνω μία ε, κρυφή κριτική σε αυτούς που συνάπτουν τις συμφωνίες στην προκειμένη περίπτωση την Ιταλία και όχι μόνο. Μα οι παραμεθόριες χώρες ε, κάνουν συνάπτουν συμφωνίες γιατί κανένας άλλος δεν τις συνάπτει. Λένε έχουμε ελάχιστη Ευρώπη για τις μεταναστευτικές πολιτικές και ο καθένας κάνει ό,τι μπορεί. Και εμείς περάσαμε ένα πρωινό σήμερα με την Βελγική Προεδρία ζητώντας μία κοινή ευρωπαϊκή προσέγγιση. Το έπανε και ο κύριος Μπουσουτή και ο κύριος Γιαρβολίνο. Και ζητήσαμε <coughs> να υπάρχει ένας να υπάρχει μία ενορχίστρωση, μία ευρωπαϊκή ενορχήστρωση ε, για αυτές τις συμφωνίες που να εγγυάται τις συμφωνίες από όλες τις πλευρές και τα κράτη-μέλη να, έχουν τις εγγύησεις τους αλλά και ε, να έχουν τις εγγύησεις τους και οι αιτούντες άσυλο. Ο κύριος Μποργκέτσιο δύο λεπτά. Εξεπλάγιν κύριε Πρόεδρε διότι το θεώρησα γκροτέσκο. Δηλαδή ότι τελικά ας πούμε είναι μανία ορισμένων χωρών να έχουν σχέσεις με τη Λιβύη. Από όλες τις συζητήσεις όμως που άκουσα με ποιον θα πρέπει να συνάψουν σχέση, διότι γνωρίζουμε πολύ καλά ποια είναι τα προβλήματα στη Μεσόγειο θάλασσα, εφόσον τα προβλήματα ε, προερχόταν από, τις, ε, από τη Λιβύη από τις ακτές της Λιβύης. Λοιπόν, αξιέπαινε η Ιταλία που κατάφερε να πείσει τη Λιβύη να συνάψει μία πρώτη συμφωνία. Άρα εμείς διευκολύνουμε την Ευρώπη, δεν την παρακολύουμε, διότι καταφέραμε να διαπραγματευτούμε. Και εγώ δεν έχω στοιχεία να το πω, αλλά πιστεύω ότι είναι απόλυτα λογικό να το λέμε, ότι αν έφτασε εκεί ξανά η ύπατη αρμοστία. Αυτό έχει να κάνει και με την διπλωματία και τις ε, πιέσεις των χωρών εκείνων που για τη μετανάστευση δεν περιορίζονται στο μπλα μπλα του κοινοβουλίου αλλά πραγματικά με, μεγάλη, με μεγάλες ε, δυσκολίες ε, και πιέσεις προσπαθούν να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα πόσο μάλλον να διαπραγματεύονται και με γραφικές προσωπικότητες σαν τον ηγέτη της Λιβύης το πρόβλημα των Αφρικανών προσφύγων imprimής είναι, μία, είναι ένα πρόβλημα της Αφρικής. Λοιπόν, εδώ ακούστηκε ότι πρέπει να γίνουν να ασκηθούν πιέσεις στις χώρες που έχουν συνάψει συμφωνίες. Μα η Λιβύη έχει υπογράψει μια Αφρικανική συμφωνία για τους πρόσφυγες και πάση περιπτώσει θα πρέπει η Λιβύη να τα βρει με την Αφρική γιατί δική της συγγενής είναι οι Αφρικανοί. Οι Αφρικανοί πρέπει να τα βρούνε μεταξύ. Ευχαριστώ κύριε Σπουσούτη. δύο λεπτά. Νομίζω έχει κάποιο δίκιο η Λιβύη όταν λέει ότι δεν έχει κάποια φιλοδοξία να είναι ο νότιος συνοριοφύλακας της Ευρώπης. Έχει κάποιο δίκιο όταν λέει ότι δεν βοηθάει επαρκώς η Ευρώπη. Και έχει κάποιο δίκιο όταν λέει ότι έχει τεράστια προβλήματα με τα νότια σύνορά τη η Λιβύη. Το γνωρίζουμε αυτό εδώ και αρκετά χρόνια και ρωτώ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τον κύριο Μάσελ ε, ιδιαίτερα τι αναμένει, τι περιμένει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να βοηθήσει τη Λιβύη ώστε η Λιβύη να μπορέσει να βοηθήσει εμά στη συνέχεια. Δεν έχει δοθεί η απάντηση μέχρι στιγμή, δεν ήταν ικανοποιητική μέχρι στιγμή. Τι περιμένει ο κύριο Μπαρόζο να πάει στη Λιβύη και να μιλήσει με την κυβέρνηση τη Λιβύη. Καλωσορίζω πολύ το γεγονός ότι μίλησε με τον Υπουργό Εξωτερικών της Λιβύης. Αλλά από το Φεβρουάριο γιατί δεν πήγε ακόμα στην Τρίπολη, την πρωτεύουσα της Λιβύης ακόμη. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πιστεύω πολλά περισσότερα ακόμα πρέπει να κάνει με τη Λιβύη. Επιτόπου, εκεί επιτόπου. Αν θέλουμε να συνεργαστεί η Λιβύη μαζί μας, πρέπει εμείς να είμαστε πρόθυμοι να συνεργαστούμε με τη Λιβύη για τις συμφωνίες. Τις επικρίσεις που έγιναν τις επικριτικές παρατηρήσεις για τις διμερείς συμφωνίες τις λαμβάνω υπόψη με πολλές επιφυλάξεις για διάφορους λόγους. Πρώτον, οι διμερείς συμφωνίες έχουν περιορίσει τη ροή παράνομης μετανάστευσης σημαντικά και αυτό όχι μόνο βοήθησε τα νότια κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης που μέχρι σήμερα επομιζόντουσαν αυτά τα βάρη μόνα τους αλλά έσωσε τη ζωή εκατοντάδων ατόμων που κάθε χρόνο πνιγόντουσαν στην Μεσόγειο χωρίς να μπορέσουν να ε, βοηθηθούν. Δεύτερον, οι διμερείς συμφωνίες ήταν το πιο αποτελεσματικό όπλο κατά του οργανωμένου εγκλήματος που βρίσκεται πίσω από όλες αυτές τις αναχωρήσεις από την Αφρικανική ακτή προς την Ευρώπη. Δεν είδα άλλη καλύτερη πρωτοβουλία να επιτεθούμε και να αντιμετωπίσουμε το οργανωμένο έγκλημα παρά αυτό όσον αφορά τις οργανωμένες αυτές κινήσεις. Είναι πολύ εύκολο, τελευταία παρατήρηση, να ασκεί κανείς επικρίσεις επί των διμερών συμφωνιών. Είναι εύκολο να είναι να είναι εναντίον κανεί. Αλλά πρέπει να αποφύγουμε να πέσουμε στην παγίδα τη υποκρισία και να είμαστε υποκριτέ. Διότι αυτοί που ασκούν επικρίσεις σε αυτέ τι συμφωνίε δεν έχουν απάντηση να δώσουν ποιο, στο ερώτημα ποιο θα επομιστεί τι ευθύνε ε, για αυτού του ετούντε άσυλο και του πρόσφυγες που θα έρθουν στην Ευρώπη. Θέλουμε να έρθουν στην Ευρώπη αλλά να μείνουν στην Ιταλία, Ισπανία, Ελλάδα, Μάλτα και στα νότια κράτη τη Ευρωπαϊκή Ένωση μόνο. Ε, αυτό δεν είναι το αποδεκτό. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ο κύριος Παντσέρη αναφέρθηκε σε συγκεκριμένα σημεία. Είναι λοιπόν δίκαιο να ακούσουμε την απάντησή του. Λοιπόν, έχει τον λόγο για μισό λεπτό και μετά θα επανέλθουμε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στον κύριο Μανσερβίση για το τελικό σημείο. Έχετε τον λόγο κύριε Παντσέρη. Εγώ ανέφερα εδώ μια άποψη ε, και μια κρίση που είναι και της ε, Κομισιόν ότι πολλές φορές οι διμερείς συμφωνίες παρακολύουν την ευρωπαϊκή δράση. Τώρα απ' την άλλη και εγώ είμαι απόλυτα πεπισμένος ότι άμα δεν υπάρχει ευρωπαϊκή πρωτοβουλία τότε εντάξει διμερείς συμφωνίες αλλά δεν πρέπει να είμαστε υποκριτές και πρέπει να ξέρουμε ότι πολλές χώρες που έχουν αυτές τις διμερείς συμφωνίες πιστεύουν ότι έχουν λύσει όλα τα προβλήματα μέσα από τις διμερείς συμφωνίες. Αυτή είναι η συμπεριφορά πολλών από τις χώρες που έχουν συνάψει τις διμερείς συμφωνίες. Και αν ζητάμε, όπως το είχα ζητήσει και εγώ, μια ευρωπαϊκή παρέμβαση σε αυτόν τον τομέα, τότε θα πρέπει να υποστούμε την ευρωπαϊκή πολιτική. Δεν μπορούμε να παίζουμε κρυφτούλη. Διότι άμα η ισχύει ήδη με τις συμφωνίες τότε θα πρέπει να τις ε, αναλάβουμε μέχρι τέλους και άμα έχουμε τέτοιου είδους ε, απελάσεις τότε θα πρέπει να τις, ε, να τις χωνέψουμε και αυτές. Ε, άμα έχουμε όμως Ευρωπαϊκή Συμφωνία θα πρέπει να υποστούμε την Ευρωπαϊκή Συμφωνία. Δεν υπάρχει εσωτερική αντίφαση. Απλώς λέω ότι είναι σημαντικό να σμπρώξουμε ούτω ώστε να, να ληφθεί μία ευρωπαϊκή πρωτοβουλία. Ο κύριος Μασεβίση. Λοιπόν, να απαντήσω για μια φορά στη γλώσσα μου, ε, γιατί συνήθω συνήθως μιλάω στα αγγλικά. Α, συνεχίζω στα αγγλικά. Αν μιλάμε για στοιχεία γιατί υπάρχουν πολλά πράγματα και σχόλια που, με τα οποία συμφωνώ προσωπικά και η Επιτροπή, μερικώς τουλάχιστον. Όμως, αν μιλάμε για στοιχεία, πρόκειται για 400 ή 250 άτομα περιπτώσει μιλάμε για άτομα που βρίσκονται αυτή τη στιγμή στη Λιβύη χωρίς να υπάρχουν αναφορές ότι έχουν επιστραφεί. Δεν υπάρχουν στοιχεία τέτοια ότι έχει γίνει επιστροφή τους προς την Λιβύη. γιατί δεν θεωρούμε ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις για κάτι τέτοιο. Μιλάμε λοιπόν για μια ομάδα ατόμων που αυτή τη στιγμή βρίσκονται στη Λιβύη και πρέπει να αντιμετωπίσουμε την κατάσταση με βάση το διεθνές δίκαιο και την πολιτική μας σχέση με τη Λιβύη. Και αναφέρομαι στην πολιτική σχέση γιατί δεν έχουμε κάποιο νομοθετικό κείμενο με την Λιβύη που να αντακαλύπτει αυτά τα θέματα. Άρα λειτουργούμε με βάση τις πολιτικές σχέσεις και το διεθνές δίκαιο. Δεύτερον, όσον αφορά την διμερή συμφωνία. Προσωπικά θα χρησιμοποιούσα μία πολύ ρεαλιστική προσέγγιση θα έλεγα ότι μια ευρωπαϊκή συμφωνία είναι σαφώς καλύτερη από μια διμερή και λύνει πολλά προβλήματα μεταξύ των οποίων και της αλληλεγγύης. Όμως έχει αποδειχθεί αποτελεσματική αυτή η συμφωνία καθώς μετά την έναρξη ισχύω αυτής της ε, συμφωνίας συνεργασίας έχουν σταματήσει οι ροές, ε, μεταναστών από τη Λιβύη προς την Ιταλία. Και αυτή η συμφωνία εναρμονίζεται με το κοινοτικό κεκτημένο. Βέβαια υπάρχει και ένα απόρριτο τμήμα, το οποίο δεν γνωρίζουμε. Και υπάρχει και το θέμα εδώ ότι δεν γνωρίζουμε πού συνελήφθησαν αυτά τα άτομα. Δεν μπορούμε λοιπόν να πούμε ότι η Ιταλία είναι υποχρεωμένη να κάνει περισσότερα από τους υπόλοιπους. Δεν γνωρίζουμε που συνελήφθησαν αυτά τα άτομα. Τώρα, όσον αφορά την μεταχείρισή τους αυτή τη στιγμή στη Λιβύη, θέλουμε να διασφαλίσουμε ότι γίνεται με τρόπους που συμβαδίζουν με την πολιτική μας. Τι πρέπει να ξέρουμε λοιπόν και τι πρέπει να κάνουμε. Καταρχάς, ε, συμφωνία συνεργασίας υπάρχει ένα κεφάλαιο που μέχρι στιγμής ε, δεν είχε παράξει τίποτα και γι' αυτό μάλλον δεν το γνωρίζει και ο συνάδελφος που αφορά αυτό ακριβώς. Το είπα και προηγουμένως. Στη συνεδρίαση που είχαν ε, η κυρία Μάλστρομ και ο κύριος Μουσακούσιλ αποφάσισαν να ξεκινήσουν συζητήσεις επί του κεφαλαίου αυτού. Θα ζητήσω συγγνώμη λοιπόν στην κυρία Πορσελίνο που δεν απάντησα χτες. Όμως, τώρα ξεκινάμε. Η κυρία Μάλστρομ θα ξεκινήσει τις διαπραγματεύσεις στη Λιβύη και βεβαίως είναι υποχρέωσή μας να σας ενημερώνουμε και για τις εξελίξεις. Άρα η κατάλληλη προσέγγιση είναι να έχουμε ένα καλό κεφάλαιο για τις εσωτερικές υποθέσεις στη συμφωνία με τη Λιβύη. Αυτό δεν θα καλύπτει μόνο το θέμα της επανεισδοχής, όπως γίνεται και με τις άλλες συμφωνίες μας. Θα καλύπτει και θέματα όπως σεβασμός ανθρωπίνων δικαιωμάτων κτλ. Τώρα, όντως δεν έχει επικυρώσει την σύμβαση της Γενέβης η Λιβύη, αλλά έχει υπογράψει τη σύμβαση του 1955, που πάνω κάτω τη δεσμεύει για τα ίδια πράγματα, μεταξύ των οποίων και συνεργασία με την ύπατη αρμαστία του ΟΗΕ. Τώρα, τι άλλα εργαλεία έχουμε. Έχουμε την κοινή στρατηγική Ευρώπης-Αφρικής. Υπάρχει η Σύνοδος Κορυφής Ευρώπης-Αφρικής φέτος τον Νοέμβριο. Αυτά μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να υπενθυμίσουμε στους φίλους μας από τη Λιβύη ότι έχουν υποχρεώσεις και στα πλαίσια των Αφρικανικών Συμβάσεων που καλύπτονται από την στρατηγική σχέση Ευρωπαϊκής Αφρικής. Όλα αυτά λοιπόν ισχύουν και το καλύτερο που μπορούμε να κάνουμε αυτή τη στιγμή είναι να κάτσουμε κάτω και να διαπραγματευτούμε με τη Λιβύη έτσι ώστε αυτά που αναφέρονται στην κοινή συμφωνία να χρησιμοποιηθούν ως πλαίσιο για ευρωπαϊκή δράση. Και επιπλέον υπάρχει και δυνατότητα να γίνει συζήτηση για το πώς μπορούμε να βοηθάμε τους ετούντες άσυλο για μεταχείριση με βάση τους κανόνες μας. Επαναλαμβάνω όμως αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει νομοθετικό πλαίσιο για όλη αυτή τη διαδικασία, άρα όλα γίνονται σε επίπεδο πολιτικών επαφών με στόχο να υπάρξει σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ας μην τα ξεχνάμε λοιπόν όλα αυτά. Αυτά πάνω κάτω έχω να πω να πω ότι δεν θα διακόψουμε το διάλογο μας με τη Λιβύη. Τώρα ελευθερώθηκαν και είναι αλήθεια ότι η απελευθέρωση 3.000 ατόμων είναι πρόβλημα. Πρόεδρο, σας ευχαριστούμε και για την, τον συνοψισμό στι ερωτήσει που έγιναν. Έχουμε ένα τέταρτο ακόμα, έχουμε ένα πρόσθετο σημείο που είναι ο προπολογισμό στην ημερησία διάταξη. Και έχουμε και του διερμηνεί ε, που θα ολοκληρώσουν στι 6.30. Έχουμε αυτά τα θέματα. Κάνω ό,τι μπορώ για να μην περικόψω τη δυνατότητα να αναφερθείτε σε κάποια σημεία στην Επιτροπή ΛΥΜΠΕ. Σε μισό λεπτό ο καθένας όμως παρακαλώ να παρέμβετε. Κοντσέτα παρακαλώ. Πέρα από το θέμα των δικαιωμάτων, υπάρχει ένα πρόβλημα και θέλω να ξέρω τη γνώμη σας Η Λιβύη έχει αναλάβει ένα ρόλο διεθνούς ε, αστυνομικού που κανένα δεν τη έχει αναθέσει. Διότι το να συλλαμβάνει τα πλοία σε διεθνή ύδατα κανένα δεν τη το Δεν, δεν, το ανέθεσε. Εντάξει, το καταλαβαίνω ότι άμα πιάσω κάποιον που θέλει να περάσει τα σύνορα, εντάξει, προστατεύω την κυριαρχία τη χώρα μου. Αλλά εδώ το λιβικό κράτο παίζει ένα ρόλο διεθνούς αστυνομίας που δεν μπορεί να τον παίξει ούτε βάσει των διεθνών συμφωνιών. Διότι κανένας δεν δίνει το δικαίωμα στην Ιταλία ή τη Λιβύη να συνάπτει διεθνείς συμφωνίες που να αφορούν στα διεθνή ύδατα. Ούτε η Ευρώπη μπορεί να το κάνει. Ο κύριος Ταβάρες. Είπαμε, μια και δεν ξέρουμε πού συνελήφθησαν αυτοί, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα παραπέρα. Τα κράτη-μέλη που συνεργάζονται με τη Frontex έχουν επίσης ευθύνε να συνεργάζονται με τη διάθεση πληροφοριών. Ζητώ από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μας πούν και να μάθουμε ακριβώ. πότε συνέβη, πού, τι και ή δυνατόν με τις συντεταγμένες πλάτους και μήκους με το GPS και αν γίνεται και να το, να το δούμε αυτό και με την βοήθεια της πολιτικής μου ομάδας να ζητήσουμε η Frontex να προσέρθει εδώ και να κάνει λόγο για αυτά τα πράγματα διότι δεν γνωρίζουμε τι έχει συμβεί και αυτό δεν μπορεί να βοηθάει. Πρόεδρος, είχαμε μια συζήτηση εδώ και από τη Γενική Διεύθυνση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έχει ζητηθεί να ληφθούν υπόψη αυτά τα σχόλια και οι παρατηρήσεις και ή δυνατόν να απαντηθούν αυτές οι ερωτήσεις γραπτός ώστε να προσχωρήσουμε στο επόμενο σημείο. Σας ευχαριστούμε λοιπόν και έτσι πιεζόμαστε να βιαστούμε και να περάσουμε στο τελικό τελευταίο σημείο της ημερήσιας διάταξης σήμερα. Απόψε, αυτό το απόγευμα δηλαδή με άλλα λόγια, που είναι αυτό το σημείο Διακόπτει ο Πρόεδρος. Το σημείο 15 λοιπόν είναι αυτό, ναι. Το σημείο που αφορά την θέση παρουσίαση της γνωμοδότησης ε, όσον αφορά το Κοινοβούλιο για το σχέδιο προϋπολογισμού του 2011. Εγώ είμαι ο σύνταξη γνωμοδότησης για αυτή τη γνωμοδότηση. Θέλω να ευχαριστήσω τους τους εισηγητές. Είχαμε μια γόνιμη συζήτηση. Καθορίσαμε την πορεία που θα ακολουθήσουμε. Όμως το σχέδιο γνωμοδότησης έχει διανεμηθεί και τώρα αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι νομίζω καλό θα ήταν αν ακούγαμε από το Συμβούλιο πρώτα τις απόψεις του και μετά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε, στα λιγότερα από 15 λεπτά που έχουν απομείνει για να κλείσει η συνεδρίασή μας. Παρακαλώ λοιπόν, ο εκπρόσωπος του Συμβουλίου πρώτα, αν θέλετε να τοποθετηθείτε, να εκφράσετε τις απόψεις σας, παρακαλώ. Τις ε, απόψεις του Συμβουλίου, λέω για τον προϋπολογισμό του 2011. Έχετε τον λόγο λοιπόν. Παρακαλώ το Συμβούλιο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Το Συμβούλιο για, το 2000, για τον ε, προπολογισμό 2011 χρειάστηκε να λάβει η Κομισιόν δύσκολες ε, αποφάσεις. Έχουμε ένα κλίμα ιδιαίτερα μπερδεμένο πιέσεις από τα διάφορα κράτη για να μειωθούν οι δημόσιες δαπάνες. Αυτό λοιπόν ισχύει και για τον ε, ευρωπαϊκό προϋπολογισμό. Τώρα για τον τίτλο πρέπει να σας πω ότι αυτό το οποίο έχει γίνει μέχρι τώρα έγινε ιδιαίτερα συγκρατημένα και μετρημένα. Δηλαδή αν φανταστεί κανείς όλες τις άλλες ε, περικοπές ε, ε, στον προπολογισμό για τις άλλες πολιτικές δηλαδή. Τώρα, για τις πιστώσεις πληρωμών βασιστήκαμε στο ποσοστό εκτέλεσης και των πράξεων, των εκτελεστών πράξεων στα πλαίσια του οικονομικού έτους 2009-2010. Ξέρουμε ότι αυτός δεν ήταν ο καλύτερος τρόπος ε, να φτιάξει κανείς ε, προϋπολογισμό, δηλαδή να εργαστεί στο επίπεδο εκτέλεσης μόνο αλλά έπρεπε να λάβουμε υπόψη ότι έχοντας ένα νέο πλαίσιο επεξεργασίας του προϋπολογισμού η δημοσιονομική συζήτηση θα γίνει όταν θα έχουμε συναλλαγή και εναρμόνιση μεταξύ Κοινοβουλίου και Συμβουλίου. Υπήρξε λοιπόν μία σχετική συγκράτηση ε, για τον τρόπο με τον οποίο με τον οποίο τοποθετηθήκαμε στο Συμβούλιο. Άμα πάρουμε τώρα το σύνολο του τίτλου, πιστώσεις υποχρεώσεων έχετε 11,7% αύξηση στις ε, πιστώσεις ε, πληρωμών έχετε μία μείωση για ένα τμήμα που δικαιολογείται από τα επίπεδα εκτέλεσης. Αυτά μπορώ να πω σε αυτή τη φάση επεξεργασίας του προϋπολογισμού. Η θέση αυτή του Συμβουλίου είναι μια πρώτη προσέγγιση σε μια συζήτηση που πρέπει να συνεχίσει. Ευχαριστώ. Ο κύριος Φερκέρεν. Α, συγγνώμη. Η κυρία Μονίκ Παγάντε εκ μέρους της Κομισιόν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ και την Βελγική Προεδρία για αυτές τις διευκρινήσεις. Θα ήθελα να εκφράσω την λύπη μου για τις περικοπές ε, του Συμβουλίου. Άκουσα αυτά που είπε ο προλαλή ότι βασιστήκανε στο ποσοστό εκτέλεσης των ετών 2009-2010. τα προγράμματα όμως έχουν ήδη και αρχίσουν και τρέχουν και έχουν αρχίσει να εφαρμόζονται σωστά οπότε με αυτές τις περικοπές θα έχουμε μεγάλα προβλήματα κυρίως για την τεχνική βοήθεια των προγραμμάτων που αφορούν στις δύο γενικές διευθύνσεις ανθρώπινα δικαιώματα και δικαιοσύνη. Θέλω να επιστήσω λοιπόν την προσοχή σας ότι αυτές οι περικοπές μέσα στα πλαίσια της τεχνικής βοήθειας θα έχουν σημαντικές επιπτώσεις. Παράδειγμα, εφαρμογή της πρόσφασης συμφωνίας για το TFTP όπου θα μπορούσαμε να χρηματοδοτήσουμε τα μέτρα βάση του άρθρου 4 και 12, το ίδιο και για τους οργανισμούς. Και εδώ ο προϋπολογισμός μας υπολογίστηκε λαμβάνοντας υπόψη τα αιτήματα των οργανισμών. αλλά προχωρήσαμε σε περικοπές από μόνοι μας. Αυτοί οι περιττέρω περικοπές όμως ε, θα δημιουργήσουν προβλήματα λειτουργίας στους οργανισμούς. Η Europol σύμφωνα με το FTP θα έχει μεγαλύτερες αρμοδιότητες και η λειτουργία της θα επιβαρυνθεί. Νομίζω ότι θα πρέπει να το σκεφτούμε πολύ καλά το θέμα. Καταλαβαίνω τις ανάγκες δημοσιονομικών περικοπών, τα προβλήματα των εθνικών προϋπολογισμών, αλλά εγώ θέλω να συνεχίσουμε τις πολιτικές και νομικές δεσμεύσεις που η Ευρωπαϊκή Ένωση δεσμεύθηκε να προχωρήσει στα θέματα εσωτερικών υποθέσεων και δικαιοσύνης. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ. Ε, και όπως είπα πιο πριν, σε σχέση με μια συνάντηση για τον καθορισμό των προτεραιοτήτων, θεμελιδών προτεραιοτήτων υπό το πρίσμα της ε, δικής μας Κοινοβουλευτικής Επιτροπής, Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών για τα πιλωτικά προγράμματα και τις προκατακτικές δράσεις. Έχουμε χρόνο για να καταθέσουμε τις προτάσεις ε, μέσα στη διαδικασία κατάθεσης τροπολογιών που έχουμε μπροστά μας. Όμως, ζήτησα να διανεμηθούν ε, το σχέδιο γνωμοδότησης ε, ε, σύντομο ως ήθιστε σε σχέση με τέτοιου είδους έγγραφα να, που πρέπει να ληφθούν υπόψη από την Επιτροπή Προϋπολογισμών και ακόμα μπορούμε νομίζω να ακούσουμε κάποιες απόψεις από πλευράς των μελών της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής. Μια και σήκωσε το χέρι η κυρία Κέλλερ για παράδειγμα. Αν θέλετε να λάβετε τον λόγο και η κυρία συνάδελφος Χιμένες και μετά ο άλλος συνάδελφος, εσείς κυρία Κέλλερ, έχετε τον λόγο. Ευχαριστώ. Για το σχέδιο γνωμοδότησης λοιπόν, θα έλεγα δεν είναι μόνο ένα θέμα να έχουμε περισσότερα κονδύλια υπό το σωστό τίτλο, στη σωστή κατηγορία. Το, θέμα, το πρώτο θέμα είναι πώς θα δαπανηθούν και για ποιο σκοπό τα κονδύλια. Και τα περισσότερα κονδύλια έχουν έλλειψη αιτιολόγησης. Θα είναι αναγκαίο λοιπόν σε σχέση με τη δημιουργία ενός κονδυλίου να δημιουργεί κανείς ένα κονδύλιο Ψ, μέγα, αλλά το θέμα του πώς θα διατεθούν και για ποιο σκοπό θα διατεθούν αυτά τα κονδύλια είναι σημαντικό. Θα ήθελα λοιπόν περισσότερες επεξηγήσεις να δοθούν. Ελπίζω ότι θα δοθούν αυτά τα στοιχεία ευελπιστώ και να δούμε περισσότερο την ποιότητα παρά την ποσότητα και να δούμε ότι σε σχέση με μία άκρηση κάποιου κονδυλίου σε κάποια κατηγορία αυτό δεν λέει και τόσα πολλά πράγματα μόνο του. Και τώρα έγκαιρα διάθεση σωστών πληροφοριών για το θέμα του συστήματος IT ή το ένα ή το άλλο. Συμφωνώ πολύ επ' αυτόν. Από την άλλη όμως πλευρά πώς μπορούμε να συμφωνήσουμε για ένα προϋπολογισμό που δίνει 20-30 εκατομμύρια ευρώ στο ΣΥΣ 2 το οποίο δεν υφίσταται. Και έτσι θα ήθελα λοιπόν να έχω έγκαιρα, κατά λεπτός εξειδικευμένα τις πληροφορίες για αυτά τα στοιχεία, προτού ψηφίσουμε, ώστε να γνωρίζουμε τι γίνεται και να έχουμε ε, σαφή επιμερισμό των ευθυνών. Είχατε πει ότι θα ζητούσατε για τις πληροφορίες πώς αυτά τα κονδύλια δαπανώνται και από το ελεγκτικό συνέδριο θα έλεγα Ελπίζω ότι θα υπάρχουν κάποια στοιχεία επ' αυτού ήδη τώρα. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Η κυρία Χιμένες παρακαλώ. Ε, ευχαριστώ Πρόεδρε. Σχετικά με το πρόγραμμα πρόληψης, διαχείρισης και λοιπά των επιπτώσεων της τρομοκρατίας βλέπω ότι έχετε μια αύξηση και αυτό γιατί αυξάνονται και οι αρμοδιότητες στον τομέα της δικαιοσύνης μετά από τη συνθήκη της Λισαβόνας. Ρωτώ, θεωρείτε ότι φτάνει αυτή η αύξηση ούτως ώστε να καλυφθούν όλες οι ανάγκες που θα έχουμε μετά την εφαρμογή της Λισαβόνας. Άμα λάβει κανείς υπόψη του όλα τα προγράμματα, θα έλεγα ότι για την προετοιμασία και την πρόληψη για την αντιμετώπιση των τρομοκρατικών επιχειρήσεων το πεδίο είναι πάρα πολύ μεγάλο και ανησυχώ δηλαδή για το κατά πόσο αυτό το ποσό μπορεί να καλύψει τα πάντα. Και αναρωτιέμαι αν θα συνεχίσουμε έτσι να προστατεύουμε τα θύματα της τρομοκρατίας. Υπάρχει ένα δίκτυο, ευρωπαϊκό δίκτυο για τα θύματα της τρομοκρατίας και αρχίζει να αντιμετωπίζει προβλήματα ως προς τη χρηματοδότηση για την κοινωνική, ψυχολογική βοήθεια λοιπά των θυμάτων θα καλυφθούν όλες αυτές οι ανάγκες. Ευχαριστώ. Κύριος Βάντερ Κάμπ. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Τέσσερα σύντομα σχόλια. Μια γνωστή Ολλανδική παροιμία λέει μην πουλήσει το τομάρι της αρκούδας προτού την σκοτώσει. Είναι σημαντικό και είναι ίσως ε, αυτό σε σχέση με τη δουλειά που έχουμε μπροστά μας να το λάβουμε υπόψη. Το επόμενο διάστημα πρέπει να προσπαθήσουμε να δεχθούμε το νόημα αυτής της παροιμίας. Συμφωνώ με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι εκείνα τα προγράμματα που με καθυστέρηση ξεκίνησαν δεν θα πρέπει να πέσουν θύματα περικοπών και συμφωνώ με την κυρία Κέλλε στην παρατήρηση Χρειαζόμαστε σε κάποια από αυτά τα σημεία περισσότερες πληροφορίες. Αν κάποια επιμέρους κονδύλια με τα προγράμματα αυτά ξεκινούν να λειτουργούν υστερότερα με καθυστέρηση, δεν μπορούν να περικόπτονται στη συνέχεια και έτσι να θυσιάζονται. Πρόκειται για το 2009-2010 και εδώ είναι δυνατόν να ε, υπάρχουν κάποιες ε, περικοπές, ε, όμως δεν είναι λόγος για περικοπές το ότι καθυστέρησαν αυτά τα προγράμματα προγράμματα και θα πρέπει πιο συγκεκριμένα να ληφθούν όλα αυτά υπόψη. Ξέρω φυσικά ότι η Κοινοβουλευτική Επιτροπή ΛΥΜΠΕ δεν εκπροσωπεί τα δικά της συμφέροντα στο ψήφισμα, αλλά μία σύντομη αναφορά στο πρόγραμμα της Στοκχόλμης, στην Ευρωπόλ. Αυτά είναι πράγματα τα οποία σίγουρα θα μπορούμε να παρουσιάσουμε. Δεν μπορούμε ως Ευρωκοινοβούλιο να εγκρίνουμε ένα τεράστιο πρόγραμμα Στοκχόλμης και στη συνέχεια να μην μεριμνούμε με κανένα τρόπο να πρικοδοτήσουμε Υποδοτείται επαρκώς από πλευράς κονδυλίων. Και γι' αυτό τον λόγο έθεσα το ερώτημα. Μήπως την πρόταση αυτή σε κάποια σημεία θα έπρεπε να την εξετάσουμε από πιο κοντά πρόγραμμα στο Κόλμης, Ευρωπόλ και υπάρχει ένα τρίτο σημείο. Αυτή τη στιγμή το ξέχασα, ελπίζω να το θυμηθώ υστερότερα. final point. Για μια τελική τελευταία παρατήρηση, θα θέλαμε να ξανακούσουμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ίσως να έχουμε μια σύντομη απάντηση επ' Και αν μπορείτε να μας ε, ε, δώσετε αυτή τη δυνατότητα για ένα επιπλέον λεπτό, να έχουμε ένα σύντομο σχόλιο για τις ερωτήσεις που σας διατυπώθηκαν. Υπήρξαν κάποια σχόλια όσον αφορά την δυνατότητα αύξησης του προγράμματος που αφορά την καταπολέμηση της τρομοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ίσως να τοποθετηθείτε σε αυτό το σημείο, να δώσετε προσοχή σε αυτό το σημείο πρωτού αυτή τη συζήτηση. Ευχαριστώ. Σημειώνω την επιθυμία σας να έχετε περισσότερες πληροφορίες ε, για τις διακοιμάσεις του προϋπολογισμού. Σας υπενθυμίζω ότι στα activity statements ε, στον προϋπολογισμό υπάρχουν ε, αναφορές στις διακυμάνσεις ε, των πιστώσεων. Ίσως είναι δύσκολο να τα διαβάσετε αυτά τα έγγραφα, αλλά εκεί αναφέρονται συγκεκριμένες πληροφορίες και βεβαίως μπορούμε να τις συμπληρώσουμε είτε σε διμερείς συζητήσει είτε γραπτός όσον αφορά τις διακυμάνσεις των πιστώσεων. Τώρα, όσον αφορά το πρόγραμμα ασφαλείας και προστασίας της ελευθερίας Έχουμε ζητήσει αύξηση κατά 24,4% για το 2011 σε σχέση με το 2010. Μιλάμε λοιπόν για σημαντική αύξηση για το πρόγραμμα αυτό. Επίσης για το προϋπολογισμό του ΣΥΣΒΙΣ. Ο προϋπολογισμός του αναθεωρήθηκε προς τα κάτω στο σχέδιο προϋπολογισμού για το 2011 εξαιτίας των καθυστερήσεων βρισκόμαστε στο milestone 1 υπήρξαν αποφάσεις ε, στο Συμβούλιο ΔΕΗ και είχαμε και διαπραγματεύσεις με τους ε, αναδόχους ε, για τη συνέχεια στο ΣΥΣΒΗ. Bis είναι Περισσότερες πληροφορίες θα σας δώσουμε τον Οκτώβριο. De manière générale, euh, je suis bien disposée. Όσον αφορά τις γενικότερες ε, πληροφορίες, ε, είμαι διατεθειμένη να σας απαντήσω με περισσότερες λεπτομέρειες είτε σε διμερείς συζητήσεις ε, είτε γραπτός σε τυχόν ερωτήματά σας. Σας υπενθυμίζω ότι το σχέδιο προϋπολογισμού σέβεται το δημοσιονομικό πλαίσιο για το 2011, το πολιετές πρόγραμμα δηλαδή, Συμμορφωθήκαμε απόλυτα με αυτό κατά την προετοιμασία του σχεδίου προϋπολογισμού. Επίσης λάβαμε υπόψη την κατανάλωση, την απορρόφηση των πιστώσεων. Βεβαίως ε, αυτή τη στιγμή το πρόγραμμα τώρα ξεκινάει να λειτουργεί και δεν θέλουμε να το τραβήξουμε προς τα πίσω. Επίσης όσον αφορά ορισμένα επιπλέον καθήκοντα για την Europol, Frontex και τον Οργανισμό Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και αυτά αντικατοπτρίζονται στις αυξήσεις. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Θέλω να ευχαριστήσω τους διερμηνείς για την κατανόησή τους για αυτά τα, τον πρόσθετο χρόνο. Σημειώσαμε αυτά τα πράγματα και έγκαιρα μπορούμε να δράσουμε διότι ακόμα βρισκόμαστε στην φάση διαδικασίας κατάθεσης τροπολογιών μέχρι τις 26 Αυγούστου. Ναι, φυσικά, φυσικά. Τώρα συνεχίζει αγγλικά και ολοκλήρωσαν οι διερμηνείς. Ευχαριστούμε